Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, καλώ ήρθατε στην ε, συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Έχουμε ένα πολύ νέο μέλος εδώ πέρα, νεαρό. Ο Καλχάιντ Λούτερ έγινε πάλι πατέρας την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε παίρνει το, το πρώτο, το μεγάλο του παιδί εδώ πέρα. Καλώς Ήρθε λοιπόν και ο μικρός. Εάν κάνει φασαρία θα βγείτε και οι δύο έξω, έτσι. Λοιπόν. Έχουμε την έγκριση της ε, ημερήσιας ε, διάταξης. Ε, υπάρχει κάποια όχι. Ανακοινώσεις του Προέδρου θα τις κάνω αργότερα. Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών της 23ης Φεβρουαρίου. Εάν ε, δεν έχει κανείς αντίρρηση μέχρι το τέλος συνεδρίας συγκρίνονται και φτάνουμε στο σημείο 4, το πρώτο ουσιαστικό. Καλωσορίζω την Επίτροπο για κλιματικές δραστηριότητες, την κυρία Κόνη Χέντεγκαρτ. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Τα είχαμε πει και στην ακρόαση και τώρα πέρασαν κάποιοι μήνες έχετε ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα εδώ στην Επιτροπή μας. Εν τω μεταξύ η 31η Ιανουαρίου είχαμε τις δεσμεύσεις των μελών του ΟΗΕ. Έχουμε μετά και την επόμενη σύνοδο που θα γίνει τον Ιούνιο στην Βόνη. Βεβαίως μας ενδιαφέρει κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις οικονομικές της υποσχέσεις, αλλά βεβαίως και με την κατάσταση στην προστασία του κλίματος, με τις διάφορες δυνατότητες μείωσης των αερίων των σχετικών. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σας δίνω τον λόγο για να μας παρουσιάσετε πώς έχουν τα πράγματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να έρθω εδώ σήμερα. Πάντα με εμπνέει όχι μόνο να σας παρουσιάσω κάποια από τα πράγματα που θα ήθελα να σας πω εγώ, αλλά να ακούσω και αυτά που έχετε να μου πείτε εσείς, να υπάρχει μια αλληλοτροφοδότηση. Ελπίζω να μην μακρηγορήσω πολύ. Καταρχάς, να σας παρουσιάσω τα κύρια στοιχεία του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2010, για τα οποία είμαι υπεύθυνη εγώ. Το περιεχόμενο του προγράμματος εργασίας είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020, η οποία την χάνει και ευρεία υποστήριξη από το Κοινοβούλιο και τα κύρια στοιχεία της υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον περασμένο μήνα. Πιο συγκεκριμένα, η βασική πρωτοβουλία για μια Ευρώπη η οποία θα είναι αποτελεσματική ως προς τους πόρους της ε, ε, δίνει έμφαση σε μια ανάπτυξη η οποία θα είναι πιο πράσινη και θα έχουμε περισσότερες ε, πιο αποτελεσματικές πηγές ενέργειας και τη χαμηλή κατανάλωση άνθρακα στην καρδιά των στόχων μας. Ε, ο στόχο αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο, διότι γύρω από αυτόν τον στόχο μπορούν να ληφθούν πάρα πολλές σοβαρέ αποφάσει τα επόμενα χρόνια. Ο στόχος είναι να αποσυνδέσουμε την οικονομική ανάπτυξη με την ε, βιώσιμη χρήση ενέργειας, καθώς ταυτόχρονα θα αυξάσουμε την ανταγωνιστικότητα, θα δημιουργήσουμε νέε θέσει εργασία και θα έχουμε και ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη. Με έχετε ακούσει πολλοί από εσά να λέω στην ακρόαση και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα συνδυάσουμε έτσι, να τα σκεφτόμαστε έξι. Ότι έχουμε τρει στόχου σε έναν. Οπότε ναι μεν θα μιλάμε για την αλλαγή του κλίματο. θα προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματο, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και την ασφάλεια της, στο επίπεδο τη ενέργεια και ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασία. Όλα αυτά συνδυασμένα. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε από κοινού, δεδομένου ότι θα υπάρχει και κατάλληλη πολιτική βούληση. Και υπάρχει ένα στόχο ο οποίο πρέπει να επιτύχουμε αν θέλουμε να διατηρήσουμε το ανταγωνιστικό μα πλεονέκτημα στην ε, χαμηλή κατανάλωση άνθρακα παγκοσμίω. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ειλικρινείς και σαφείς. Υπάρχει ένας κύριος κινητήριο μοχλό από όλε τις μεγάλες οικονομίες να επενδύσουν στην ενέργεια του μέλλοντος. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Εάν δούμε τα μεγάλα προγράμματα αποκατάστασης, από την Κίνα, τις Ηνωμένε Πολιτείε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, βλέπουμε ότι η Κίνα έχει ένα μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων, περίπου της τάξης των 230 δις ευρώ. Μετά ακολουθούν οι Ηνωμένε Πολιτείε με 80 εκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις για καθαρή ενέργεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δείτε τα στοιχεία που έχουμε από τις μεγαλύτερες χώρες μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε οι επενδύσεις ανέρχονται στα 25 δις ευρώ τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό του. Έχουμε λοιπόν μεγάλο ανταγωνισμό και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τις τρέχουσες πολιτικές μας και να προχωρήσουμε τις ε, ε, καινοτομίες μας και τον ηγετικό μας ρόλο ώστε να μπορέσουμε να είμαστε η πιο φιλική προς το περιβάλλον περιοχή στην Ευρώπη, στον κόσμο. Συγγνώμη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλές πρωτοβουλίες και εγώ και οι υπηρεσίε μου ετοιμάζουμε το σχετικό έγγραφο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να έχουμε μείωση των εκπομπών κατά 30% μέχρι το 2020. Βλέπω ότι έχουμε βρει αποδοχή εδώ, με χαροποιεί αυτό. Η οικονομική κρίση έχει μειώσει τις εκπομπές και τις τιμές του άνθρακα και επομένω αυτή τη χρονική συγκυρία θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς θα μπορέσει η Ευρώπη να προάγει την ε, βιώσιμη ανάπτυξη, να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας και να μειώσει την εξάρτησή μας από την εισαγόμενη ενέργεια. Από τις αναλύσεις μας δεν προκύπτει ότι μόλις ε, θα έχουμε την ανακοίνωση θα ληφθούν και σχετικές αποφάσεις την επόμενη μέρα. Δεν αρκεί αυτό. Αν θέλουμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι από το 20% θα πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι συνέπειες, τι επιπτώσεις θα έχουμε στις διάφορες ε, τομείς και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ο στόχος της ανακοίνωσης και σκοπεύουμε η ανακοίνωση αυτή να βγει πριν από το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος στις 20 Ιουνίου και επομένως να μπορέσει να συζητηθεί και για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορώ να σας αναφέρω κάποιες ε, πολύ συγκεκριμένες ε, ε, αποφάσεις και στοιχεία. Η ανάλυση μας όμως υποδηλώνει ότι το να προχωρήσουμε στο 30% είναι εφικτό από τεχνική σκοπιάς και θα μπορέσουμε να το αναπτύξουμε και οικονομικά, θα είναι και οικονομικά βιώσιμο. Και ένα στοιχείο που θα υπάρχει στην ανακοίνωση είναι το εξή. Πριν από δύο χρόνια όταν αποφασίσαμε για το πακέτο για το κλίμα, εκτιμήθηκε ότι το κόστος ε, του να περάσουμε από το 20% να περάσουμε συγγνώμη στο 20% θα ήταν γύρω στα 70 δις ευρώ. Σήμερα γνωρίζουμε ότι λόγω της κρίσης είναι πολύ πιο εύκολο και φθηνότερο να επιτύχουμε αυτό το στόχο του 20%. με όλους τους προληπτικούς κανόνες που πρέπει να λεφθούν και όλα τα στοιχεία με μεγάλη επιφύλαξη θεωρούμε ότι είναι κατά ένα τρίτο φτηνότερο να επιτύχουμε το στόχο αυτό από ό,τι όταν το αποφασίσαμε πριν από δύο χρόνια. Και υπάρχουν φυσικά και ωφέλη για την ποιότητα του αέρα και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λεφθούν υπόψη και επομένως το 20% είναι ακόμα πιο ε, εφικτό από οικονομικής πλευράς. Και αυτό σημαίνει ότι ίσως να μην είναι τόσο ακριβό όσο φοβούνται κάποιοι το να πάμε στο 30% από την τεχνολογία που έχουμε αυτή τη στιγμή ε, και λόγω και της κρίσης από ό,τι πιστεύαμε πριν από κάποια χρόνια. Δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτό θα γίνει εν μία νυχτή και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι λόγω της κρίσης, εάν έχουμε τη δυνατότητα και είμαστε διατεθειμένοι να επενδύσουμε το ίδιο ποσό χρημάτων που θέλαμε να επενδύσουμε πριν από δύο χρόνια, θα καταφέρουμε όχι μόνο να φτάσουμε στο 20% που θέλαμε, αλλά να φτάσουμε και στο 20% και γι' αυτό ακριβώς παρουσιάζουμε και αυτό το επιχείρημα και προσπαθούμε να το διευκρινίσουμε στην ανακοίνωση της Επιτροπής. Να πω και κάποια πράγματα επιπλέον. Στις επόμενες εβδομάδες και μήνε θα παρουσιάσουμε και κάποια μέτρα τα οποία χρειάζονται για την εφαρμογή του πακέτου κλίματος και ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε συμφωνία για ένα κανονισμό για την ε, δημοπρασία ε, εκπομπών ε, και επιτρεπωμένων ωραίων. Έχουμε κανόνες για τους διάφορους τομείς που θεωρούνται ότι είναι σε κίνδυνο λόγω διαρροής άνθρακα και τη δημοσίευση του ε, βασικού στοιχείου για το 2000, των βασικών στόχων για το 2013. Κοιτώντα τώρα στο μέλλον, θέλουμε να έχουμε και μια ανακοίνωση για μια οικονομία χαμηλής ενέργειας για το 2050 και αυτή η ανακοίνωση θα αναλύσει του στόχους τους οποίους θέλουμε να επιτύχουμε καθοδόν προς το 2050 και επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε πού θα πρέπει να βρισκόμαστε μέχρι το 2030 ώστε να είναι ομαλή η πορεία μέχρι το 2050 και να μην ε, ε, αναβάλουμε συνεχώς και να είναι πολύ απότομη η ανηφόρα μέχρι τους στόχους του 2050. Επίσης να σας πω ότι θα έχουμε και μια ανακοίνωση για του χρόνου η οποία θα περιλαμβάνει μια στρατηγική και συγκεκριμένες δράσεις για να ε, μετριάσουμε τις επιπτώσεις αλλαγής του κλίματος στις διάφορες ευρωπαϊκές πολιτικές και στα χρηματοοικονομικά μέσα και κυρίως ε, θέλουμε να ελέγξουμε το σύνολο των πολιτικών από τη γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου μέχρι τη βιομηχανία, την έρευνα. Οι πρωτοβουλίες αυτές ε, μπαίνουν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παγκόσμιας δράσης, συνολικής δράσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που εστιάζει στο 2020 και την Ευρώπη του 2020. Θα πρέπει να εστιάσουμε στην ενέργεια, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη φορολόγηση αν θέλουμε να επιτύχουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους μου, θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με το θέμα της, ε, των μεταφορών και την ε, μη χρήση άνθρακα στις μεταφορές. Η Γενική Διεύθυνση Κλίμα εξετάζει την περίοδο μέχρι το 2050 και τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι εκπομπές από τον ε, τομέα των μεταφορών κατά πάσα πιθανότητα θα αυξηθούν κατά 30% στο ίδιο χρονικό διάστημα, εάν δεν κάνουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε ήδη αποφασίσει. Με βάση λοιπόν την κύρια πρωτοβουλία μιας Ευρώπης αποδοτικής ως προς τις πηγές της ενέργειας ε, και της στρατηγικής του 2020 θα πρέπει να έχουμε και τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών ώστε να έχουμε ένα τομέα μεταφορών ο οποίος θα είναι σύγχρονος, αποδοτικός και φιλικός προς το περιβάλλον. Η ανακοίνωση για το mainstreaming, την οποία σας ανακοίνωσα ήδη, δεν θα εξετάζει μόνο τις μεταφορές αλλά και τα θέματα της μη άνθρακα εν γέννη δεδομένου ότι είναι πολύ σημαντικές οι επιπτώσεις του κλίματος στις μεταφορές. Ε, θα υπάρχει ένας από τους βασικούς παράγοντες που θα εξετάσουμε εδώ, το θέμα του κλίματος και θα δούμε και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες οι οποίες θα προκύψουν και, σε συγκεκριμένα, ε, και θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένα μέτρα. Όπω σα είπα στη διάρκεια τη ακρόαση, ε, σκοπεύω από εκεί και πέρα να προχωρήσω και με ένα πακέτο κλίμακο και μεταφορών. Θα ξεκινήσουν και συζητήσει φέτο για τι επόμενε δημοσιονομικέ προοπτικέ θα ήθελα να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου προκειμένου να λάβουμε υπόψη πλήρω ε, το θέμα τη αλλαγή του κλίματο, το πώ μπορούμε να μετριάσουμε τι συνέπειε και να προσαρμοστούμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσεις του κλίματο σε όλε τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ. Τώρα, για να μιλήσω λίγο και για τον κανονισμό ο οποίος προτείνεται για τη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρωπου, τον οποίο ξέρω ότι έχετε ήδη ξεκινήσει να συζητάτε εδώ για τα μικρά φορτηγά οχήματα. Ο κανονισμός λοιπόν αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο για την αντιμετώπιση των εκπομπών στις οδικές μεταφορές και θα κάνει πολύ σημαντική συνεισφορά για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να πετύχουν τους στόχους μέχρι το 2020 και θα καλύπτει το 5% της μείωση που απαιτείται στου διάφορου τομούς που δεν καλύπτονται από το σύστημα εμπορία εκπομπών. Ε, ξέρω ότι έχουν δημιουργηθεί κάποια ερωτηματικά για το κατά πόσον το χρονοδιάγραμμα είναι εφικτό και το επίπεδο των ε, στόχων εκπομπών για το 2014 έως το 2016 και για το 2020 και είχα και την ευκαιρία να το συζητήσω και με αρκετούς από εσά την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Πράγματι, τα στοιχεία είναι πολύ φιλόδεξα. Αλλά πιστεύουμε ακράδοντα ότι είναι εφικτό δεν θα είχαμε προτείνει τα στοιχεία αυτά εάν δεν ήμασταν πεπισμένοι γι' αυτό και δεν έχουν προκύψει και από το πουθενά, έχουν προκύψει από συγκεκριμένε αναλύσεις. Ο κανονισμός αυτός θα βοηθήσει τους κατασκευαστές να ενισχύσουν την μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και να γίνουν πρωτοπόροι στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες, προχωρώντας περαιτέρω την ε, ενεργειακή απόδοση από ό,τι θα είχαν πετύχει σε άλλη περίπτωση. Είναι μια δυνατότητα μεγάλη και ελπίζω οι Ευρωπαίοι να είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα την αρπάξουν. Ελπίζουμε ότι η μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση θα εξοικονομεί στον ιδιοκτήτη κάθε νέου μικρού φορτηγού περίπου 2.000 ευρώ σε καύσιμα ετησίως. Η σταδιακή, ε, το σταδιακό phase-in του στόχου για το 2014-2016, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι έγινε γνωστό, είναι γνωστό από το 2007, ε, λαμβάνει υπόψη και τις ανάγκες της βιομηχανίας για πλήρη συμμόρφωση. Ο στόχος του 2020 είναι ε, βεβαιότητα για τους κατασκευαστές, για το μέλλον και ε, έχουμε λάβει υπόψη και τις ανησυχίες του κλάδου. Θέλουμε να επιβεβαιωθεί ο στόχος μόλις θα έχει επικαιροποιηθεί η ανάλυση το 2013. Συνοψίζοντας λοιπόν, η πρότασή μας είναι τόσο εφικτή όσο και απαραίτητη. Γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να ζητήσω από την, ε, ε, την Επιτροπή σας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολό του να λάβει υπόψη αυτό το στόχο όταν θα συζητά το σχετικό κανονισμό στους επόμενους μήνες. Επειδή είμαστε στα οχήματα, δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύριο θα εγκρίνει μία ανακοίνωση για την ε, στρατηγική για πιο αποδοτικά ως προς την ενέργεια και πιο καθαρά αυτοκίνητα οχήματα, την οποία θα παρουσιάσει ο Επίτροπος Ταγιάννη. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που τα βαρέα οχήματα είναι πλέον αυτή, τμήμα αυτή της στρατηγική, είναι κάτι νέο το οποίο ανακοινώνουμε, είναι μια πρόταση που θα στοχεύει στην κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από βαρέα οχήματα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω και λίγα πια πράγματα για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτό και να δούμε και κάποιες λεπτομέρειες, αλλά όπως ξέρετε ο Πρόεδρος Μπαρόζο μου ζήτησε να κάνω κάποια πράγματα στις αρχές ε, Μαρτίου και επειδή ε, υπάρχει και το θέμα της, ε, των ΗΠΑ, του Μεξικού, των Μαλδιβών, της Ινδία. Αύριο θα πάω στην Κίνα, αργότερα στην Αιθιοπία, στην Αφρικανική Ένωση και αργότερα στο Μάιο στο Μπαγκλαντές. Από το φόρουμ στο οποίο συμμετείχα την περασμένη Δευτέρα, διαπιστώνω ότι αυτό το οποίο εμείς προσπιζόμαστε είναι κάτι το οποίο είναι πλέον ευρέως αποδεκτό. Υπάρχει το θέμα του Κανκούν, υπάρχει ένα μεγάλο ε, βασικό σημείο το οποίο θα πρέπει να αποφασίσουμε στο Κανκούν, αλλά κατά πάσα πιθανότητα η πρόκληση θα είναι μία όσες προσπάθειες και να κάνουμε. Ο στόχος θα είναι οτιδήποτε και αν συμφωνήσουμε να γίνει ένα νομικό δεσμευτικό πλαίσιο. Όπως ξέρετε το πρόβλημα δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ. Έχουμε προσπογράψει το Κιώτο, έχουμε δεσμευθεί, ε, δίνουμε αποτελέσματα με βάση το Κιώτο. Δεν είμαστε εμείς το πρόβλημα. Αλλά από τις ενδείξεις που έχουμε από τις άλλες χώρες ε, οι άλλοι το βλέπουν διαφορετικά. Και επομένω αυτό είναι το πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε πιο πρακτικοί, να εστιάσουμε στο περιεχόμενο, να συμφωνήσουμε συμφωνήσουμε προς ένα περιεχόμενο και ίσως αργότερα να είναι πολύ πιο εύκολο να συμφωνήσουμε και προς τη νομική μορφή. Έτσι έχει το παιχνίδι αυτή τη στιγμή και θα συναντηθούμε στη Βόνη το Μάιο για να ε, δούμε και τι γίνεται σε επίπεδο διαπραγμάτευσης, αλλά την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα οι Υπουργοί για πρώτη φορά θα συναντηθούν σε ευρύτερη μορφή και θα ήθελα να ζητήσω σε όλους να εστιάσουν στην ουσία και όχι στη διαδικασία, διότι ε, αυτό χρειάζονται σε αυτή τη φάση οι διευθύνσεις διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Äh, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Μα παρουσιάσετε τι σχέσει σα τι σκέψει σα για, για τα περαιτέρω βήματα για το, την προστασία του κλίματο. Ακούσαμε μερικές φορές με τις ψηφοφορίε ένα σαφέ. ναι, μερικές φορές ακούσαμε με τον νεαρό Δανό ε, να φωνάζει για, για φαίνεται ότι είναι αρκετά τολμηρός ε, και δέχεται τις προτάσεις σας. Ακούσαμε τι έχετε στο πρόγραμμα. Δεν ακούσαμε τίποτα συγκεκριμένο για τη χρηματοδότηση. Το 2,7 δισεκατομμύρια δηλαδή της ε, κλιματικής αλλαγής. Και ο χρόνος περνάει. Τι σχέδια έχετε για να συντονίσετε αυτές τις ε, προσπάθειες της Ενέργειας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να δώσετε ένα σαφές μήνυμα και πριν από το Κανκούν προς τα αναπτυσσόμενα κράτη. Την Πέμπτη, την προηγούμενη Πέμπτη μετά το Στρασβούργο, μια ομάδα από την Επιτροπή μας, μια ομάδα βουλευτών ασχολήθηκε με τα ελαφρά λεγόμενα οχήματα, light vehicles, τα συζήτησε, είδε πόσο εφικτό είναι, πόσο υλοποιήσιμο είναι το όραμα τέτοιων ελαφρών ε, οχημάτων και ίσως θα πρέπει να το δούμε πιο συγκεκριμένα. Έχουμε μία ώρα στη θέσή μας, αρκετοί συνάδελφοι έχουν στήσει το λόγο μπορείτε να δώσετε, να κάνετε ερωτήσει, παρατηρήσεις. Ο κύριο Ζέμπαρτ, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε να μας μιλήσετε. Μιλήσατε για το mainstreaming. Ξέρετε ότι είναι ένα καυτό θέμα, η του κλίματος. Πώς λοιπόν μπορείτε να χειριστείτε το θέμα αυτό και σε σχέση με τους ε, συναδέλφους σα στην Επιτροπή, τους άλλους ε, επιτρόπους. Πώς γίνεται η συζήτηση εντάσσεται η προστασία του κλίματος σε κάθε πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει θετική ανταπόκριση στην ιδέα αυτή. Και ιδιαίτερα και στις μεταφορές Φερρυπίν, διότι η ε, πρόσφατη έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία προκάρελεσε πάρα πολλά προβλήματα και οδήγησε σε κινητοποίηση πάνω από ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα αφού δεν μπορούσαν να ε, πετάξουν τα αεροπλάνα. Άρα Πρέπει να δούμε και αυτή τη διάσταση. Μια άλλη ερώτηση έχει να κάνει με την ενέργεια και την προαγωγή της ε, βιώσιμης βεβαίω ενέργειας, των βιώσιμων μορφών ενέργειας, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει αναγκαστικά να διατηρήσουμε και τις ε, παραδοσιακέ συμβατικέ μορφέ ενέργεια, διότι οι ανανεώσιμε λεγόμενε μορφέ παρουσιάζουν διακυμάνσει και δεν μπορούμε να στηριχθούμε αποκλειστικά σε αυτέ. Υπάρχει λοιπόν κάποιο δίκτυο, ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, ε, διατήρηση, την αποθήκευση ενέργειας προκύπτει από υδροηλεκτρικά έργα κτλ. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο, κάποια πρόβλεψη αντίστοιχη για την ε, ενέργεια που προκύπτει από τον άνθρακα ή από, άλλα, από άλλες συμβατικές μορφές ενέργειας και το συνδυασμό με τις ρανόσμες. Επίσης, η κρίση σχετική με την Ελλάδα δείχνει στα δημοσιονομικά πολύ δύσκολη εικόνα, τραγική εικόνα και βλέπουμε ότι στα κράτη-μέλη δυσκολευθούν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, τις οικονομικές. Ποια είναι η κατάσταση εδώ και η λεγόμενη χρηματοδότηση fast track, η ταχεία μορφής χρηματοδότηση, μπορεί να προχωρήσει όπως περιμέναμε ή έχουν ανατραπεί όλα αυτά. Ο υπεύθυνος για τον προπολογισμό, ο συνάδελφός σας τι λέει. Ευχαριστώ πολύ Λίντα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και την Επίτροπο που ξαναήρθε στην Επιτροπή μας. Ε, δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα για τα νούμερα που μας δώσατε για την επένδυση σε πράσινη ενέργεια και καινοτομία. Δεν έπιασα το νούμερο της Κίνας. Είπατε για 200 δισεκατομμύρια και μετά 80 δισεκατομμύρια η και 25 δισεκατομμύρια μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι μετράτε για να βγάλετε αυτά τα νούμερα. Ε, προφανώς η Κίνα και λόγω του μεγέθους και του πληθυσμού είναι αναμενόμενο, αλλά το κενό μεταξύ ΙΠΑ ΕΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μεγάλο. Τι κάνετε πέρα από την ανάλυση των αριθμών. Μπορείτε να μας το αναλύσετε λίγο, να δούμε τι σε τι επενδύει η Κίνα και, και δεν επενδύει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μεγαλώσει το χάσμα ανταγωνιστικότητας. Επίσης, μιλήσατε για τη συγκριτική αξιολόγηση που θα απασχολήσει και θα ανησυχήσει τις εταιρείε για το πώς θα λειτουργήσει. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά σας τώρα γι' αυτό και πώς διαβουλεύεστε και πότε μπορούμε να περιμένουμε κάποιο αποτέλεσμα από την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Chris Davis. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, μάλλον δεν το είδατε, αλλά η αυτοκινητοβιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου είπε πως οι εκπομπές νέων αυτοκινήτων έπεσαν κατά 6% πέρσι. Πριν, ε, ενώ προηγούμαστε και του στόχου που προβλέπει η νομοθεσία. Γιατί λέμε πως κάνει λόμπι η αυτοκινητοβιομηχανία και μόλις περνάει η νομοθεσία ξεπερνάνε τις απαιτήσεις. Οπότε δεν ξέρω αν είναι τόσο φιλόδοξη η νομοθεσία για, τις, ε, για τα ελαφρά φορτηγά. Γιατί νομίζω ότι αυτό που ανισχύει τις βιομηχανίες είναι τιμή πώληση και όχι το κόστος χρήσης των αυτοκινήτων ε, που αφορά μετά τους οδηγούς. Όσον αφορά το στόχο του 30% Είστε βεβαίως επιφυλακτικοί, αν και λέτε πως οικονομικά μοιάζει εφικτός, αλλά δεν είμαστε στο Μάρτιο του 2007, έχει αλλάξει, μεταβληθεί αρνητικά η κατάσταση στο Συμβούλιο. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η διάθεση ε, του Συμβουλίου όσον αφορά τις φιλοδοξίες μείωσης του διοξιδίου του άνθρακα. Και τέλος το σύστημα εμπορίας εκπομπών που είναι μισό επιτυχημένο, Μειώνει, βοηθάει να μειώσει τις εκπομπές από τις μεγάλες εγκαταστάσεις, αλλά δεν προωθεί τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα λόγω της χαμηλής τιμής του άνθρακα. Οπότε η Κομισιόν έρευνα άλλα ρυθμιστικά μέσα για να προωθήσει αυτές τις τεχνολογίες. Η οι Ταλιμπάν έχουν μπλοκάρει το σύστημα και λένε όχι, όχι, δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο, μόνο αυτό το μηχανισμό της αγοράς. Εάν επιτρέπετε να μου δώσετε ένα παράδειγμα με την οδηγία βιομηχανικών εκπομπών, έχουμε αφενός τη γενική απέτηση πως μπορούν να πάει, είναι πιο αυστηρά τα κράτη-μέλη, αλλά σε μια άλλη οδηγία στο άρθρο 9 αναφέρεται πως ε, τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να εισαγάγουν εθνικές ε, διατάξεις για τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Ποια είναι η ερμηνεία σας, πώς μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να έχουν εθνικούς στόχους εάν θεωρούν πως έτσι θα επιτύχουν μείωση των εκπομπών. Ευχαριστώ. Σα του χάσει θα ακούσουμε ακόμα και μετά θα απαντήσει η κυρία Επίτροπος. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ την Επίτροπο που ήρθε να συζητήσει μαζί μας. Το ερώτημά μου συνδέεται με αυτό το μείον 30 των στόχων αυτών. Μας εξηγήσατε τι κάνει η Κομισιόν, αλλά Ξέρουμε πως στόχοι σημαίνουν διαφορετικά πράγματα ανάλογα με το πόσα παραθυράκια έχει η νομοθεσία. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε πως το μείον 30% στο οποίο αναφέρεστε σημαίνει όντως μείον 30%. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν παραθυράκια. Π.χ. δημιουργική λογιστική και τα λοιπά. Τι εννοείται δηλαδή ακριβώς με αυτό το μείον 30%. Ένα άλλο ερώτημα που σχετίζεται με το μείον 30% το κοινοβούλιο είπε πως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει το στόχο του 20% δεσμευτικό. Πώς το βλέπετε αυτό να συνδέεται με το στόχο του 30%. Και τέλος τα κράτη-μέλη υποσχέθηκαν 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ που να δοθούν γρήγορα, δηλαδή 2,4 δισεκατομμύρια φέτος. Βεβαίως αυτό δεν αφορά τόσο την Κομισιόν αλλά θα ήθελα να γνωρίζω τι κάνει η Κομισιόν για να διασφαλίσει πως αυτά τα χρήματα θα ξεκινήσουν να ρέουν. Γιατί βεβαίως αυτό είναι και θέμα αξιοπιστίας της πολιτικής ε, της κλιματικής της Ένωσης. Ευχαριστώ πολλές ερωτήσεις. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω με το τελευταίο τμήμα της ερώτησης. γιατί σχετίζεται και με την αρχική ερώτηση του κυρίου Λάιρεν ως προς την χρηματοδότηση. Νομίζω ότι είναι απόλυτα ζωτική σημασία για την αξιοπιστία μας να υλοποιήσουμε τα όσα υποσχεθήκαμε στην Κοπενχάγη. Και γι' αυτό άλλωστε το ονομάζουμε και fast start, γιατί πρέπει να υλοποιήσουμε και ταχύτατα, όχι δηλαδή κάποτε στο μέλλον. Και αυτό ακριβώς συζητήσαμε και αυτή την εβδομάδα. Είμαστε έτοιμοι για την συζήτηση στη Βασιλεία φέτος ε, τον Ιούνιο ή ε, στη Βόνη φέτος τον Ιούλιο ε, να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Και οι Υπουργοί των Οικονομικών είπαν ξεκάθαρα ότι τα τρία, τρεις φορές 2,4 δισεκατομμύρια που έχουμε υποσχεθεί θα τα διαθέσουμε. Είναι βέβαιο αυτό. Ένα πράγμα μόνο πρέπει να επισημάνω εδώ, που με εκκρεμές. Πόσα από τα κονδύλια αυτά θα είναι πρόσθετα ή καινούρια χρήματα, φρέσκα χρήμα. Μπορεί να σας πει κανείς ότι είναι πολύ θεωρητική αυτή η υπόθεση, πολύ θεωρητικό ερώτημα, αλλά παρόλα αυτά για τα αναπτυσσόμενα κράτη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δούμε πόσο εύκολο είναι να αντλήσουμε δημόσιο χρήμα από τους προϋπολογισμούς των κρατών σε αυτή την χρονική περίοδο, όπου θα σας απαντήσω να είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά υπάρχει το εξής ότι όσο πιο καινούριο φρέσκο χρήμα ή πρόσθετο χρήμα έχουμε, τόσο πιο ουσιαστικές συνέπειες θα έχει ή αντίστροφα. Εάν ε, φανεί ότι ναι, δόθηκαν τα 13 δισεκατομμύρια, αλλά τελικά αποδειχθεί ότι ήταν μόνο ένα ανακυκλωμένο χρήμα. Τι είδου εικόνα θα δώσουμε. Γι' αυτό και είναι απόλυτα ζωτική σημασία στο κάθε κράτος να σκεφτεί πολύ προσεκτικά τι είδους χρήματα προτείνει να προσφέρει. Και σας διαβεβαιώνω ότι αυτά τα οποία ε, έχει υποσχεθεί και προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όντω καινούριο χρήμα, φρέσκο χρήμα. Έχει ήδη εγγραφεί στον προπολογισμό του 2010 και θα συνεχίσει να εμφανίζεται και στον προπολογισμό του 2011. Είναι απαραίτητο εμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε το δικό μα μερίδιο τη δουλειά και να φανεί κιόλα ότι και οι ε, αναπτυσσόμενε χώρε κάνουν ε, επιτελούνται επισχυμένα. Επίσης έγινε μια ερώτηση για το mainstreaming. Θα ήθελα να πω τα εξής. Η Επιτροπή αυτή καθεύτη θεωρεί ότι δεν είναι μόνο ο Επίτροπος του Περιβάλλοντος ή ο Επίτροπος Αρμόδιος για τα θέματα του κλίματος ε, αρμόδιος να συζητήσει και να αποφασίσει για το 2020, αλλά ολόκληρη η Επιτροπή στο σύνολό τη. Και την προηγούμενη εβδομάδα ακριβώς μπορέσαμε να συζητήσουμε και πρέπει να σας πω ότι έχουμε συζητήσει μια ομάδα για το κλίμα, τη οποία θα ηγηθώ εγώ, και που θα αποτελεί το φυσικό χώρο στον οποίο θα συζητούνται τα προβλήματα όποτε υπάρχουν. Και αυτό όχι μόνο κάθε φορά που εμφανίζεται νέο νομοθέτημα προς συζήτηση, αλλά οποτεδήποτε βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Η κυρία Μαγκάβν ρώτησε για τα στοιχεία αυτά, αν μπορούμε να δώσουμε μια μεγαλύτερη κατανομή. Ναι, το όντι, αλλά εάν δούμε τις αναλογίες και άλλωστε τα κινέζικα στοιχεία είναι μάλλον προσπάθειες, ε, τα αμερικανικά σχετίζονται περισσότερο με την ενέργεια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς πρέπει να δείξουμε ότι πιστεύουμε πως και ο υπόλοιπος κόσμος και οι επιλεγόμενοι ανταγωνιστές μας θα κάνουν και πρέπει να καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες. Διαφορετικά θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Και αυτό μας το δείχνουν ήδη τα στοιχεία που έχουμε μπροστά μας. Αποτελούν μια σαφέστατη ένδειξη του τι μας περιμένει στο μέλλον. Εξού και το χρονοδιάγραμμα που στόχο έχει να ε, έχουμε συγκεκριμένη δράση μέχρι το τέλος του χρόνου, να έχουμε συγκεκριμένη κόμμα να πάμε πιο πέρα, έχουμε διαβουλές εντατικέ, σας διαβεβαιώνω και πρέπει να σας πω ότι ίσως γίνεται και αντίστροφα, δηλαδή ο κόσμος μας πιέζει και μας ζητάει συνέχεια ε, η προσφορά ιδεών και συμβουλές κτλ. Για το benchmarking για τα ορόσημα, θα ήθελα να σας πω το εξή ότι αγωνιστήκαμε αρκετοί από εμά να φτάσουμε μέχρι το 100% στους πληστηριασμούς. Τώρα είδαμε με τα ορόσημα ότι έχουμε να κάνουμε μάλλον με έναν εφικτό πολιτικό συμβασμό. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε αυτό το πράγμα μόνο σαν μία ε, δουλειά που γίνεται ανατομέα και δεν έχει καμία ουσία και είναι κατακαιρματισμένη κτλ. Όχι, έχει πολύ μεγάλη σημασία και είναι πολύ περίπλοκη δουλειά. Ο Κρυς Ντέιβις μίλησε για τα αυτοκίνητα και την βιομηχανία. Ναι, συμφωνώ. Πολλά είναι τα προβλήματα και οι δυσκολίες, αρχικά τουλάχιστον, αλλά πολλές φορές βλέπουμε στην πορεία ότι ήταν ε, στην πράξη πολύ λιγότερα τα προβλήματα και οι δυσκολίες από ό,τι περιμέναμε και τελικά και με μικρότερο κόστος υλοποιούνται αυτά που θέλουμε. Ίσως λοιπόν είναι πιο εύκολο να πείσουμε την βιομηχανία εάν είναι σαφές ότι θα προχωρήσουμε και έτσι θα βρει τους τρόπους και για την καινοτομία χωρίς τις μεγάλες δυσκολίες. Ακούστηκε από κάποιον από του ομιλητέ ότι δεν είμαστε πια στο Μάρτιο του 2007. Ναι, όντω έχουν αλλάξει συνθήκε. Αλλά δεν είμαστε πια στο Μάρτιο του 2007 και ω προ τι τάσει και τη συμπεριφορά των ανταγωνιστών μα. Δεν κινούνται προ διαφορετικέ ε, κατευθύνσει ο καθένα. Έχουν αλλάξει και αυτοί οι παράμετρο. Και άρα πρέπει να δούμε θετικά ε, τη νέα περίοδο που διανύουμε. Επίσης και με το ETS αλλά και με την πρόταση για την φορολογία στην ενέργεια που θα κατευθεί αργότερα βλέπω αρκετές λύσεις. Υπάρχουν και άλλες βέβαια συμπληρωματικές του ETS. Δεν αρκεί δηλαδή μόνο το ETS. Επίσης αναφερθήκατε στις ε, προδιαγραφές αποδοστικότητας των εκπομπών. Το ίδιο είχε υποθεί σε μια προηγούμενη συνεδρία για την αποδοτικότητα των φυτών, ε, εκπομπές φυτών. Όλα αυτά θα τα δούμε. Των εργοστασίων, συγγνώμη. Ε, όλα αυτά θα τα δούμε λοιπόν, θα έχουν πιο συγκεκριμένα ε, δεδομένα. Και προσπαθούμε επίσης να κλείσουμε και τα διάφορα κενά που υπάρχουν, τα παραθυράκια, ε, με την προσοχή μας ανακοίνωση. Μιλήσατε για το UCF, ναι μπορεί να υπάρχουν 20-30% αλλά θα πρέπει μέσα από αυτό να βρούμε και εμείς μια πολιτική ως ένωση και να διατυπώσουμε συγκεκριμένα τις ιδέες μας. Είναι κάτι το οποίο δεν είδαμε στην Κοπεχάγη, δεν υπήρχε δηλαδή μια ενωμένη, σαφή και στεναρή θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Κώστα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε. Μας δώσατε ήδη αρκετές ενδείξεις με την ομιλία σας. Βλέπω ότι έχετε αγώνα σε δύο μέτωπα να αναπτύξετε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στη εθνική σκηνή. Μετά το Κοπεχάγη και μας τα είπατε άλλωστε και στην ε, ακρόαση 14 Απριλίου πώς μπορεί να υπάρχει ακόμη η Ευρώπη μετά το Κοπενχάγη, τι είδους κατευθύνσεις και προσανατολισμούς διαβλέπετε στα προσεχή βήματα που θα μας ε, πάνε μέχρι το Κανκούν. Μίλησατε για την στάση των ΗΠΑ, για την Κίνα, η οποία φαίνεται να λαμβάνει τόντι αποφάσεις με μεμονωμένες αποφάσεις, αλλά πώς μπορούμε να υπολογίσουμε την αποτελεσματικότητα ως προς τον άνθρακα. Βλέπουμε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος της Ινδίας μια σαφή βούληση, εκδήλωση μάλλον σαφούς βουλήσεως για πρόοδο, αλλά είναι μόνο εκδήλωση ή υπάρχει αυτή η βούληση το όντι. Και επίσης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσπαθήσουμε να πείσουμε, αλλά το είπατε κι εσείς, ε, κατά τρόπον ώστε κατά προτεραιότητα να υποστηρίζονται οι επενδύσεις ε, που τίνουν προς την ε, καινοτομία, δηλαδή η περιβαλλοντική πολιτική να συνδυαστεί με την πολιτική για το κλίμα και αντίστοιχα με τις επενδύσεις. Ερωτώ λοιπόν πώς μπορούμε εμείς ως πολιτικοί να σας υποστηρίξουμε, τι ζητάτε από εμάς δηλαδή, Και όταν μας λέτε ότι είναι χάρη στην κρίση δυνατόν να μειώσουμε κατά 30% τις εκπομπές του άνθρακα, θα σα απαντήσω ότι πολύ καλά, αλλά εμεί δεν υπάρχει κανεί που να θέλει να μείνουμε στην κρίση. Θέλουμε το ταχύτερο δυνατό να διαφύγουμε από την κρίση. Ως εκ τούτου λοιπόν το 38% της μείωσης θα το διατηρήσουμε και αν είναι πώς, χωρίς δεδομένο, δεδομένη την κρίση. Αυτά θα θέλαμε κάποιες απαντήσεις λοιπόν για να δούμε πιο ξεκαθαρά την κατάσταση. Γιώργενσον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επίτροπο για την παρουσίασή της. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη σχετίζεται με την ανάλυση που μόλις κάνατε για το κατά πόσον είναι εφικτό να πάμε από το 20% στο 30% στόχο για τη μείωση των εκπομπών. Από ό,τι βλέπω εδώ, οι διάφορες πηγές ανάλυσης έχουν προβλήματα. Πρώτον, όπως είπατε, ε, πολλές φορές ε, το κόστος ε, είναι υπερβολικό. Ακόμα και αν έτσι, και αν δεν είναι έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις τα ωφέλη δεν εκτιμούνται καταλήλως. Πώς μπορούμε να μετρήσουμε τα ωφέλη. Είναι εύκολο να μετρήσουμε το κόστος μιας δράσης, είτε και το κόστος του να μην κάνει κανείς τίποτα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε το πρώτο αποτέλεσμα, πώς θα το υπολογίσετε αυτό και επίσης πώς μπορείτε να υπολογίσετε το αποτέλεσμα του να πιέσουμε ένα συγκεκριμένο κλάδο να καινοτομήσει. Ορισμένε φορέ, όταν κάνουμε νομοθεσία, αυτό υποχρεώνει κάποιου κλάδου τη βιομηχανία να κάνουν κάποιε αλλαγέ και καινοτομίε που δεν θα είχαν κάνει ποτέ αν δεν του είχαμε υποχρεώσει. Αυτά τα ωφέλη είναι πολύ δύσκολο να τα υπολογίσουμε, γιατί δεν ξέρουμε πού θα γίνουν αυτέ οι βελτιώσει. Ξέρουμε απλώ ότι πρέπει να πιέσουμε για βελτιώσει. Φοβάμαι λοιπόν ότι μπορεί να έχετε μία ανάλυση η οποία ε, προφανώς θα αποδείξει όπως ε, λέτε εσείς ότι μπορεί να είναι εφικτό να το κάνουμε αλλά δεν αποδεικνύει ποιος είναι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο θέλουμε να το κάνουμε για να είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί για το μέλλον. Θα έχουμε την πρώτη ε, επίπτωση, θα πιέσουμε τον κλάδο μας να καινοτομήσει, τους, τη βιομηχανία μας να καινοτομήσει αλλά το θέμα είναι πώς μπορούμε να έχουμε απτά στοιχεία από τις αναλύσεις. Η δεύτερη ερώτησή μου έχει σχέση με αυτό που ρώτησε και ο Chris Ντέιβις με το σύστημα εμπορία εκπομπών, διότι νομίζω δεν απαντήσατε διεξοδικά. Ο Chris Ντέιβις ρώτησε τι εναλλακτικά μέτρα λαμβάνονται υπόψη. Θα ήθελα να το ξέρω κι εγώ αυτό. Μήπως έχετε σκεφτεί την εισαγωγή κάποιας ελάχιστης τιμής. Αυτό συζητήθηκε και πριν από την Κοπεχάγη, αλλά μετά φάνηκε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα βρισκόμαστε σε μια διαφορετική κατάσταση μάλλον. Γιατί να μην είναι λοιπόν αυτό ένα από τα βασικά επιχειρήματα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουμε μια ελάχιστη τιμή για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ωραία. Ο συνάδελφος δεν ήταν εδώ. Πέτρ Λίζε λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Επίτροπε, κάποια σημεία στα οποία θα ήθελα να σας παρακαλέσω να διευκρινίσετε την απάντηση που δώσετε στον κύριο Ζέμπερ. Πρώτα απ' όλα για το θέμα των ανανεώσιμων πηγών όσον αφορά την ρύθμιση γιατί λέτε πως ε, Πράγματι πρέπει να απομακρυνθούμε από τις ε, παραδοσιακές πηγές, αλλά οι ανανεώσιμες δεν είναι αξιόπιστες. Η υδροηλεκτρική είναι βεβαίως και βεβαίω αυτό είναι θέμα άλλου συναδέλφου. Δεύτερον, για τις αεροπορικές συγκοινωνίες. Ξέρετε, ε, και ήσασταν πρόεδρος του COP15 πρώτης ε, Κοπενχάγης, οπότε θα ήθελα να σας παρακαλέσω να το προσέξετε αυτό το θέμα και στις διμερείς ε, συγκοινωνίες. Στις ΕΠΑ ακούγονται ανησυχητικές ειδήσει, αλλά τελικά μάλλον θα υπάρξει κάποια σχετική νομοθεσία. Καλύπτονται από ό,τι φαίνεται οι αεροπορικές συγκοινωνίες, αλλά υπάρχει βεβαίως και η απειλή της προσφυγής στα δικαστήρια. Οπότε καλό θα είναι με τους Αμερικανούς διμερώς να βρούμε μια λύση τέλος να υπογραμμίσω αυτό το οποίο είπε ο Νταν Γέργενσεν. Δεν είναι πολύ πολύπλοκο. Υπάρχουν χιλιάδες πλεονεκτήματα που δεν μπορούν να υπολογιστούν, αλλά τα πλεονεκτήματα που μπορούμε να υπολογίσουμε πρέπει να μπουν στην ανάλυση. Και νομίζω πως είναι σχετικά απλό να δούμε την αύξηση θέσεων εργασίας, να μπουν και αυτά στην ανάλυση, όχι μόνο το κόστος, αλλά και το όφελος μπορεί να υπολογιστεί. Ευχαριστώ. Με την νομοθεσία τον είπα δυστυχώ τα νέα δεν είναι καλά. Αναβλήθηκε το νομοσχέδιο, δεν θα γίνει ψηφοφορία σήμερα. Ε, εξακολουθεί λοιπόν η κατάσταση να παραμένει ανοιχτή το τι θα γίνει. Αν Βάις Ναι και εγώ ήθελα να το αναφέρω ακούγοντας ε, την Επίτροπο, εντάξει, εμείς ικανοποιούμαστε γιατί στην Ευρώπη είμαστε φιλόδοξοι και έχουμε στόχους, αλλά πρέπει να δούμε, εντάξει, τι γίνεται με το 30% κτλ. Αλλά οι στόχοι αυτοί, 20-20-20 και πιθανώς ε, και ακόμη παραπέρα, είναι δικαιολογημένοι. Αλλά αν ρίξουμε μια ματιά στη ΣΥΠΑ, ανησυχούμε πάρα πολύ εγώ ήμουν υπερήφανη όταν άκουσα τον Ομπάμα στην πρώτη του ομιλία στο Κογκρέσο που είπε «Θέλω εγώ να φτάσουμε την Ευρώπη στο κλίμα». γιατί είχα εγώ συνεργαστεί στην νομοθεσία τη σχετική και λέει, είπε πώς θα το κάνει θέμα. Βεβαίως ξεκίνησε με την υγεία, αλλά μπορούμε να ελπίζουμε πώς θα προχωρήσει και εκεί. Οπότε το ερώτημά μου είναι μετά την Κομεχάγη τι γίνεται με τις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Ε, δεν ξέρω αν έχετε επαφές σε υψηλό επίπεδο στην Αμερική γιατί αν συζητάμε εμεί εδώ πέρα ένα 30% το νόημα είναι τι κάνουν και οι άλλοι. Και ειδικά είπα στο πλαίσιο αυτό. Κατόπιν ε, να σας ευχαριστήσω και για την επικοδομητική συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαι αρμόδια του κόμματός μου. Γνωρίζω τη συζήτηση για τα γιοταχή και γνωρίζω πως οι απαιτήσει ε, της αυτοκινητομηχανίας πρέπει να εξεταστούν και να, να τις δούμε για να δούμε τι συμβιβασμός θα προκύψει αλλά παρόλα αυτά θέλω να πω πως ε, με τα φορτηγά είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αργούν, οι κύκλοι είναι πιο αργοί, ο αριθμός των οχημάτων είναι πιο μικρός, οπότε θα ήθελα να δώσω το μήνυμα. Η νομοθεσία μας να αποτελέσει κίνητρο και να μην έχει τόσο μεγάλο χαρακτήρα τιμωρητικό. Βεβαίως να υπάρχει και τιμωρία εντάξει, αλλά να έχουν την ευκαιρία να επιτύχουν οι εταιρείε ε, αυτούς τους στόχους. Γιατί τι θα γίνει στο τέλος, θα πληρώσουν τα πρόστιμα, δεν θα υπάρξει καινοτομία. Γιατί ε, αν μπορείτε να δείτε το τι γίνεται με τα γιοταχή για την πρόταση που θα έρθει, για να το εξετάσουμε ως εξής το ερώτημα είναι όντως κίνητρο για καινοτομία. Και αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Θα μπει τώρα η βάση με τα γιόταχη για να φτάσουμε μετά και στα φορτηγά. Π.χ. όταν λέτε ότι δεν μπορεί να υπολογιστεί η καινοτομία ε, ή ότι έχει μόνο ένα 10% επίδραση στον κύκλο δοκιμών πως υπάρχουν γραφειοκρατικά επί εμπόδια, αποστέλει 12 μήνες η Κομισιόν για να γνωρίσει αυτές τις καινοτομίες. Δηλαδή, κίνητρο δεν υπάρχει. Γι' αυτό σας ευχαριστώ που θέλετε να επανεξετάσετε το όλο θέμα και κάτι ακόμα για τις ε, υπερπιστώσεις. Πράγματι πρέπει να υπάρχουν ε, κίνητρα και για ελαφρά φορτηγά να έρθουν στην ε, αγορά και θα πρέπει αυτές οι super credits να επεκταθούν και πέρα από το τωρινό χρονικό πλαίσιο. Γενικά λοιπόν το μήνυμα πρέπει να είναι κίνητρα για καινοτομίες και λιγότερο τιμωρία. Για τους στόχους μετά το βλέπουμε. Όταν έρθει και η πρότασή σας, τόσο ή άλλως θα έρθει στην Επιτροπή. Ευχαριστώ τελειώνει εδώ ο κατάλογος των ομιλητών. Θα δώσουμε μετά τον λόγο στον συνάδελφο, τον κύριο Γκερμπράντι. Ευχαριστώ. Θα να ευχαριστήσω την ε, Επίτροπο για τις αφήσεις τώρα απαντήσεις της. Έχω δύο ερωτήσεις. Καταρχάς, είπατε ότι θα είναι λιγότερο ακριβό το να επιτύχουμε τους στόχους για το κλίμα το 1 τρίτο δηλαδή από ό,τι μπορούσαμε να υπολογίσουμε πριν από μερικά χρόνια. Αλλά αυτό δεν οφείλεται στο ότι η παραγωγή είναι και πολύ χαμηλότερη από ό,τι μπορούσαμε να περιμένουμε. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να επενδύσουμε και πάλι στην καινοτομία και ότι τώρα που αναπτύσσεται και πάλι η οικονομία θα έπρεπε να ξεπεράσουμε τα αρχικά μας, ε, τις αρχικές μας προβλέψεις. Ε, για να προχωρήσουμε περαιτέρω. Επίσης, ε, το τσιμέντο, με τσιμέντο βιομηχανία, από ό,τι γνωρίζουμε, ασκεί πιέσει πολλές με τα λόμπι τη και σε άλλα κράτη-μέλη βέβαια, όχι μόνο στην Αγγλία, ώστε να μην ε, μπει στα ορόσημα στο benchmarking ολόκληρη διαδικασία ε, παραγωγής του τσιμέντου, αλλά ένα προϊόν που ονομάζεται clinker, που είναι κάπου στα μισά της αλυσίδας παραγωγής του τσιμέντου, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο να τηρήσει και τις προδιαγραφές στόχους. Και ίσως η Επιτροπή υποκύπτει για να είναι και πιο ρεαλιστική η στάση της στις ε, προτιμήσεις ε, ορισμένων κρατών μελών και της, ε, της και, ότι, και φαίνεται ότι κινείται προς μία λύση ενός προϊόντος που θα ονομάζεται Clinker Plus. Μια νομοθεσία που ονομάζεται Clinker Plus. Υπάρχει λοιπόν αυτό. Ή μπορείτε να αντισταθείτε στις πιέσεις της μετροφημηχανίας και ορισμένων κρατών μελών που είναι μάλιστα και μεγάλα και μεγάλη επιρροή και θα μπορέσετε τελικά να περιλάβετε στους στόχου αυτούς ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγή του τσιμέντου. Ευχαριστώ η Μαρίτα Ουλσκοκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Με ε, εξέπληξε θελτικά τα, με εξέπληξαν θετικά τόσα όσα άκουσα σήμερα από εσάς. Πριν από ένα μήνα περίπου που είχαμε την ευκαιρία να σας δούμε στο Στρασβούργο, κύριε Χιλτουργκόρτ, ήταν ε, πολύ διαφορετικό το επίπεδο των φιλοδοξιών σας. Είχαμε πει ότι είναι καλό να υπάρχουν φιλοδοξίες ε, υψηλές πριν από το Κανκούν. Καλό να έχουμε το στόχο του 30% για τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Και, και στις δύο περιπτώσεις έδειξε η Επίτροπος ε, διστακτικότητα, επιφυλακτικότητα. Έλεγε ότι ναι, ίσως να μην είναι τελικά και πολύ κακό να έχουμε πιο μέτριο μέτριοπαθείς προσδοκίες σε σχέση με το Κανκούν. Δηλαδή απογοητευτήκαμε, ορισμένοι από εμάς απογοητευτήκαμε πολύ ειδικά στην ομάδα μου. Και τώρα βλέπω κάτι το τελείως διαφορετικό. Βλέπω πολύ πιο θετική αποφασιστική στάση και αυτά που μας λέει σήμερα η κυρία Χέντεγορτ είναι ότι είναι καλές οι προσδοκίες μας, είναι καλό να έχουμε υψηλές φιλοδοξίες γιατί αυτό συνεπάγεται και περισσότερη δυναμικότητα, ε, σημαίνει και όθηση για νέες επενδύσεις και καινοτομία και αναζήτηση νέων αγορών από πλευρά της βιομηχανίας. Και μας λέτε κιόλας ότι τα χρήματα από ούτως ή άλλως είναι λιγότερα από ό,τι αρχικά είχαν αποφασιστεί, θα μπορέσετε να επιτύχετε το στόχο του 30%. Ε, μπράβο λοιπόν. Τι να πω. Αυτό λέγαμε εμείς από την αρχή όμως. Με τις ερωτήσεις που σας υποβάλαμε στην ακρόαση εκείνη, αυτό λέγαμε. Ε, τώρα λοιπόν μας ενθαρρύνετε με την θετική σας στάση. Καλή αρχή, ελπίζω να μην έρχεται πολύ αργά, τουλάχιστον για το Κανκούν. Αυτές οι στόχοι για τη μείωση των εκπομπών λοιπά εξαρτούνται πάντα από τι σαφές αποφάσεις. Από τις σαφείς αποφάσεις χρειαζόμαστε πέραν αυτών και σαφείς τοποθετήσεις, ξεκάθαρες δηλώσεις ώστε να αποδεχθούμε αξιόπιστοι και του Κανκούν. και νομίζω και για τις φιλοδοξίες και για τις προσδοκίες που ορίζουμε για μας τους ίδιους καταρχάς και ως στόχους για το περιβάλλον νομίζω πρέπει να είμαστε στο δυνατόν πιο σαφείς με σαφείς δηλώσεις για να παρασύρουμε και τα άλλα τα αναπτυσσόμενα κράτη του κόσμου για να δείξουμε ότι δεν τα εγκαταλείπουμε, δεν θα επαναλάβουμε τα λάθη του Κιώτο και ότι δείχνουμε αλληλεγγύη και προς τους πιο αδύναμους. Αυτή ήταν η συζήτηση από το Κιώτο μέχρι το Ιωπεχάγη. Για μένα αυτό είναι το νόημα όλου του διαλόγου που έγινε. Και βεβαίω, αν κάπου φρονεί η Επίτροπο ότι χρειάζεται τη βοήθειά μου, πολύ ευχαρίστω να τη την προσφέρω. Βλέπετε λοιπόν από τη μια άκρη στην ε, άλλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ακούγονται εγκόμια για τις αφήσεις απαντήσεις και για τα φιλόδοξά σας ε, προγράμματα. Ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσω πολύ σύντομα στην κυρία Γκροστέτ που με ρώτησε αν είναι απλώς ε, προφύλαξη αυτό που κάνει η Ινδία και η Κίνα κτλ. Δεν νομίζω. Αφενός έχουμε τη διαπραγματεύσεις και ξέρουμε ότι τα πράγματα προχωρούν πολύ αργά εκεί, θα επανέλθω σε αυτό σε λίγο, αλλά δεν θα πρέπει να το συγχαίουμε αυτό με όλα όσα συμβαίνουν στην κάθε χώρα. Και εκεί πραγματικά φρονώ ότι κινούνται, επενδύουν σε πιο ε, καθαρές λύσεις για διάφορους λόγους, όχι λόγω των διεθνών διαπραγματεύσεων, όχι λόγω του τι πιστεύουμε εμείς, αλλά γιατί γνωρίζουν ότι για την οικονομία τους και για όλα τα θέματα κοινωνικής πρόνοιας τα δικά τους είναι πολύ ε, πιο επιτακτικό να βρουν τρόπους να έχουν πιο καθαρή ενέργεια. Πραγματικά πιστεύω ότι είναι ειλικρινής λοιπόν. Είπατε ότι ίσως εάν μπορέσουμε να βγούμε πιο γρήγορα από την οικονομική κρίση δεν θα είναι εύκολο να αξιολογήσουμε το κόστος του να κάνουμε το τάδε ή το δίνα, διότι αυτή τη στιγμή είναι κειμενόμενο το κόστος και αυτό το γνωρίζουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σίγουρα είναι να χρησιμοποιήσουμε την ανάλυση για να λάβουμε τα στοιχεία, να δούμε λίγο κάποιες μελλοντικές προοπτικές και να έχουμε και κάποιες αναλογίες. Συμφωνώ μαζί σας ότι οποιοδήποτε στοιχείο μπορούμε να έχουμε σε αυτούς τους αβέβαιους καιρούς δεν θα πρέπει να γραφεί σε, πέτρα. Είναι στόχοι οι οποίοι μπορούν να μεταβληθούν. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας είναι να αναγνωρίσουμε είναι ότι δεν έχουμε ένα παιχνίδι που ξεκινάει από το μηδέν όπως και να κινηθεί η Ευρώπη, εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι οι ανταγωνιστές μας κινούνται, επενδύουν, κάνουν διαφορετικά πράγματα σήμερα από ό,τι έκαναν πριν από 5, 10, 15 χρόνια και αυτό νομίζω θα πρέπει να το έχουμε κατά νου εάν θέλουμε να είμαστε ε, ηγέτες, πρωτοπόροι σε αυτό το τομέα και να διατηρήσουμε τη θέση μα. Με ρωτήσατε επίση πώ μπορούμε να υπολογίσουμε το αποτέλεσμα του να προχωρήσει να αλλάξει η βιομηχανία. Έχετε δίκιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδείξουμε τι θα είναι το αποτέλεσμα κάποιου πράγματος που θα κάνουμε στο μέλλον. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Από την άλλη βέβαια, θεωρώ ότι παρά το γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολη αυτή η ανάλυση και δεν μπορεί να γίνει εύκολα, εκείνο που είναι σίγουρο σχεδόν είναι ότι αν εμείς μείνουμε στάσιμοι, αν και οι κύριοι ανταγωνιστέ μα δεν μείνουν στάσιμοι αλλά κινηθούν πολύ γρήγορα, το λογικό είναι ότι ελοχεύει ο κίνδυνο να χάσουμε θέσει εργασία, εισοδήματα και δυνατότητες εξαγωγών και μάλιστα σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Ε, Ρωτήσετε αν έχουμε αναλλακτικά μέτρα και αναφερθήκατε και σε αυτή ε, την ελάχιστη τιμή, το κατόφλι για τις τιμές του διοξιδίου του άνθρακα. Γνωρίζω ότι οι συζητήσεις ε, γίνονται και εδώ στο Κοινοβούλιο και το έχετε πει και στο παρελθόν. Αυτό που θεωρώ βέβαιο είναι ότι εφόσον ε, εισαχθεί κατόφλι θα υπάρξει και αίτηση για ανώτατο όριο. Τα αποτελέσματα των τιμών του άνθρακα δεν ε, είναι το, τα ίδια με τις τιμές του πετρελαίου. Δεν είναι τόσο μεγάλες οι διακοιμάνσεις δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι απαραίτητο να έχουμε αυτό το κατόφλι γιατί θα αρχίσουν να κινούνται κατόπιν οι τιμέ του άνθρακα προ αυτή την κατεύθυνση. Δεν είμαι τόσο βέβαιη ότι θα έχουμε τα ίδια πράγματα που έχουμε και με το πετρέλαιο. Η αγορά του άνθρακα έχει αντιδράσει όπως θα περιμέναμε μια κάποια αγορά να αντιδράσει. Αφού υπάρχει μικρότερη ζήτηση για εκπομπές και δικαιώματα εκπομπών, τότε προφανώς πέφτει και η τιμή. Ε, δεν είναι τίποτα ε, το περίεργο. Είμαι βέβαιη ότι μόλις ξεφύγουμε από την κρίση θα δούμε, όπως βλέπουμε και τώρα, ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά να ανεβαίνουν οι τιμές. Τώρα, το πότε θα είναι η πρώτη ομαλή χρονιά, ελπίζουμε να είναι το 2010, αν όχι το 2011, δηλαδή να είναι η χρονιά που θα αρχίσουν οι αγορές να επιλύουν τα προβλήματά τους και θα μπορούν ε, από μόνες τους να προχωρήσουν. Ο Πίτερ Λίζα με ρώτησε κάποια πράγματα για τις μεταφορές. Ναι, γίνονται συζητήσεις σε πολύ ψηλό επίπεδο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχετε δίκιο, υπάρχει πρόβλημα, το συζητάμε. Γίνεται και μια συνεδρίαση εδώ στις 5 που θα συζητήσει μεταξύ άλλων και αυτό. Είναι ένα από τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε και συζητώνται και σε πολύ ψηλό επίπεδο στη Washington αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να δούμε και τα κοινά ωφέλη και αυτό θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε στην ανακοίνωση και επίσης να δούμε τι θα σημαίνει εάν έχουμε μεγαλύτερη και αποδοτικότερη ενέργεια και πρέπει να έχουμε μεγαλύτερες εισαγωγές, τι θα σημαίνει αυτό για τη δική μας ενεργειακή ασφάλεια και τι εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων ευρώ θα έχουμε. Επίσης, αναφερθήκατε και στην κατάσταση στις ΗΠΑ και έχετε δίκιο, το είπε και ο πρόεδρος αυτό. Είναι συναρπαστικά αυτά που συμβαίνουν εκεί αυτή τη στιγμή θα μπορούσε ίσως να μας θλίβει το γεγονός ότι εμείς ακόμα προσπαθούμε να προχωρήσουμε. Πρέπει να πούμε όμως ότι υπάρχει ελπίδα ακόμα. Είδα τι είπε η Λίντσι Γράχαμ και τι ε, είπαν ε, ότι είπε το Σάββατο και τι είπαν ότι είπε την Κυριακή. Δεν είχε χάσει την ελπίδα του. Το Σάββατο είχε φύγει από την ομάδα των τριών που συνέτασε την ε, νομοθεσία που παρουσιάστηκε σήμερα και μετά ήταν πάρα πολύ σαφές και γιατί το έκανε. Δεν ήθελε η ενέργεια να είναι προτεραιότητα ε, σε, ε, εις βάρος της νομοθεσίας για τη μετανάστευση. Αυτά είναι εσωτερικά θέματα βέβαια. Ε, εμείς από πλευρά Ευρωπαϊκής θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι προχωρά ακόμα το θέμα και προσπαθεί να έχει νομοθεσία για την ενέργεια στη Γερουσία. Οι Ηνωμένε Πολιτείες ή μάλλον ο κόσμος δεν έχει την πολυτέλεια να αποτύχουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Αλλά θα πρέπει να δούμε και τι μπορούν να κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε στο θέμα αυτό. Επίσης, ρωτήσατε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε τι διεθνεί διαπραγματεύσεις για το κλίμα και νομίζω ότι αυτό συνάδει και με αυτό που ακούσαμε στο τέλο από την Μαρίτα Ούλσκο και θα επανέλθω και σε αυτό. Δεν μπορώ να σας πω πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. Έλαβα πολλά στοιχεία από εσά και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Τα αναλύουμε τα στοιχεία. Θα συναντήσω και τις υπηρεσίες μου αύριο και θα το συζητήσουμε. Αλλά Ω υπουργό ε, θυμάμαι όταν είχαμε τι συζητήσει Ευρωπαϊκή Ένωση 5 ε, και 6 μεταξύ Επιτρόπου Δήμα και Φερχόγγεν και άκουσα όλα τα επιχειρήματα ότι οι οικονομίε θα καταρρεύσουν αν δεν κάνουμε τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Εξ όσου γνωρίζω ακόμα εκεί είναι τα πράγματα, δεν έχουν καταρρεύσει οικονομίες. Και νομίζω ότι το χειρότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για τους ε, για όσους ασχολούνται με τον άνθρακα είναι να κάνουμε αυτό που μας ζητούν να κάνουμε. Γιατί τότε δεν θα είναι αρκετά φιλόδοξοι και τελικά θα χαθούν οι αγορές. Και αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό. Με ρωτήσατε επίσης, ο κύριος Γκεμπράντη ρώτησε αν θεωρώ ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει σχετική νομοθεσία για το θέμα. Συμφωνώ 100%. Το 20% και το 30% και συζήτηση για το επίπεδο φιλοδοξίας που είχαμε προβλέψει το 2007 και 2008. Τι θα πρέπει να κάνουμε για τις ευρωπαϊκές καινοτομίες. Αυτή τη στιγμή λόγω της κρίσης μπορούμε να φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο μείωσης χωρί να υπάρχει η ίδια φιλοδοξία για καινοτομία. Και αυτό είναι ο μεγάλο κίνδυνο για την Ευρώπη και γι' αυτό ακριβώ την κρίση, λέω ότι δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι πάμε στο 30% λες και είναι πανεύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο. Θα πρέπει να σκεφτούμε όμως ότι θα μπορούσε να είναι και μια εναλλακτική λύση ακριβώς επειδή έχουμε δυνατότητες να καινοτομήσουμε. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Ένα ακόμα benchmark δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά και εσείς είπατε ότι είναι φήμες αυτά τα πράγματα. Θέλω να έχω κάποιους σχετικά εύκολα διαχειρίσιμους κανόνες, ε, παρά το γεγονός ότι το αποτέλεσμα μπορεί να είναι και απίθανο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, δεν θα πω περισσότερα πράγματα, έχουμε χρόνο γι' αυτό. Τελευταία παρατήρηση από τη Μαρίτα Ούλσκα. Σα ευχαριστώ πολύ για τα καλά σα λόγια. Δεν είμαι βέβαιη ότι κατάλαβα πώ μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου. Μου φάνηκε ότι είπα το ίδιο πράγμα. Η εξαίρεση είναι ότι όταν έγινε η ανακοίνωσή μας το Μάρτιο του 2009, στις 9 Μαρτίου, συγγνώμη, δεν μπορούσα να γνωρίζω ότι το Συμβούλιο θα έλεγε ότι είναι πολύ καλά αυτά, μπορείτε να προχωρήσετε. Για το Κανκούν, να σας πω ότι η στρατηγική που παρουσίασα εγώ στις αρχές Μαρτίου, η σταδιακή προσέγγιση για την Κανκούν, Νομίζω ότι αυτή είναι πλέον η συνολική προσέγγιση. Η προσέγγιση που οι περισσότερες χώρες θα πούν ότι αυτή είναι η μόνη οδός να προχωρήσουμε. Αν θέλουμε να διαβεβαιώσουμε θα χρησιμοποιήσουμε την ορμό που έχουμε αυτή τη στιγμή και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε αποτελέσματα στο Κανκούν. Χαίρομαι που αυτό κυριάρχησε. Τελευταία σας παρουτήρηση για το G77 και το πώς το βλέπουν. Ε, συμφωνώ, είναι ένας από τους χώρους ο οποίος χρειάστηκε να αλλάξει λίγο και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θεωρώ ότι ήταν κρίμα που το Σεπτέμβριο στη συνάντηση των διαπραγματευτών η Ευρώπη κατηγορήθηκε ότι σκότωσε το Κιώτο. Δεν κατάλαβα υπό ποια λογική θα πρέπει να κατηγορούμεθα εμείς ότι εμείς το κάναμε αυτό ενώ εμείς το έχουμε δεκτεί, έχουμε δεσμευτεί για το Κιώτο και έχουμε δώσει και αποτελέσματα βάσει του Κιώτο. Βέβαια, αν κανένας άλλος δεν θέλει να είναι εκεί και δεν θέλει ε, να βελτιώσει τις αδυναμίες του Κιώτο, οι αναπτυσσόμενες χώρες, το G77, θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν είμαστε εμείς το πρόβλημα για το Κιώτο. Οι χώρες που δεν θέλουν να συμμετέχουν στο Κιώτο και δεν έχουν και καμία άλλη αναλλακτική λύση, δεν έχουν προτείνει τίποτα για το πώς μπορούμε να έχουμε μια νομικώς δεσμευτική συνθήκη, ενώ ισχυρίζονται ότι αυτό θέλονται, αυτές είναι αυτές που πρέπει να αποδείξουν κάτι ενώπιον των αναπτυσσόμενων χωρών. Η δικιά μου η άποψη είναι ότι καλό θα ήταν εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ε, δεχόμαστε τις ευθύνες όταν δεν είναι δικές μας. Έχετε απόλυτο δίκιο, λέει ο Πρόεδρος. Μαθαίνουμε από τις διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Εθνών ότι δεν είμαστε εκείνοι που θα πρέπει να κάτσουν στο δόλο του κατηγορουμένου, αλλά κάποιοι άλλοι που προσφέρουν λιγότερα από εμείς. Έχω 7 ακόμη εγγεγραμμένους. Δύο λεπτά λοιπόν με μεγάλη αυστηρότητα γιατί έχω πολύ λίγο χρόνο στη θέση μου έτσι ώστε να μας ε, απαντήσει και η επίτροπο. Δύο λεπτά και το χρονόμετρο τρέχει παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε κύριε Λεπάζ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. τρει ερωτήσει πολύ σύντομε. Καταρχάς υπάρχει κρίση εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Την βλέπουν, την αισθάνονται πολλοί από του συμπολίτε μα και ω προ τη σημασία των κλιματικών αλλαγών και των μελετών του GED. Ερωτώ λοιπόν τι σκοπεύετε να κάνετε έτσι ώστε να αποκαταστήσετε την εμπιστοσύνη που χρειάζεται για να υλοποιηθούν αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι, του οποίου και εμεί συμμεριζόμαστε. Επίσης, θεωρείτε ότι μπορούμε να επηρεάσουμε, να τροποποιήσουμε τις οδικές μεταφορές όταν όλες οι άλλε οικονομικέ δραστηριότητε άλλο αποτέλεσμα δεν έχουν παρά να την ενισχύουν. Αναφέρομαι στο, στο ε, ηλεκτρονικό εμπόριο, e-commerce, το οποίο διαρκώς και δημιουργεί περισσότερη ανάγκη για οδικές μεταφορές και το ζήτημα των εκπομπών των μονάδων ε, που θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να πείσουμε τους βιομηχάνους, τις βιομηχανίες να επενδύσουν στην πράσινη οικονομία για να επιτύχουμε τον, στην πράσινη παραγωγή, για να επιτύχουμε το στόχο του 30% και που αποτελεί ταυτόχρονα αυτό, εκεί πρέπει να τους πείσουμε και το μόνο τρόπο να επανεκβιομηχανιστεί η Ευρώπη για να βγει και από την οικονομική κρίση. Ευχαριστώ κύριο Σκυλακάκης παρακαλώ. Thank Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ. Εγώ θέλω να επανέλθω στο σύστημα της εμπορίας λέτε πως ε, μπορούμε να φτάσουμε στο 30%. Εάν το κάνουμε αυτό, θα κοιτάξετε να βελτιώσετε την ομοθεσία της εμπορίας, ειδικά όσον αφορά τα εξαιρετικά κέρδη, τα έκτακτα κέρδη. Είχαμε έκτακτα κέρδη αυτή την περίοδο λόγω κρίσεως. Θα έχουμε έκτακτα κέρδη όταν θα ξεκινήσει το, προ... το σύστημα ε, γεωγραφικά προστατευόμενες από τον ανταγωνισμό εγκαταστάσεις. Ε, θα έχουμε εκεί πέρα μπόνους ε, διαρροής άνθρακα. Θα κοιτάξετε αυτά τα έκτακτα κέρδη και να λάβετε υπόψη το κόστος μεταφορών την επόμενη φορά, εάν πάμε στο 30%. Ευχαριστώ Βιτόριο Πρόντι. Ευχαριστώ κυρία Πίτροπε για την παρουσία σας εδώ. Αύριο μεταβαίνω στη Νέα Υόρκη για τη συνεδρίαση για τους αυτόχθονους λαούς. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να διασυνδεθεί και με την πολιτική ε, διαφύλαξη των δασών και θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι και αυτή που θα μπορούσε να φέρει τα πιο γρήγορα αποτελέσματα εάν μπορέσουμε να έχουμε αμέσω του διαθέσιμους, τους διαθέσιμους πόρους. Θεωρείτε ότι μπορούμε να δώσουμε κάποια ελπίδα στους πληθυσμούς αυτούς, ότι θα μπορέσουμε δηλαδή να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά τους με συστημικό τρόπο βάσει αυτού και να προσφέρουμε και τις κατάλληλες εγγυήσεις ώστε να είναι οι ίδιοι οι φύλακες αυτών των δασών να διαφυλάξουν την βιοπικιλότητα και την, ε, τις δυνατότητες που έχουν να ε, αποτρέψουν την αλλαγή του κλίματος. Υπάρχει και αυτή η κοινή ευθύνη παρά το γεγονός ότι είναι διαφοροποιημένη. Εγώ μέχρι τώρα δεν έχω δει κάποιες ε, σοβαρές πολιτικές προτάσεις επί του θέματος αυτού. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε να δίνουμε αυτές τις απαντήσεις διότι θα πρέπει να έρθει κάποια στιγμή και αυτή η παγκόσμια συνένεση την οποία έχουμε ανάγκη. Ευχαριστώ. Να δούμε πώς θα κρίνεται και την ε, σχετική και τη διάσκεψη για το κλίμα και τη δικαιοσύνη και τα λοιπά όλα αυτά τα θέματα που ενδιαφέρουν τον κύριο Πρώτη με την διάσκεψη που έγινε πριν από μια εβδομάδα περίπου από Έλληνα εκπροσώπους ε, με έτοιμα να εκδικάζεται η περιβαλλοντική ε, εγκληματικότητα από τα παιδικά δικαστήρια και την πρόταση για το δημοψήφισμα. Γιούλη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Μια ερώτηση έχω μόνο και θα ήθελα να μου δώσετε την απάντηση γιατί έχω επανέλθει πολλές φορές. Την έχω υποβάλει πολλές φορές και θα συνεχίσω να την υποβάλω μέχρι ότου πάρω τις απαντήσεις μου. Το ερώτημα του εάν μιλούμε με μία φωνή στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Στην Κοπενχάγη 28 κράτη-μέλη ήμασταν, δεν μπόρεσαν να μιλήσουν μια φωνή. είναι 28 εκπρόσωποι. Ερωτώ λοιπόν και ρωτώ και πάλι γιατί έχω ξανακαταθέσει την ερώτηση. Μπορείτε να εξασφαλίσετε αποκλαστική εντολή εκπροσώπηση Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κλιματικές διαπραγματεύσεις ή υπάρχει τουλάχιστον μια δυνατότητα ad hoc, αν δεν μπορείτε να έχετε ε, να έχετε μια μόνιμη εντολή, μια πάγια εντολή, τουλάχιστον για το κανκούν ad hoc. Ή θεωρείτε ότι δεν χρειάζεται αποκλειστική εντολή. Και δεν τρέφεται πλέον ελπίδες για μια θετική έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων για το κλίμα του κανκούν. Ευχαριστώ, Σλίτερ. Ευχαριστώ. Ο γιο μου, αφού εξέφρασε την υποστήριξή του στη μείωση 30% προ την Επίτροπο, αποφάσισε να πάει για ύπνο. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξή. Ναι, θα έπρεπε να γίνει μια πρόταση για τις εκπομπές από τα αυτοκίνητα. Από την Επιτροπή περιμένω να μου πείτε λοιπόν τι προβλέπετε και επίσης για την, ε, αερο... για την ε, αεροπορία και τα στοιχεία τα σχετικά με τα οξύδια του αζότου. Έχετε κάποια συγκεκριμένη πρόταση ξεκινήσει στην Επιτροπή, στο pipeline όπως λέμε. Ευχαριστώ, Ματίας Χρότε. Ευχαριστώ, δυστυχώς άργησα να έρθω, αλλά θα ήθελα παρόλα αυτά να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Αναφέρθηκαν τα ελαφρά φορτηγά και χαίρομαι για το ότι αναφέρατε το Euro 5, Euro 6, ότι δεν θα είναι η καταστροφή της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά από ό,τι φαίνεται ότι δεν είχε διαφορά στο κόστος σχετικά, με πάση περιπτώσει. Και μάλιστα ε, η κρίση κατέδειξε πως ε, το κάναμε αυτό την κατάλληλη στιγμή. Και αυτό γιατί υπάρχει και ασφάλεια για τις επενδύσεις στην αυτοκινητομηχανία αλλά και για τους πελάτες όσον αφορά την νομοθεσία. Τώρα πίεση κόστους στα ελαφρά φορτηγά, τα οποία διακρίνονται από τα γιοταχή. Εδώ πέρα συμφωνώ με τον συνάδελφο. Γιατί αυτοί οι οποίοι αγοράζουν αυτοκίνητο δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Οπότε ένα μέτρο εδώ πέρα θα μπορούσε να είναι νομίζω να υπάρχουν για τα μεγαλύτερα φορτηγά κάποιοι περιορισμοί της ε, ταχύτητας και είχαμε και μία συνάντηση νομίζω με τις υπηρεσίες σας και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να επανεξετάσετε αυτό το μέσο. Ε, γνωρίζω πως ε, μπορεί να μην υπάρχει ακόμα στον κύκλο των δοκιμών, αλλά όπως ξέρετε στον ε, πραγματικό κόσμο με την ταχύτητα αυξάνεται στο τετράγωνο η αντίσταση του αέρα και άρα η κατανάλωση της βενζίνης. Οπότε δείτε αυτό το μέτρο. Θα έχει και αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος και θα, βοηθού, θα τους βοηθούσαμε όλους νομίζω. Για δείτε το όριο ταχύτητας ε, στην νομοθεσία. Ε, ευχαριστώ. Βεβαίω, στη Γερμανία έχουμε τελείω ε, διαφορετικά όρια ταχύτητας. Λοιπόν, Άννα Ρόσμπαχ. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ που ήρθατε. Ακούσαμε πολλά, πολλές θεωρητικές αλλά και σημαντικές ερωτήσεις, αλλά εγώ θα ήθελα λίγο να επανέλθουμε στην πραγματικότητα. Γιατί εγώ ανησυχώ για το πώς θα εφαρμοστούν στην καθημερινότητα των πολιτών αυτές οι ωραίες ιδέες. Εντάξει, οι μεγάλες εταιρείες θα αλλάξουν τον τρόπο παραγωγής, θα βάλουν φίλτρα στις τσιμινιέρες και τα λοιπά, αλλά ο μέσος πολίτης ο οποίος δεν είναι συνδεδεμένος με κεντρική θέρμανση, όταν λέω κεντρική εννοώ ανασυνοικίες, ε, είναι σε απομονωμένη κατοικία στην Ήπεθρο, πώς θα αλλάξει εκείνος καύσιμο για την θέρμανση. Το επόμενο ερώτημά μου είναι, αναρωτιέμαι τι σκέφτεται να κάνει η Επίτροπος για την αναβάθμιση των ε, γραμμών ε, συγκοινωνιών υψηλής ταχύτητας. Είδαμε τώρα την κρίση με τις αεροπορικές ε, εταιρείε ε, και είδαμε πόσο δύσκολο είναι να μειωθούν οι αεροπορικές συγκοινωνίες. Νομίζω ότι τώρα λοιπόν υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα, ρεαλιστική πιθανότητα επιτυχίας για συγκοινωνίες υψηλής ταχύτητας και τώρα νομίζω για τρένα υψηλής ταχύτητας και να να δούμε τι θα γίνει. Βεβαίω δεν ξέρω αν μπορούμε να εισαγάγουμε τρένα, αλλά νομίζω εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι μπορεί να γίνει. Με εδώ πέρα λοιπόν κλείνω ο καταλόγο ομιλητών. Πρώτα απ' όλα για την Ανά Να απαντήσω σε σένα. Ε, εξαιρετικό το ερώτημά σου. Το ευκολότερο, ευκολότερος τρόπος για να ενσωματώσουμε τους πολίτες είναι τα προϊόντα που αγοράζουν, είτε είναι το στιέρα είτε αυτοκίνητο. Δηλαδή ε, να υπάρχει μια λογική τεχνολογία που εξοικονομεί ενέργεια και χρησιμοποιείται στην παραγωγή. Και νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά, ενημερώνουμε τους πολίτες και βλέπουμε τα αποτελέσματα ήδη και στη Δανία και σε άλλες χώρες ε, πράγματι μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας αλλά πράγματι η συζήτηση αυτή σχετίζεται και ε, με το πώς ε, θα το κάτι τέτοιο οι πολίτες. Δηλαδή, εάν όλη η Ευρώπη μείνει στάσιμη και ο υπόλοιπος κόσμος προχωρήσει, τότε βέβαια αυτό θα κοστίσει σε ευημερία και αυτή τη σχέση πρέπει να τονίσουμε τώρα. Θα είμαι σύντομη γιατί είχαμε ακούσει πράγματι και την άλλη φορά την πρόταση σας για το όριο ταχύτητας. Να δούμε τι θα προκύψει ε, ω σύσταση του Κοινοβουλίου και θα το, θα το εξετάσουμε όπως συμφωνήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Καρλ Σλούτερ ρώτησε για το μονοξίδιο του αζότου και τις ετικέτες ε, των αυτοκινήτων για τις ετικέτες των αυτοκινήτων θα έλεγα πως δεν έχουμε ακόμα χρονοδιάγραμμα. Είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό θα αναφερθεί στην αυριανή ανακοίνωση. Γνωρίζω πως στην προηγούμενη θητεία Κοινοβουλίου και Κομισιόν είχαν γίνει κάποιες συζητήσεις. Τώρα για εμένα, και αυτό σχετίζεται με αυτό το οποίο είπε η Άννα είναι πάρα πολύ λογικό να διαφημίζουμε ένα αυτοκίνητο και εγώ ως καταναλωτής να βλέπω τι κατανάλωση ενέργειας έχει. Είναι εύκολο. Είναι απλά θέμα να το κάνουμε. Και να είναι διαφανές για τους ανθρώπους. Τώρα για αυτό το οποίο είπατε να μιλάμε μία φωνή δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά είναι σημαντικό. Μην πιστεύετε ότι το να μιλάμε με μία φωνή σημαίνει πως ε, μόνο μία φωνή θα είναι η ευρωπαϊκή φωνή. Πολύ διαφορετικοί άνθρωποι μπορούν να εκπροσωπήσουν την Ευρώπη. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να έχουν το ίδιο μήνυμα. Το μήνυμα να μην μπερδεύει τους άλλους. Τους ανθρώπους με τους οποίους διαπραγματευόμαστε δηλαδή. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καλύτεροι όσον αφορά την παρουσίαση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων και να μην ξοδεύουμε όλοι μας την ενέργεια να συμφωνήσουμε εμεί μεταξύ μας και στο τέλος να μην μπορούμε να παίξουμε τα χαρτιά μας στο διαπραγματευτικό τραπέζι. Και να διορθώσω κάτι άλλο, γιατί είπατε πως δεν έχω πολλές ελπίδες για το Κανκούν. Κοιτάξτε, θεωρώ πως εάν λέγαμε πως ο στόχος μας είναι να επιτύχουμε όλα όσα δεν επιτύχαμε στην Κοπενχάγη, τότε διατρέχουμε τον κίνδυνο να μην κάνουμε τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, ούτε ο κόσμος ούτε το κλίμα δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια. Οπότε να πάρουμε τη συμφωνία της Κοπενχάγης και να μπει σε επίσημες διαπραγματεύσεις. Οι δύο βαθμοί, η γρήγορη χρηματοδότηση που πρέπει να ξεκινήσει το αργότερο στο Κανκούν. έμαρβη ε, Για την δασοκομεία είχαμε πρόοδο στην Κοπενχάγη, για την προσαρμογή, για την τεχνολογία. Υπάρχουν πολλές αποφάσεις που πρέπει να γίνουν επίσημες, οπότε έχουμε αρκετά πράγματα συγκεκριμένων αποφάσεων που θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα στο Κανκούν. Εάν ξεκινήσουμε να συζητάμε μόνο τη νομική πτυχή, ο κίνδυνος είναι να μην κάνουμε τίποτα για να μην έχουμε συγκεκριμένες αποφάσεις στο Κανκούν. Αυτό είναι ο στόχος μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω φιλοδοξία, είναι να δούμε τα σίγουρα στο Κανκούν χωρίς να μας εμποδίζει η νομική συζήτηση να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα. Κορίν μετά Λεπάζ για την κρίση εμπιστοσύνη των πολιτών. Είναι πολύ πολύπλοκο τώρα να απαντήσω. Βασικά εγώ δεν έχω δει τίποτα Α, που να έχει βγει από το IPCC που να αλλάζει κατά βάση την πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Ναι εντάξει κάποια λάθη να διορθωθούν αλλά κατά βάση η πρόκληση υπάρχει και όλοι πρέπει να βδούν και να συνειδητοποιήσουν ακόμη και όσοι είναι σκεπτικιστές πως ε, ούτως ή άλλως θα γίνουμε 9 δισεκατομμύρια όταν, τα, όταν φτάσουν τα παιδιά μου στην ηλικία μου. Οπότε πρέπει ούτως ή άλλως να είμαστε πιο αποτελεσματικοί για τις εκπομπές και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε στους πολίτες Ευρώπης. Επίσης λέτε πώς μπορούμε να πείσουμε τη βιομηχανία πως ε, οι επενδύσεις στην πράσινη οικονομία είναι η μόνη δυνατότητα να υπάρχει βιομηχανία στην Ευρώπη. Παρά το ότι κάποιοι το καταπολεμούν αυτό, νομίζω πως ε, το έχουν λάβει οι, τα μεγάλα κεφάλια της βιομηχανίας το, το μήνυμα. Και ορισμένοι πρωτοπόροι είχαν, ε, θα συγκεντρωθούν εδώ πέρα στις 17 Μαΐου. To convey the message για να τους δώσω το μήνυμα πως οι πρωτοπόροι ξέρουν πως πρέπει να είναι ισχυροί εδώ ή θα χάσουν την θέση τους και όσο περισσότερα τέτοια παραδείγματα βρούμε τόσο το καλύτερο νομίζω εδώ πρέπει να το δούμε και επικοινωνιακά. Τέλος, ο κύριος Κυλακάκης ρώτησε για το σύστημα εμπορίας εκπομπών και τα έκτακτα κέρδη δύσκολο ερώτημα. Σύντομη απάντηση. Νομίζω πως όσο πιο α, επακριβώς μπορούμε να κατανοούμε τους πόρους, λιγότερα έκτακτα κέρδη θα δούμε και νομίζω πως ε, όπως προχωράμε πρέπει να βελτιώνουμε τους μηχανισμούς συστήματος εμπορίας. Εάν δείτε το τι θα σας παρουσιάσω τους επόμενους ε, δέκα μήνες, υπάρχουν πολλές βελτιώσεις του συστήματος εμπορίας. Και ο Βιτόριο Πρόντι με ρώτησε για τους αυτόχθονες λαούς. Είναι ένας ε, τομέας που είχαμε σημαντική πρόοδο. Ξέρετε, οι Αμερικανοί πάντα είχαν αυτή την αντίσταση για τους αυτόχθονες, όπως τους λέμε εμείς, για τη διατύπωση δηλαδή και εκεί πέρα νομίζω στα της δασοκομείας είχαμε σημαντική πρόοδο. Και τέλος για την ε, διαφοροποίηση. Έχω ακούσει τα της κλιματικής δικαιοσύνης και είναι δύσκολο γι' αυτό ακριβώς να συμφωνήσουμε με τους στόχους του 2015, αλλά θέλω να πω πως παρά το ότι δεν είναι δίκαιο, είναι γεγονός πως χωρίς ε, μακροπρόθεσμα κάποια συνεισφορά από οικονομίες όπως τη Βραζιλία, την Ινδία, την Κίνα, ο κόσμος έχει ξεφύγει τόσο πολύ που δεν θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή όπως θα θέλαμε. Αλλά ο λόγος για τον οποίο οι οικονομίες αυτές δεν θα του ζητηθεί να κάνουν τίποτα ουσιαστικό βραχυπρόθεσμα είναι γιατί υπάρχει αυτή η γενική αναγνώριση πως βεβαίως πρέπει να υπάρχει μια διαφοροποίηση. Και εκεί πέρα έχουμε την ευθύνη και αυτό το συνδέω με αυτό το οποίο είπα ήδη για την σημασία του ότι η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να είναι πρωτοπόρος σε αυτόν τον τομέα. Πράγματι είναι και προ το δικό μας συμφέρον, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αξιοπιστία την νομοποίηση, δηλαδή εμείς που είμαστε τυχεροί και ζούμε στα μέρη κοινά του κόσμου που εφημερούν, έχουμε και μια ιδιαίτερη ευθύνη. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Σας ακούσαμε μεγάλη προσοχή. Βλέπατε κι εσείς ότι και έχουμε υψηλούς στόχους και φιλοδοξίες και θέλουμε ως Επιτροπή να σας υποστηρίξουμε. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία λοιπόν, έχοντας για άλλη μια φορά την ευκαιρία να σας δούμε και ελπίζουμε ότι θα σας ξαναδούμε και πριν από το Κανκούν. Για να με ενημερώσετε για μια κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ και κάθε επιτυχία. Και τώρα πάμε στο επόμενο θέμα τη ημέρα τη διάταξη, το υπαριθμό 5. Πρόκειται για τα ψευδεπίγρα... ψευδεπίγραφα φάρμακα. Τροποποίηση οδηγία 2001-83. Η Μαρίσα Ματία είναι η συγκήτρια. Έχουμε πολλέ τροπολογίε συμβιβαστικέ. Και παρακαλώ αφού αφήσουμε να παρέλθουν ένα-δύο λεπτά για να φύγουν εκείνοι που ενδιαφέρονται κυρίως για την προστασία του κλίματος και να μείνουν όσοι ενδιαφέρονται και τα υπόλοιπα θέματα, αφού βέβαια όσοι αποχωρούν ανταλλάξουν και απόψεις, so, could I ask those who want to leave the room do so, because we now continue. Παρακαλώ λοιπόν να αποχωρήσουν όσοι είναι να αποχωρήσουν για να συνεχίσουμε εμείς με το θέμα της Μαρία Ματίας και τα ψευδεπίγραφα φάρμακα. Μαρία, Μαρίσα, έχεις το λόγο να μας παρουσιάσεις uh, τις συμβαστικές κυρίες αλλά και τις υπόλοιπες. E Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη μικρή παρουσίαση πριν από την ε, ψηφοφορία. Εδώ συζητάμε πώς μπορούμε να προασπίσουμε καλύτερα την υγεία των εκατομμυρίων ε, Ευρωπαίων πολιτών και να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούν να εμπιστεύονται περισσότερο τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούν, ε, αποφεύγοντας να έχουμε ψευδεπίδερα γραφά φάρμακα στην αλυσίδα διαμονής θα πρέπει να είναι βέβαιοι οι ασθενείς ότι τα φάρμακα τα οποία καταναλώνουν θα πρέπει να είναι αυτά που πρέπει να καταναλώνουν. Αυτό θα πρέπει να είναι βεβαιότητα πάντα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς για ε, την βοήθεια και την διαθεσιμότητα των σχεδόν εισηγητών. Η βοήθειά τους ε, μου επέτρεψε να βελτιώσω την πρόταση του κειμένου μου και χάρη στην ε, συνδρομή τους νομίζω ότι φτάσαμε και σε ευρία υποστήριξη η οποία εκφράζεται και στις 15 συμβιβαστικές τροπολογίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ευρωβουλευτές που παρουσίασαν τροπολογίες στην αρχική έκθεση. Ε, για την οποία θα κάνω και κάποια σχόλια. Όπως σας είπα και πριν, καταλήξαμε σε πολύ σημαντικούς συμβιβασμούς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να έχει λοιπόν μια στεναρή θέση για όλα τα σημεία τα οποία ε, συζητούνται. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να συμβιβάσουμε τις, τα διαφιλονικούμενα συμφόροντα με ένα κοινό γνώμονα. Έχουμε τρεις βασικούς ε, και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτούς εν συντομία. Καταρχάς θα πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο ορισμό για το ψευδεπίγραφο ε, φάρμακο. Αυτός είναι ο συμβιβασμός υπαριθμών 6. Είναι πάρα πολύ σημαντικός διότι ένα ψευδεπίγραφο φάρμακο είναι αυτό το οποίο παραποιείται ε, σκοπίμως και Στόχος είναι να αποκρύψει την ε, αρχική του ταυτότητα. Ο ορισμός αποκλεί κάποια ελαττωματικά προϊόντα και δεν συσχετίζεται και με παραβιάσεις νομοθεσίας για την ε, πνευματική ιδιοκτησία. Δεύτερον, διατάξεις ασφαλείας. Συμβιβασμοί 7 έως 10. Έγιναν αρκετές προτάσεις εδώ και νομίζω ότι αυτός ήταν ο τομέας στον οποίο υπήρχαν οι πιο διστάμενες απόψεις. Κάποιες ε, αναφέρονται σε συγκεκριμένες υποχρεωτικές ε, διατάξεις ε, για όλα τα φάρμακα, κάποιες άλλες αναφέρονται στις ελαχιστοποίησεις του κινδύνου, κάποιες αναφέρονται στη διαφορά μεταξύ φαρμάκων τα οποία δίνονται με ιατρική συνταγή και φαρμάκων που δίνονται χωρίς. Η λύση στην οποία καταλήξαμε δεν αποκλείει κανένα φάρμακο, αλλά κάνει μία πρόταση πολύ λογική εκ παραλίλου. Θα πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικές απαντήσεις οι οποίες θα βασίζονται στην πραγματικότητα. Α, σε πρώτη φάση θα πρέπει να έχουμε καταρχάς ε, τα φάρμακα τα οποία παρέχονται με ιατρική συνταγή, τα οποία είναι και τα πιο επικίνδυνα για τους ασθενείς και είναι και αυτά τα οποία παραποιούνται περισσότερο τα πρώτα χρόνια θα γίνει μια συστηματική και πολύ αυστηρή ανάλυση της κατάστασης και στα πρώτα τέσσερα χρόνια η έναρξη ισχύω της οδηγίας και οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να αποφασίσουμε για το κατά πόσο θα πρέπει να ε, το πεδίο εφαρμογή. Αυτά τα τέσσερα χρόνια θα μπορέσουν να βοηθήσουν και τα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν προς την νομοθεσία. Τρίτο συμβιβασμό, πωλήσει μέσω διαδικτύου, συμβασμοί 12 και 13. Εδώ ε, συμφωνούμε όλοι, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε από την νομοθεσία τη μεγαλύτερη δυνατότητα εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στον ευρωπαϊκό χώρο. Πρέπει να γίνει βέβαια διάκριση μεταξύ παράνομων και νόμιμων φαρμάκων. Ε, και φυσικά θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας χώρος ασφάλειας. Ε, το να υπάρχει κοινοτική νομοθεσία, να υπάρχει ένας κατάλογος ε, εγκεκριμένων online φαρμακείων, ο οποίος θα πρέπει να επικαιροποιείται συνεχώς και θα πρέπει να ενισχύσουμε και τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για όλους όσους ε, αγοράζουν από φαρμακεία τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα. Τέταρτο σημείο, κύριε Πρόεδρε, Επιθεωρήσει. Και εδώ αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στο συμβιβασμό 14, ο οποίος ε, βασίζεται σε έκτακτους ελέγχους ε, χωρίς πρώτερη προειδοποίηση από τις αρμόδιες αρχές ε, για την εποπτεία υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Ο συμβιβασμό 11, η πέμπτη πρόθεση, αναφέρεται στην προστασία των δεδομένων των ασθενών. Δεν θα πρέπει να ε, διακυβεύεται η εμπιστευτικότητα, θα πρέπει να διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών δεν θα χρησιμοποιούνται για εμπορικού σκοπούς. Έκτον, κυρώσει. Και εδώ ολοκληρώνω με τις συμβιβαστικές προτάσεις. Ε, αναφέρομαι στο συμβιβασμό 1 σε αυτή την περίπτωση. Και εδώ υποστηρίζουμε τη νέα σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την παραποίηση των φαρμάκων και ανάλογες ε, παράνομες πράξεις οι οποίες ε, διακυβεύουν την δημόσια υγεία. Ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν ανάλογες κυρώσεις ε, για την παραποίηση των φαρμάκων. Κάτι τελευταίο για τους συμβιβασμούς αυτούς. Δύο πράγματα τα οποία έχουν σχέση με δύο τροπολογίες αντιστοίχως. Ο συμβιβασμός 15, ο οποίος γράφει should, θα πρέπει να αλλάξει σε shall, διότι έχουμε άρθρο εδώ και δεν είναι εκτιμώντα, Όσον αφορά τώρα στον ε, συμβιβασμο Α11 για την προστασία δεδομένων, δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποια αναφορά στις, στα φαρμακεία. Για να παρακολουθούμε αποτελεσματικά τα φάρμακα θα πρέπει να συμπεριλάβουμε όλη την αλυσίδα διανομής και επομένως δεν θα πρέπει να αναφέρονται τα φαρμακεία συγκεκριμένα. Επίσης δεν θα πρέπει να δημιουργείται πρόβλημα με την εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Ολοκληρώνοντας να πω ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς οι οποίοι δεν καλύπτονται στις συμβιβαστικές προτάσεις και θα πρέπει να αποφασιστούν αύριο. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες στις οποίες είμαι αντίθετη και εδώ προτείνω αρνητική ψήφο και σε κάποιες άλλες συμφωνώ. Ε, αλλά υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες τις οποίες με βρίσκει σύμφωνη με το περιεχόμενο, αλλά προτείνω αρνητική ψήφο γιατί περιλαμβάνονται στους συμβιβασμούς που σας ανέφερα και ή προτείνονται σε άλλες παραγράφους του ίδιου άρθρου. Γι' αυτό λοιπόν ε, δεν ε, υπάρχει λόγος να ε, τις δεχτούμε. Σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν η ψήφος θα πρέπει να είναι αρνητική, διότι θέλουμε να διασφαλίσουμε τη συνοχή του διατακτικού και να μην έχουμε επαναλήψεις να επισημάνω επίσης ότι έχουμε μία στεναρή βάση συμφωνίας και πολιτικές θέσεις οι οποίες θα μπορέσουν να μας οδηγήσουν σε μία ισχυρή θέση του Κοινοβουλίου χωρίς να δημιουργήσουμε προβλήματα στο γενικότερο πνεύμα της οδηγίας. Γι' αυτό λοιπόν είμαι στη διάθεσή σας για να ακούσω όλες σας τις προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λοιπόν την εισηγήτρια. Είναι η πρώτη της έκθεση και σοβαρή υπόθεση και αυτά τα οποία βλέπουμε και ακούμε μας λένε πως πήγε καλά η συνεργασία. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για τη δουλειά που έχετε κάνει η οποία θα ωφελήσει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα έχουμε τα σχόλια και τις συμπληρώσεις ε, των σκιωδών. Φρανσουάς Γκροστέτ λοιπόν beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais m'associer. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια όπως και εσείς για την εξαιρετική δουλειά της και για το γεγονός ότι άκουσε τα σχόλια μας και προσπάθησε κατά το δυνατόν να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις μας. Ως προς τις συμβαστικές τροπολογίες, συμφωνώ εν γέννη με τις τροπολογίες αυτές κυρίως στην πρώτη θα ήθελα να επισημάνω εκεί που γίνεται λόγος για την διεθνή διάσκεψη για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα και ενώ γνωρίζουμε ότι θα πρέπει η Ευρώπη να υιοθετήσει στις 11 Μαρτίου, Μαΐου μια πρώτη πρόταση, σημειώνω ότι πρόκειται για μια πρώτη προσπάθεια σε οικουμενικό επίπεδο με συνδρομή και τη δυνατότητα να καταστούν συμβαλόμενα μέρη και τρίτα κράτη. Μια προσπάθεια λοιπόν πρέπει απολύτως να υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ίντερνετ που είναι αυτό που λέμε βασιλική οδός για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, για την πώλησή τους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ελέγξουμε την πώλησή τους μέσω του ίντερνετ και να ξεκινήσουμε εκστρατείες ενημέρωσης και δεστοποίησης. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται πιστεύω μία, ε, μία οδηγία η οποία θα ρυθμίσει το παράνομο εμπόριο ψευδεπίγραφων προϊόντων στο ίντερνετ. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το αναλάβει αυτό η Επιτροπή. Πρέπει να τους το στήσουμε. Για, τα... για τις διατάξεις ασφαλείας. Πολλές νοτροπολογίες που έχουν διατυπωθεί είναι απαραίτητο να καταστούν υποχρεωτικές οι διατάξεις ασφαλείας για τα φάρμακα χωρίς συνταγή. Τώρα ασχολούμαστε με αυτά τα οποία χορηγούνται με συνταγή ιατρική. Θα πρέπει λοιπόν μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να αποφασιστεί να συμπεριληφθούν και αυτά στι ε, διατάξεις ασφαλεία. στο διατακτικό. Και ναι, μεν πιστεύω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τι συμβαστικέ ε, τροπολογίε, αλλά προσωπικώ και το υπογραμμίζω προσωπικώ έχω ιδιαίτερε επιφυλάξει ω προ το packaging τη συσκευασία, Τροπολογίε, συμβαστικέ 7 και 8. Δηλαδή, άπαξ και έχει λάβει την άδεια για τη διάθεση στην αγορά ένα προϊόν πάνω στην συσκευασία του θα πρέπει να παραμένει αυτή αμετάλλακτη, να μην παραβιάζεται δηλαδή, μέχρι την ώρα που φτάνει στον καταναλωτή. όπως γίνεται και με τα τρόφιμα. Το ίδιο που είχαμε και με το lever boxing που μιλούσε για, τις αρχικές, για την αρχική συσκευασία. Νομίζω ότι θα υπάρξει δυσκολία, γιατί ξέρω ότι κάποιοι συνάδελφοι διαφωνούν και δεν θα δεχθούν εύκολα αυτές τις προτάσεις. Πλην όμως, εάν δεν γίνει δεκτή αυτή η πρόταση, θα παρακαλέσω στο πλαίσιο της ε, τροπολογίας υπαριθμών 10 να εισαγάγουμε την διαλειτουργικότητα. Και τότε την απέτηση για τη διαλειτουργικότητα θα πρέπει να την εισαγάγουμε στην διάθεση του ε, φαρμάκου και αν υπάρξει διαφορά μεταξύ δύο κρατών μελών θα πρέπει να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα με κοινό αριθμό, συριακό αριθμό και εναρμόνιση συστημάτων. Διαλειτουργικότητα λοιπόν των φαρμάκων, των στοιχείων των φαρμάκων και εδώ θα πρέπει να επιμείνουμε ιδιαίτερα. Και επίση για την εναρμόνιση των συστημάτων ασφαλεία, η τετραετής περίοδο μου φαίνεται ικανοποιητική. Για την υπαριθμόν 9 συμβιβαστική τροπολογία. Τα ε, ανώνυμα λεγόμενα φάρμακα, τα generic δηλαδή, θα έλεγα ότι εφόσον αυτά υπάγονται σε ιατρική συνταγή, θα πρέπει να υπαχθούν στην οδηγία με την ανάλυση του κινδύνου. Γιατί μιλούμε και αγωνιζόμαστε για την υγεία των πολιτών. Εκεί πρέπει να είμαστε απαιτητικοί. Η ε, αντιγραφή δεν ε, γίνεται μόνο με γνώμονα την τιμή ενός προϊόντος, αλλά και με γνώμονα τους όγκους πώληση. Και ξέρουμε ότι ορισμένα πολύ σημαντικά και δεδομένα φάρμακα σύντομα θα κυκλοφορούν κυρίως ε, έξω από τις ε, μάρκες ε, τις φαρμακευτικές ως generic δηλαδή και σε αυτά θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή. Για τη 14. Είναι πιστεύω απαραίτητο να ενισχυθεί το επίπεδο των επιθεωρήσεων και σε τρίτα κράτη. Πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό για να περιοριστεί και ο κατάλογος των ε, κρατών που έχουν υποτίθεται προδιαγραφές αντίστοιχες με τις Ευρωπαϊκές Ένωση. Κάτι δηλαδή πάνω απ' όλα που έχουν ε, ε, συμφωνήσει αμοιβέ αναγνώριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί πέρα πρέπει ιδιαίτερα να δώσουμε έμφαση. Κατά τα ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι πάντοτε ιδιαίτερα απαιτητικό έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή προστασία των ασθενών. Ροτ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με την εισηγήτρια συνεργαστήκαμε καλά και θεωρώ πως οι 15 συμβιβαστικές τροπολογίες είναι πραγματικά υπόδειγμα συνδυαστικών τροπολογιών. Συνδυάζονται εδώ πέρα διαφορετικές απόψεις για να επιτύχουμε τον μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας στην πρώτη ανάγνωση ήδη στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο. Γι' αυτό προτείνω εγώ στην ομάδα μου να τις υποστηρίξουμε όλες και θα το κάνω και εγώ. Βεβαίως, όπως ξέρουμε, το ιδανικό δεν υπάρχει ποτέ, αλλά αν δούμε τι γίνεται στο Συμβούλιο, στην ομάδα εργασίας, είναι διαφορετική η προσέγγιση, όχι καταστροφικά διαφορετική όπως σε άλλα νομοθετήματα, όπως παραδείγματο χάρη στη συνοριακή παροχή υγείας ή στην πληροφόρηση του ασθενούς, αλλά παρόλα αυτά είναι όπως είναι πάντα το Συμβούλιο. Γι' αυτό πρέπει στην πρώτη ανάγνωση ήδη να συμφωνήσουμε ή να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στο Συμβούλιο. Ανεξαρτήτως του τι θα κάνουμε στη δεύτερη ανάγνωση. Δεν είναι τώρα η στιγμή να κάνουμε συμβασμούς με το Συμβούλιο. Το λέω αυτό προς κάποια μέλη της δικής μου ομάδας και άλλων ομάδων τροπολογίες ε, που θα κατατεθούν, που θα επαναλαμβάνουν το κείμενο του Συμβουλίου δεν μας βοηθάνε. Οι συμβιβασμοί που πρότεινε η συγγήτρια και αυτό το οποίο είπε Φανσός Κωστέτη είναι θετικά. Με όλα τώρα τα δευτερεύοντα εκείνα σημεία τα οποία αναφέρονται στην όλη συζήτηση, σαν να θέλουμε δηλαδή να δυσκολεύσουμε κάποιες πτυχές του εμπορίου. Εδώ πέρα επανερχόμαστε πάλι στον πυρήνα της νομοθεσίας που είναι να αποφευχθεί να αποφευχθούν τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, να μπορέσουμε δηλαδή να τα αναγνωρίσουμε όσο δυνατόν πιο νωρίς για να προστατεύσουμε τους ασθενείς. Αυτό είναι το θέμα μας εδώ πέρα, η προστασία της ανθρώπινης υγείας είτε από βλαβερά είτε από φάρμακα τα οποία δεν επιδρούν γιατί δεν έχουν δραστική ουσία. Οπότε πρέπει από την παραγωγή ήδη να γίνεται ένας εσωτερικός έλεγχος ε, του φαρμάκου και ίσως να βελτιωθεί αυτός ο έλεγχος όσον αφορά τα συστατικά οπουδήποτε και αν είναι στον κόσμο. Να αναφέρω κάτι άλλο τώρα το οποίο μου είναι ιδιαίτερα αγαπητό, θα έχουμε όλο και περισσότερα ψευδεπίγραφα φάρμακα που θα έχουν ψεύτικα συστατικά. Οπότε πρέπει να μπορούμε να βασιζόμαστε στους ελέγχους του κατασκευαστή. Και από πού προέρχονται αυτά τα φάρμακα είναι χώρες ε, στις οποίες δεν λέμε τίποτα γιατί είναι σημαντική εμπορική εταίρη και θέλουμε να τους πουλήσουμε, ξέρω εγώ, μετρό ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ θα ήθελα να είμαστε κάπως πιο σκληροί εναντί Κίνας, Βιετνάμ, Κορέας, Ινδίας, αλλά δεν έχω ψευδεστήσεις. Είμαστε εμείς και η Επιτροπή μας πολύ μικρή. Οπότε τουλάχιστον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διασφαλίσουμε πως ε, πλαστά συστατικά αλλά και συνολικά ψευδεπίγραφα φάρμακα πρέπει να ανοιχνεύονται. Οπότε πρέπει να δούμε ολόκληρη τη διαδρομή του φαρμάκου και αυτό δεν αφορά μόνο το εάν έχει ή όχι κάποια... κάποιο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που το προστατεύει, που πωλείται επίσης και αυτό αδιάφορο και που χρησιμοποιείται. Αλλά και εδώ πέρα παραπέμπω σε μία βεβαίως δική μου τροπολογία. Ένα είναι το σημαντικό. Εάν παίρνουμε στα σοβαρά την ε, ασφάλεια, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να ανοίγουν οι συσκευασίε, να σπάνε οι καρτέλες και να βγάζουν από μέσα τα χάπια. Πρέπει να τελειώσει αυτό. Μέσω πρόθεσμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Εάν είναι να εναρμονίσουμε, ε, δεν μπορεί να μην εναρμονίσουμε το μέγεθος της συσκευασία. Και αυτοί οι οποίοι μας δώσαν ε, πληροφορίες στο παρελθόν, αυτοί οι οποίοι μας είπαν ε, πως ε, ίσως θα προξενήσουμε και ζημία αν παρεμβούμε δυναμικά πρέπει να δουν και τι γίνεται στα, στα κρατημέλη. Γιατί υπάρχουν συσκευασίε των 10, 30, 50 κομματιών. Και εκεί πέρα υπάρχει το παράλληλο εμπόριο, γιατί δεν είναι δυνατόν να σπάνε ούτε οι καρτέλες, ούτε τίποτα. Δεν λείπει και ο κ. Χατζημαρκάκης τώρα. Το α και το ω λοιπόν είναι αυτό. Κάθε παραγωγός, κάθε διακινητής, κάθε έμπορος ε, πρέπει να τα δει αυτά. Τώρα τι γίνεται με αυτά που δίνονται χωρίς συνταγή εδώ πέρα υπάρχει ένας κίνδυνος για τους ασθενείς. Ναι, εντάξει, εάν αγοράζω ένα χάπι για τον πονοκέφαλο που δεν περιέχει δραστική ουσία, εντάξει, κρίμα, δεν θα περάσει πονοκέφαλος. Αλλά δεν είναι και ευχάριστο να αγοράζω ένα φυτικό προϊόν το οποίο εγώ θεωρώ ότι θα με καθησυχάσει και ανταυτού να με εξάψει. Πάλι εδώ πέρα. Αλλά αν δεν υπάρχει η παρήνη εδώ πέρα, η οποία είναι απαραίτητη σε ορισμένους ανθρώπους για το κυκλοφοριακό, μιλάμε πραγματικά για βλάβες στην υγεία. Και εδώ πέρα στο άρθρο 54α νομίζω μπορεί να κάνει η Κομισιόν κάποιες εξαιρέσεις, ε, όπως π.χ. σε μεγάλες συσκευασίε για νοσοκομεία. Και βεβαίω πρέπει να να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Ελπίζω λοιπόν αύριο να είναι λογική η ψηφοφορία και να είμαστε και ενωμένοι στην Ολομέλεια για να στείλουμε ένα μήνυμα στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Αντωνία Παρβάνοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα παρουσιάσω τη θέση των φιλελευθέρων εξ ονόματος του κυρίου Κράμερ, ο οποίος είναι ακόμα στα αεροπλάνο και επομένω δεν είναι σε θέση να τα παρουσιάσει ο ίδιο ε, και να παραστεί. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρου του. Καταρχά, να ευχαριστήσω τη Μαρίσα Ματία για όλα όσα έχει κάνει για αυτό το τόσο σημαντικό και τόσο δύσκολο θέμα και για το πνεύμα διαλόγου και συνεργασίας που τη διακρίνει. Είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι προσπάθησε να κάνει πάρα πολλά πράγματα με τον ορισμό και νομίζω ότι ο συμβιβασμός είναι ό,τι καλύτερο και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι με την πρόταση αυτή ασχολούμαστε μόνο με το 1% των ψευδεπίγραφων φαρμάκων, ε, τα φάρμακα τα οποία εντάσσονται στην αγορά από την όμιμη αλυσίδα διανομής. Ε, επομένως αυτή είναι μόνο η αρχή. Χρειαζόμαστε πολύ πιο στεναρή δράση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω και να καταπολεμήσουμε την ε, παραποίηση φαρμάκων. Γι' αυτό και με χαροποιεί το γεγονός ότι ασχολούμαστε με τις διαδικτυακές πολίτησεις και κυρίως τις συμβαστικές τροπολογίες 2, 3 και 12 και την κατάλληλη περιγραφή της συμβιβαστική ε, τροπολογίας 12. Εύχομαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει να ενισχύσει το θέμα της τελωνιακής συνεργασίας στον τομέα αυτό, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε πλήρως το θέμα των παραποιημένων φαρμάκων, όπως αναφέρεται και στη συμβαστική τροπολογία 1. Όσον αφορά τώρα την νόμιμη αλυσίδα διανομής, ε, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται βασίζονται στις βασικές αρχές που αναφέρονται στην τροπολογία 279, την αποτελεσματικότητα ω προς το κόστος του συστήματος, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι κάθε φάρμακο που παρέχεται βασίζεται σε σχέση ωφέλου ε, κόστους και επίση θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι διασυνδέεται το κόστος ε, με την τιμολόγηση του προϊόντος κυρίως όταν μιλάμε και για τα generic φάρμακα, τα οποία είναι μεγάλο ποσοστό των φαρμάκων, ε, ε, ε μικρό συγγνώμη, ποσοστό των φαρμάκων που παραποιούνται. Ελπίζω ότι αυτή η προσέγγιση θα υποστηρίζεται για να μπορέσουμε να ε, προχωρήσουμε περαιτέρω το θέμα αυτό προς το συμφέρον της ασφάλειας ε, των ασθενών για τη συμβαστική τροπολογία 9 Χαίρομαι ιδιαίτερα για την προσέγγιση που βασίζεται στον κίνδυνο και τις ε, σχετικές συμβαστικές ε, τροπολογίες, όχι μόνο για τα χενόσιμα φάρμακα όπως σας είπα, αλλά αυτό αφορά και τις ε, ανάλογικές και αποτελεσματικές δράσεις και για την τροπολογία 231 της Dagmar Rothberend και την επανασυσκευασία. Εγώ έκανα μια τροπολογία η οποία ήταν πολύ πιο ισχυρή και συμφωνώ ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε συμβιβαστικά την ε, τροπολογία της κυρίας Ροτμπέρεντ. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι θα γίνεται άμεση επανεσυσκευασία ε, του προϊόντος ε, και κανονικά δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε αυτόν ο οποίος κάνει την επανασυσκευασία να αγγίζει την προστατευτική ε, το προστατευτικό τμήμα του φαρμάκου. Νομίζω ότι η ασφάλεια των ασθενών είναι αυτή η οποία προέχει και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αμήλικτοι στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Στρομαπούλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, είμαστε εμείς μπορούμε να δηλώσουμε εξ αρχής ότι είμαστε ικανοποιημένοι σε γενικές γραμμές και από το πνεύμα της ε, εισηγήτριας και από τη διαδικασία των διαβουλεύσεων με τις άλλες πολιτικές ομάδες και από το περιεχόμενο των περισσότερων συμβαστικών τροπολογιών για το σχέδιο που συζητάμε. Σε μερικές ε, βέβαια ε, τροπολογίες υπήρχαν ε, αποκλήσεις από τις αρχικές μας θέσεις αλλά τελικά τις στηρίζουμε όλες. Και θα ήθελα να αναφερθώ πολύ σύντομα σε τρεις βασικές συμβαστικές τροπολογίες και μόνο σε αυτές γιατί στην ε, κοινωνική σημασία και στην πολιτική ουσία ε, του θέματος α, ε, αναφέρθηκα σε άλλη συνεδρίαση. Αν και αρχικά είχαμε ζητήσει να επεκταθούν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας σε όλα τα φάρμακα, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις παραποίησης μη συνταγογραφούμενων ε, φαρμάκων. Τελικά στηρίζουμε τη συμβαστική πρόταση για επέκταση σε συγκεκριμένα μη συνταγογραφούμενα σε τέσσερα χρόνια στη βάση της ανάλυσης ρίσκου παραποίησης αλλά και κατόπιν ανάλυσης των νέων χαρακτηριστικών ασφαλείας συγκεκριμένων συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Κινούμε τις συμβαστικές τροπολογίες 4, 7 και 15. Επίσης, είμαστε ικανοποιημένοι που οι συμβαστικές ε, τροπολογίες 5 και 8 ακολούθησαν την αρχική μας πρόταση και επιτρέπουν την ανασυσκευασία εφόσον οι ανασυσκευαστές χρησιμοποιούν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Και τέλος, είμαστε επίσης πολύ ικανοποιημένοι που οι συμβαστικές τροπολογίες 3, 4, 12 και 13 συνάδουν με τις αρχικές μας προτάσεις σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση των χαρακτηριστικών ασφαλείας και ειδική άδεια για πωλήσει φαρμάκων μέσω διαδικτύου. Καθώς και για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από την διαδικτυακή πώληση φαρμάκων. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε τελικά ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Thank you, Marina Thank you. Um, first of all, my congratulations. Ευχαριστώ. Θέλω καταρχά να ευχαριστώ τη Μαρίσα την εισηγήτρια. Πολύ καλή έκθεση και πολύ καλή συνεργασία. Μα επέτρεψε να συμμετάσχουμε όλοι στι συζητήσει. Και Βλέπω ότι οι συμβαστικέ τροπολογίε στείλουν προ τη σωστή κατεύθυνση, έχουν δώσει την έμφαση στα κατάλληλα σημεία. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τι εγκρίνουμε και αύριο ίσω με την ψηφοφορία για να έχουμε ακόμη περισσότερη αποτελεσματικότητα την ώρα που θα φτάσουμε στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Χωρί να είναι τέλεια βέβαια, γιατί κάποια σημεία θα ήθελα και εγώ να ε, δουν συμπληρώσει με περισσότερα φάρμακα ή ε, θέματα που έχουν να κάνουν με τις μεγάλες συσκευασίε κτλ. Βλέπω όμως ότι είναι μια έκθεση καλή, θετική, που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι θα πρέπει το θέμα αυτό σε μερικά χρόνια να το ξαναδούμε. Γιατί η απομίμηση αποτελεί ποινικό αδίκημα. Και ξέρουμε ότι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την απομίμηση, οι εγκληματίε, βρίσκουν πάντα έναν τρόπο, ένα παραθυράκι. Και έτσι θα ξαναβρούμε μπροστά μα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα. Εν πάση περιπτώσει πάντω, σαν πρώτο βήμα η οδηγία αυτή μπορεί να προχωρήσει και να τη δώσουμε συνέχεια σε μερικά χρόνια. Ο πρόεδρο. Ο κύριο Λύση έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ και εγώ, ευχαριστώ την εισηγήτρια και, τους, ε, και τις κοιόδης εισηγητές και εισηγήτρες, κυρίως την κυρία Γκρόστατ εκ μέρους του ΕΛΚ. Ξέρω και από τα όσα παρακολούθησα στην υπόθεση αυτή ότι δεν ήταν εύκολο να βρεθούν οι συμβαστικέ λύσει πάντα, αλλά τώρα έχουμε συμφωνήσει όλε οι ομάδε, ιδιαίτερα ω προ το να πάρει το χαρακτήρα των στοιχείων και το ίντερνετ. Οι συμβαστικέ τροπολογίε ήταν πολύ επιτυχημένε. Δυσκολίε βλέπουμε ακόμη ω προ το πώ θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την συνέχιση, την επιβίωση, αν θέλετε, του, παρα... του παράλληλου εμπορίου, χωρί όμω ταυτόχρονα να θέτουμε σε κίνδυνο την ασφάλεια των ε, ασθενών. Και επίσης ένα άλλο ζήτημα είναι αυτό των μεγάλων συσκευασιών. Είπα όμω και η κυρία Ροθβέρον ότι πρέπει να προχωρήσουμε πλέον στην κατάσταση στην οποία αντιμετωπίζουμε τώρα, που δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αγορά για τα φάρμακα. Θα είχε πολύ σοβαρές επιπτώσεις για τον Ευρωπαίο ασθενή το να ε, καταστεί πολύ δύσκολη και αδύνατη η αγορά μέσω του ίντερνετ. Διότι αν είναι πολύ ακριβό το φάρμακο, εάν δεν υπάρχει δυνατότητα του παράλληλου εμπορίου, αν υπάρχει η ε, αν υπάρχουν οι περιορισμοί στην πρόσβαση για τον ασθενή στα φάρμακα αυτά και στι αγορέ μέσω του ίντερνετ, θα έχουμε καταστροφικέ συνέπειε. Πλην όμω πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε ταχύτατα σε μια έκθεση για την ανάπτυξη μιας εσωτερικής αγοράς τις συνέπειες, το κόστος, ε, τα ωφέλη και ενώ το παράλληλο εμπόριο υπάρχει και πρέπει να υπάρχει για να βοηθάει στην ε, μείωση των τιμών, πρέπει και εμείς να είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε την κατάσταση έτσι ώστε να, ε, να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη ασφάλεια για τους ασθενείς μας. Πριν από τέσσερα χρόνια, όταν είχαμε την αναθεώρηση νομοθεσίας για τα φάρμακα, ε, στην Ευρώπη. Είχε γίνει μια προσπάθεια από τον συνάδελφο Μούλερ για ε, συζήτηση και του θέματος των τιμών που η Γερμανία ιδιαίτερα είχε απορρίψει αλλά τώρα βλέπουμε ότι επανέρχεται το θέμα. Με πιο πολύ λοιπόν ενθουσιασμό και αδημονία θα έλεγα μπορούμε να ε, ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Για δε τις τροπολογίες 225 και τη δική μου δηλαδή και της κυρίας Παβάνοβα και άλλων θα ήθελα να σημειώσω ότι μιλούμε για ένα πρώτο βήμα στο οποίο δεν υπάρχουν υποχρεωτικά στοιχεία ασφάλειας, αλλά προσπαθούμε να πείσουμε τον τρόπο αυτό την φαρμακοβιομηχανία ε, εθελοντικά να προχωρήσει στην εισαγωγή των στοιχείων ασφαλείας. Και για την 179, τις ουσίες δηλαδή, θα παρακαλούσα τους συναδέλφους να εξετάσουν με προσοχή και ε, θετικό πνεύμα την ε, τροπολογία αυτή, τη δική μου και του μου, που κοιτάει περισσότερο τη διάκριση των ουσιών, ποιες είναι εκείνες οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν ε, επιβλαβείς, πώς θα πρέπει να διακρίνουμε δηλαδή τις ε, ουσίες, τις ενεργές και τις ωφέλιμες από εκείνες που ενδεχομένως να παρουσιάζουν κίνδυνο. Αυτά ευχαριστώ πολύ και πιστεύω αύριο να γίνει μια καλή ψηφοφορία. Ευχαριστώ Πανιού, Ζήλα. Όχι, δεν θέλετε το λόγο. Μπορώ να συμφωνήσω με όσους είπαν πως βρήκαμε καλές συμβαστικές λύσεις ε, στον ορισμό. Ε, μπει και το εμπόριο του διαδικτύου και στις κυρώσεις ε, που απαιτούνται. Ο Πέτερ Λίζε επίσης έχει δίκιο πως θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το χάος αυτό στην αγορά των φαρμάκων. Το είπε και η Ντάγμαρ. Δεν υπάρχει λόγος για τον οποίο σε μία χώρα έχει 12 χάπια συσκευασία, σε άλλη 10, σε άλλη 36 και δεν ξέρω και εγώ τι. Τώρα το εάν θα έχουμε και τις ίδιες τιμές βέβαια με την ίδια συσκευασία είναι άλλο θέμα. Καλό θα ήταν αλλά υπάρχουν και διαφορετικές ε, κουλτούρες όσον αφορά το κόστος της υγείας. Σωστά επίσης είπε η Ντάγμαρ πως ε, δεν θέλουμε να παραποιούνται φάρμακα ή συστατικά των φαρμάκων. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν είμαι τελείως ε, πεπισμένος για το ότι η ανασυσκευασία είναι η πηγή του προβλήματος, γιατί εκεί πέρα δεν παραποιούνται φάρμακα, εκεί πέρα αλλάζει συσκευασία για να πουληθούν στη χύψη αγορά για το ότι διαφέρει το μέγεθος, και ο λόγος είναι ότι διαφέρει το μέγεθος συσκευασία από χώρα σε χώρα. Το φάρμακο το ίδιο δεν αλλάζει, οπότε δεν ξέρω αν αυτό επιτυγχάνει τον στόχο που θέλουμε. Και νομίζω επιτρέπεται κιόλας, είναι υπερβολικό, επιτρέπεται στην εσωτερική αγορά να χρησιμοποιήσει κανείς αυτά τα πλεονεκτήματα και το παράλληλο εμπόριο επιτρέπεται πλην μιας ε, μόνο περίπτωση. πλην ε, Μεγάλης Βρετανίας. όπου όμως ε, δεν νομίζω ότι ε, αυτή είναι η αιτία εδώ πέρα της παραποίησης. Ο μόνος θα ωφεληθεί είναι η φαρμακευτική βιομηχανία με την ε, επανεισαγωγή των φαρμάκων δηλαδή. Και δεν ξέρω αν τελικά η όλη αυτή η πρακτική οδηγήσει σε μια ρύθμιση του τι πρέπει να κοστίζει το φάρμακο. Οπότε φαίνεται είναι διαφορετικές ε, οι απόψεις. Και δεν ξέρω, κάποιοι εδώ πέρα βλέπουν πράγματα τα οποία δεν, δεν ισχύουν και δεν συμβαίνουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είχα να πούν συνάδελφοι. Αν θέλει να πει κάτι η συγκήτρια, μπορεί να το πει. Όχι. Όχι, όχι, κύριε Πρόεδρε, τίποτα το ιδιαίτερο δεν έχω να προσθέσω. Απλά συμφωνώ με αυτά τα οποία ακούστηκαν για τις παράλληλες αγορές είναι μια πραγματικότητα που υπάρχει στην ε, εσωτερική αγορά και πράγματι το θέμα είναι εδώ πέρα και οι θέσεις εργασίας που συνδέονται με το φαρμακό αλλά πέρα από αυτά δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Αύριο ψηφίζουμε. Οπότε Περνάμε στα σημεία 6 και 7 για την φαρμακοεπαγρύπνηση και εκεί πέρα η συγγήτρια είναι η Λίνα Μακάβαν η οποία έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα τα δούμε αυτά τα δύο θέματα μαζί. Συνάδελφοι, μοιράσουμε τώρα τις ε, συμβαστικές τροπολογίες που στις οποίες συμφώνησαν οι περισσότεροι σκιώδεις ηγητές των ομάδων. Δεν, ε, έχει όμως, δεν είχε το χρόνο η γραμματεία να κάνει το σχετικό έγγραφο να σου πει ποιοι συμφωνούμε πια, οπότε θα σας τα πω. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τους Ήταν δύσκολη η προηγούμενη εβδομάδα, πολλοί δεν μπορέσαμε να πάμε στο Στρασβούργο και ξέρω πως εργάστηκαν σκληρά για να συμφωνήσουμε στις συμβαστικές τροπολογίες κατά το οποίο θα μας επιτρέψει να έχουμε μια απλή ψηφοφορία αύριο στην Επιτροπή μας. Η γενική αξιολόγηση που θα έκανα εγώ για το τι θα ψηφίσουμε αύριο είναι πως θα βελτιώσουμε το σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης στην Ευρώπη και όπως και με την παραποίηση μιλάμε εδώ πέρα για την ασφάλεια των ασθενών για την τήρηση των κανόνων, για την πληροφόρηση των ασθενών εάν τα φάρμακα είναι νέα ή περιέχουν νέες δραστικές ουσίες, για να αναφέρουν τυχόν παρενέργειες στις αρχές και οι αρχές μετά μαζί με τις φαρμακευτικές εταιρείες να δουν και να δώσουν μια συνέχεια στις παρενέργειες για να δούνε αν πρέπει να γίνει τίποτα άλλο ή να δοθεί κάποια συμβουλή στους ασθενείς. Αυτό το οποίο θα έχουμε λοιπόν ως αποτέλεσμα είναι η βελτίωση της ασφάλειας ε, των ασθενών. Εάν δούμε τώρα τις συμβαστικές τροπολογίες στην οδηγία η 1α και η 1β, όπως ε, είναι η αριθμίση αυτή τη στιγμή, αναφέρονται σε βελτιώσεις στα φυλάδια πληροφόρησης των ασθενών. Στην τελευταία συζήτησή μας κατέστη σαφές πως δεν υποστήριζαν οι συνάδελφοι την πρόταση της Κομισιόν για να μπει μια κατηγορία στο φυλάδιο που θα λέγεται ουσιαστικές πληροφορίες. Δηλαδή η Κομισιόν λέει πως ε, είναι αρκετά λεπτομερές στο φυλάδιο, οπότε να βάλουμε με παχιά γράμματα τα βασικά. Αλλά δεν το υποστήριξαν αυτό οι ομάδες των ασθενών, γιατί αυτό το οποίο είναι κέριο για τον έναν δεν είναι σημαντικό για τον άλλον. Οπότε αυτό το οποίο προτείνουν όλοι οι σκιώδεις ηγητές είναι να ζητήσουμε από την Κομισιόν να ξαναδεί τα φυλάδια ε, πληροφόρηση των ασθενών ε, από την αρχή και προτείνουμε αυτό να γίνει εντός 18 μηνών και οι οργανώσεις των ασθενών και των καταναλωτών, οι επαγγελματίες υγείας να εκφραστούν όλοι. Αυτό για το 1α και το 1β. Δεύτερη ομάδα τροπολογιών 2α και 2β καλύπτουν μία άλλη ομάδα προϊόντων και εδώ πέρα είχαν πάρα πολύ συζήτηση, τα αποδέχονται όλοι όλες οι πολιτικές ομάδες πλην των πρασίνων. Ένα αρκετά επίμαχο ζήτημα ήταν πώς θα πρέπει να ονομάσουμε αυτά τα φάρμακα. Είναι φάρμακα τα οποία είτε είναι νέα στην αγορά ή περιέχουν δραστικές ουσίες και το σκεπτικό είναι να ενημερώνουμε τους ασθενείς πώς ε, παίρνουν νέα φάρμακα και να προσέχουν για παρενέργειες. Πρώτο ζήτημα λοιπόν είναι πώ θα τα πούμε αυτά τα νέα φάρμακα. Και πάλι αφού μίλησα με τους συναδέλφους, φαίνεται πως δεν είμαστε υπέρ ε, της ε, πρώτας κομισιόν που μιλάει για προϊόντα υπό αυστηρή επιτήρηση. Οπότε προτείνουμε στο φυλάδιο να συμπεριληφθεί ο όρος το φάρμακο αυτό υπόκειται σε επιπλέον επιτήρηση ασφαλείας και να υπάρχει και ένα σύμβολο το οποίο θα γίνει γνωστό και θα σημαίνει πως ε, το φάρμακο αυτό είναι καινούριο ή έχει καινούρια και δραστική ουσία. Οπότε ήταν μεγάλη συζήτηση για το σύμβολο αυτό. Ένα ανάποδο τρίγωνο χρησιμοποιείται ήδη από τους επαγγελματίε, αλλά δεν άρεσε σε κάποιους συναδέλφους καθώς σε κάποιες χώρες σημαίνει κίνδυνος ή δηλητήριο οπότε αναθέσαμε στην Κομισιόν να βρει ένα σύμβολο. Και πάλι συμφωνήσαμε πως θα πρέπει να είναι μαύρο το σύμβολο και απλό. Κάποιοι συνάδελφοι ήθελαν να είναι και στην εξωτερική συσκευασία και στο φυλάδιο αυτό, αλλά δεν υπήρχε συνένεση μεταξύ των σκιωδών. Οπότε προς στιγμή το αφήνουμε στο φυλάδιο. Και τα ίδια ισχύουν και για την 2Β. Εγώ προσωπικά δεν είχα πρόβλημα με την ιδέα των προϊόντων υπό αυστηρή επιτήρηση, αλλά βλέπω πως δεν υπήρχε συνένεση. Και αφού μίλησα με την Κομισιόν, νομίζω πως το βασικό είναι ότι οι ασθενείς πρέπει να ξέρουν ότι, οι ασθενείς πρέπει να ξέρουν ότι παίρνουν ένα καινούριο φάρμακο ή φάρμακο με νέα δραστική ουσία, οπότε πρέπει να αναφέρουν τυχόν ζητήματα. Οι δύο γαμανέ, ναι. Όλες αυτές ε, που ξεκινάνε με δύο καλύπτουν το ίδιο ζήτημα. Η υπαριθμόν 3 αναφορά από τους ασθενείς ε, την έχουν υπογράψει όλες οι πολιτικές ομάδες και οι περισσότερες τοπολογίες λένε πως το να λέμε ότι ο ασθενής ε, θα πρέπει να μπορεί να δίνει αναφορά μέσω ίντερνετ φτάνει, θα μπορούν να χρησιμοποιούν και τηλέφωνο ή γράμματα ή τέτοιες, απλές δηλαδή τροπολογίες. Και μετά βελτίωση στο ποιε πληροφορίες δίνονται στο κοινό μέσω της δικτυακής πύλης και τέλος προσθέτουμε κάτι για, για τα φάρμακα για τα οποία δεν θα πρέπει να υπάρχει ε, καταλογισμός ευθύνης γιατί εάν είναι να αναφέρονται αυτά θα πρέπει πράγματι μετά να μην κατηγορείται κανείς αλλά συμφωνήσαμε να φύγει το η ιδέα εδώ πέρα της ανώνυμης ε, καταγγελίας γιατί είχαμε περιπτώσεις ε, κακοήθους ε, αναφοράς από τους ανταγωνιστές. Οπότε προτείνουμε να μην είναι ανώνυμο και νομίζω σωστό είναι. Και για να υπάρχει και σωστή παρακολούθηση άλλωστε πρέπει να μπορούμε να ερχόμαστε σε επαφή μετά με το άτομο. Αυτά με την τρία. Συμβαστική λύση. Τέσσερα είναι η πιο οι τέσσερα πιο επίμαχες, ε, αφορούν τις επιδράσεις στο περιβάλλον. Την τελευταία φορά που το συζητήσαμε, εγώ δεν ήθελα στην ομοθεσία εδώ πέρα να μπουν διατάξεις που απαιτούν από τις αρχές που ασχολούνται με τη φαρμακοεπαγρύπνηση να έχουν και αρμοδιότητες περιβαλλοντικές. Που είναι σημαντικό ζήτημα, αλλά δεν ε, αφορά η φαρμακοεπαγρύπνηση ή αφορά την ανθρώπινη υγεία. Τώρα έχουμε δύο συμβαστικές ε, τροπολογίες. Η μία έχουμε το 5α νέο, το εκτιμώντας και άλλη μία αφορά το άρθρο. Η πρώτη που αφορά το εκτιμώντας έχει υπογραφεί από όλες τις ομάδες πλην του ΕΛΚ και η ενοποιημένη τροπολογία για το άρθρο για το διατακτικό υπογράφτηκε από τους σοσιαλιστές τους πράσινους και την ΚΟΕ. Νομίζω οι περισσότεροι συμφωνούν πως κάτι πρέπει να γίνει για το περιβάλλον. Μίλησα με την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Υπάρχει επιθυμία να δούμε το όλο ζήτημα του περιβαλλοντικού αντικτύπου των φαρμάκων, χωρίς όμως να, να βλάψουμε την ανθρώπινη υγεία. Πρέπει να το καταλάβουμε. Κάποια φάρμακα και όταν έχουν επίδραση στο περιβάλλον ε, υπερισχύει ανθρώπινη υγεία σε κάποιες περιπτώσεις. Μετά, συμβαστική λύση 5 για τους κινδύνους και τα ωφέλη νομίζω είναι αυτεξήγητο. Δηλαδή μελέτες μετά την αδειοδότηση γίνονται από τις εταιρείε όταν το ζητούν οι αρχές. Υπήρχε πρόβλημα στο παρελθόν καθώς όταν δίνονταν άδεια δεν έγιναν μετά όλες αυτές οι μελέτες. Οπότε έχει αυτή εδώ πέρα μια νέα έννοια για τις μελέτες αποτελεσματικότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, μετά από συζητήσεις με τους συναδέλφους και την Κομισιόν για το θέμα του όταν ένα φάρμακο είναι στην αγορά επί πολλά χρόνια, στη φάση της αδειοδότησης πρέπει να αποδεικνύεται και αποτελεσματικότητα αλλά μετά από χρόνια δεν χρειάζεται να επανεξεταστεί. Οπότε το συμπεριλάβουμε αυτό εδώ πέρα για να καλύψουμε κάποιους συναδέλφους. Κάποιοι συναδελφοί ήθελαν τα φάρμακα να μπορούν να διατεθούν εάν ανταποκρίνονται σε κάποια ιατρική ανάγκη. Δεν συμφωνώ. Γνωρίζουμε πως κάποιες ασθένειες ε, κινούνται σε ένα φάσμα και κάποιοι αντιδρούν διαφορετικά στο ένα φάρμακο από ό,τι στο άλλο. Το ότι υπάρχει ένα φάρμακο δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκλείσουμε ένα άλλο. Αλλά υπάρχει η προσθέμενη αξία του φαρμάκου. Πρέπει πράγματα να προσφέρουν κάτι στον ασθενή που τα παίρνει. Οπότε έχουμε εδώ πέρα μια συμβαστική τροπολογία που χρειάστηκε πάρα πολύ κόπο και ευχαριστώ τους συναδέλφους και ελπίζω να αποτελέσει βάση συζητήσεων στο Συμβούλιο για το σοβαρό αυτό ζήτημα η έξι για τα τέλη, κανένα πρόβλημα, την υπέγραψαν όλες οι ομάδες. Θέλουμε να διασφαλίσουμε πως υπάρχει εγγύηση της ανεξαρτησίας φαρμακοεπαγρύπνησης. Και τέλος η 7 για τη δικτυακή πύλη αφορά το ποιες πληροφορίες πρέπει να είναι δημόσιες και πρώτα απ' όλα ευχαριστώ την Κομισιόν που ήθελε όλο το σύστημα της φαρμακοεπαγρύπνησης στην Ευρώπη να γίνει πολύ πιο διαφανές είναι πιο διαφανές ε, από ό,τι της ε, είπα. Έχουμε υποβάλει σχετικές τροπολογίες και εγώ προτείνω να μην υποστηρίξουμε τροπολογίες που θα περιορίσουν τις πληροφορίες. Οι άλλες πέντε τροπολογίες ε, αφορούν την επιτροπολογία. Κατατέθηκαν μετά από πρόταση της γραμματείας γιατί είχε συνταχθεί το νομοθέτημα πριν από την ε, συνθήκη της Λισαβόνας, οπότε είχαμε και τις ε, σχετικές αλλαγές. Περνάμε στον κανονισμό. Σημείο 1. Κανένα πρόβλημα. Τα προϊόντα με εντονή επιτήρηση το υπέγραψαν όλοι πριν πρασίνων και εδώ πέρα το θέμα αφορά το όνομα. Και πάλι χρησιμοποιήσαμε τον όρο επιπλέον παρακολούθηση. Συμβαστική τροπολογία για το περιβάλλον. Μόλις μου είπαν να διορθώσω αυτό το οποίο είπα πριν. Το ΕΛΚ έχει υπογράψει τη συμβαστική τροπολογία για τα εκτιμώντας, οπότε έχουν υπογράψει όλες οι ομάδες. Αλλά για το διατακτικό ήταν σοσιαλιστές, πράσινοι και γκουε. Μετά συμβαστική τροπολογία 3 το ίδιο, τέλη το ίδιο, διαδικτυακή πύλη το ίδιο. Ε, παρόμοιο ζήτημα και στον κανονισμό πρόσβαση εδώ πέρα στην ε, συμβαστική τροπολογία 6 και αυτό το έχουν υπογράψει όλες οι ομάδες, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά να διευκρινίσω το εξή γιατί κάποιοι συνάδελφοι, όχι ισχυώδεις ηγητές, που δεν το είχαν παρακολουθήσει τόσο στενά, έχουν μπερδευτεί λίγο η διαδικτυακή πύλη, είναι το site ε, όπου υπάρχουν οι πληροφορίες για το κοινό. Η βάση δεδομένων όμως είναι για τους ειδικού. Και εκεί πέρα συμπεριλαμβάνονται οι παρενέργειες ε, και οι, ειδικοί, οι εθνικές αρχές δηλαδή και οι εταιρείε μοιράζονται τα δεδομένα τους. Πτυχές αυτής της βάσης δεδομένων, κάποια κομμάτια είναι δημόσια και θέλουμε να είναι όσο δυνατόν πιο διαφανής, αλλά βεβαίως ε, οι λεπτομέρειες ε, συγκεκριμένων ατόμων ε, βεβαίως δεν θα γίνουν γνωστές. Αυτές είναι λοιπόν οι συμβαστικές τροπολογίες, όπως είπα οι περισσότερες έχουν υπογραφεί από όλες τις ομάδες και ελπίζω αύριο το πρωί να πάει καλά η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. You, Ευχαριστώ Λίντα. Και για όλη τη δουλειά βέβαια που έχεις κάνει μέχρι τώρα για μας για τα δύο αυτά νομοθετήματα, για τις συμβαστικές λύσεις που έχει εξασφαλίσει. Η Πιλαραγιούσο τώρα για να ακούσουμε και τους κοιόδης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω ειλικρινά την κυρία Μακάβαν για την ε, πάρα πολλή δουλειά που έκανε προκειμένου να καταλήξει στους συμβιβασμούς ο οποίο επέτυχε και εμείς τους υποστηρίζουμε ουσιαστικά όλους και να ευχαριστήσω και τους κοιόδης εισηγητές ε, και τους ε, βοηθούς μας οι οποίοι χρειάστηκε να εργαστούν πάρα πολύ σκληρά και καταλαβαίνετε και ότι με όλα τα προβλήματα που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και οι περισσότεροι από εμά δεν μπορούσαμε να παραστούμε στο Στρασβούργο, η βοήθειά του ήταν πολύτιμη. Οι συμβαστικέ προτάσει ε, περιλαμβάνουν τα πιο σημαντικά και πιο δύσκολα σημεία που συζητήθηκαν. Πρόκειται για μια οδηγία και ένα κανονισμό που θέλουν ο ασθενής να γνωρίζει καλά και να είναι καλά ενημερωμένος ε, για τις ε, συνέπειες και τις παρενέργειες που μπορεί να έχει ένα φάρμακο και τι άγουσα μπορεί να ακολουθήσει προκειμένου να κοινοποιήσει το πρόβλημα που διαπιστώνει είτε σε μια ιστοσελίδα, είτε στο γιατρό του, είτε σε κάποιον αρμόδιο σε θέματα υγείας και θεωρώ ότι αυτέ οι τροπολογίε βελτιώνουν κατά πολύ την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα υποστηρίξουμε τι τροπολογιε 1 1α, 2α, 2b, 4α, 5, 6 και 7. Η κυρία Βακάβαν εξήγησε πάρα πολύ καλά κάθε μία από τι τροπολογίε. Επομένω, εγώ δεν θα ε, σπαταλήσω το χρόνο σας αναφέροντας τις ε, ε, τροπολογίες. Ε, όσον αφορά τώρα αυτό το ενδεικτικό τρίγωνο για τα φάρμακα, εγώ είπα εχθές ότι συμφωνούσα με αυτό το τρίγωνο, αλλά διαπίστωσα ότι υπάρχουν κάποιες χώρες ότι για αυτές ε, που για αυτές σημαίνει ότι μπορεί να είναι τοξικό το προϊόν. Καλό θα ήταν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το μελετήσει και σε 18 μήνες να μας προτείνει ένα άλλο σύμβολο και το ίδιο ισχύει και με αυτό που θα πρέπει να κάνουν για το ε, φυλάδι οδηγιών του φαρμάκου. Ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει στις βασικές τροπολογίες είναι το θέμα του περιβάλλοντος. Συμφωνούμε όλοι ότι είναι πολύ σημαντικό μεν, αλλά θεωρούμε ότι η οδηγία αυτή αναφέρεται στις παρενέργειες που μπορεί να έχει ένα φάρμακο. Και είναι αλήθεια ότι ένα φάρμακο μπορεί να έχει και κάποιε αρνητικέ επιπτώσει για το περιβάλλον, αλλά ένα φάρμακο είναι πάρα πολλά πράγματα. Καλό θα ήταν λοιπόν να αναφέρεται μεν ε, το θέμα του περιβάλλοντο σαν εκτιμώντα, αλλά όχι στο διατακτικό. Γι' αυτό ακριβώ και εγκρίνουμε την 4α και όχι την 4β τροπολογία. Όσον αφορά στον κανονισμό τώρα, το ίδιο ακριβώς ε, υποστηρίζουμε όλες τις συμβαστικές τροπολογίες πέραν της ε, λεπτομέρειας της τροπολογίας για το περιβάλλον. Θέλουμε και πάλι να μην συμπεριληφθεί στο διατακτικό αυτό παρά μόνο σε ένα Ευχαριστώ πολύ. Ε. Ευχαριστώ πολύ, πλέον. Αντώνη Παβάνοβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τη Λίντα για τα θέματα αυτά που έχει επεξεργαστεί. Έκανε μια εξαίρετη δουλειά. Και μια και την προηγούμενη εβδομάδα μας δυσκόλεψε η έκρηξη του ηφαιστείου, νομίζω ότι στηριχθήκαμε σε μεγάλο βαθμό στην επικοινωνία μέσω του ίντερνετ για να καταλήξουμε σε αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες, αυτό μπορούμε να μετακινηθούμε. Θα συμφωνήσω λοιπόν με τις προσθέσεις συμβαστικές τροπολογίες και τα κύρια θέματα της έκθεσης. Ασφάλεια κυρίως, διαφάνεια, εμπιστοσύνη του ασθενούς. Είναι τα κύρια στοιχεία που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι φορείς, οι υπηρεσίες, οι ευρωπαϊκές αρχές ε, και στα μέτρα τα οποία θα καταγράφονται στο ενημερωτικό φυλάδιο, πρέπει να ε, είναι σαφή. Λέμε ότι τα μέτρα έχουν μεγάλη σημασία και για το φάρμακο, αλλά για τον ασθενή πάνω απ' όλα. Και ζητούμε από την όλων των ομάδων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει μια πρόταση ώστε να βελτιωθεί η αναγνωσιμότητα, η παρουσίαση στο φυλάδιο, γενικά η δυνατότητα κατανόησης το ευανάγνωστον αυτού του φυλαδίου που απευθύνεται στον ασθενή. για τα προϊόντα και την εντατική παρακολούθηση. Βλέπαμε χαρά ότι μπορέσαμε να αποφύγουμε την εντατική παρακολούθηση για να βρούμε μια καταλληλότερη διατύπωση προϊόν δηλαδή και πρόσθετη ε, παρακολούθηση ασφαλείας ή επιτήρηση ασφαλείας. Νομίζω ότι αυτό είναι καταλληλότερο ως διατύπωση και για τα φάρμακα και για την φαρμακοβιομηχανία ως λύση. Οι επιπτώσεις των φαρμακευτικών ε, προϊόντων με το 1α, 1β και με τα 2α, 2β για την ενημέρωση στα παραρτήματα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε απλοί και ρεαλιστές σε κάθε τομέα πολιτικής. Είναι απαραίτητο οι συζητήσεις μας να στηρίζονται σε στοιχεία, σε τεκμήρια. Εδώ δυστυχώ και βλέπω ήδη από τη λειτουργική σκέψη ότι κάνουμε κάποιε δηλώσει περιβαλλοντικών προβλημάτων, διακηρύξει, αν θέλετε για τι ανησυχίε μα για το περιβάλλον, για τι εκτό των περιβάλλων που όμω δεν στηρίζονται στη στοιχεία. Το να κατηγορούμε λοιπόν τα φάρμακα ανθρώπινη χρήση για την ρήπανση ή επιδείνωση τη ρήπανση του περιβάλλοντο, είναι νομίζω μια τοποθέτηση μάλλον εφάνταστη όταν δεν υπάρχουν δεδομένα και στοιχεία. Εμείς όμως, όμως κοινοβούλιο πρέπει να είμαστε πολύ υπεύθυνοι, σοβαροί και να, δίνουμε τις, να κάνουμε τις επιλογές μας στηριγμένοι σε στοιχεία. Δεν ε, κάνουμε αρθράκια για, τα, για τις εφημερίδες και το τύπο γενικά. Πρέπει να έχουμε στοιχεία στα όσα λέμε. Και γι' αυτό θα ήθελα και η Επιτροπή να μας δώσει τα δεδομένα που έχει στη θέσή της. Εάν αποδεικνύεται επιδείνωση του περιβάλλοντος, ρήπανση κτλ. Να ξέρουμε πώς θα την προσμετρήσουμε και, την, και πού ακριβώς. Θα είναι άλλωστε κάτι το πολύ δαπανηρό αυτή η μέτρηση. Και έστω ότι απεδείχθη ρήπανση, θα απαγορεύσουμε την κυκλοφορία των φαρμάκων αυτών. Ιδιαιτέρως ορισμένων, το, τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν άκρος επικίνδυνα, αλλά έχουν πολύ περιορισμένη ε, διάδοση, γιατί μόνο ορισμένοι ασθενεί, ορισμένε κατηγορίε ασθενών δηλαδή τα παίρνουν. Ή τα άλλα τα οποία, ε, όντα λιγότερο επικίνδυνα, έχουν πολύ ευρία διάδοση. Και άρα ω εκ του όγκου του μπορεί να επηρεάζουν το περιβάλλον. Φερρυπίν, γυναικείε ορμόνε και ούτω καθεξής. Ή φάρμακα για καρδιακές παθήσεις. Πώς θα τα κρίνουμε όλα αυτά. Εγώ υποστηρίζω την ε, προσέγγιση της εισηγήτριας γενικότερα με την προφορική ε, καταγραφή, με την δυνατότητα ο ασθενής να δηλώνει κάποιες παρενέργειες που έχει ενδεχομένως επισημάνει. Συμβαστική τρία της οδηγίας, κρίσιμη σημασία. Άλλωστε πολλές ήταν οι οργανώσεις των ε, ασθενών που μας έχουν ζητήσει να δραστηριοποιηθούμε προς το στόχο αυτών για την κοινοποίηση και την ενημέρωση, για την αδειοδότηση, έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να ενημερωθούν εγκαίρως και να είναι σε θέση να αντιδράσουν εγκαίρως. Βεβαίως οι αδειούχοι ενημερώνονται εγκαίρως για τη χορήγηση της άδεια και για ενδεχόμενες ε, παρενέργειες θα ενημερώνονται από τις αρμόδιες αρχές ή από τους ασθενείς. Σε περίπτωση ε, σοβαρών παρενεργειών και άμεσων παρενεργειών θα πρέπει να υπάρχει ένα πιο ταχύ σύστημα αντίδρασης. Ιδιαίτερος θα ήθελα τώρα να συγχαρώ την εισηγήτρια γιατί θα πρέπει εδώ να κάνουμε διάκριση μεταξύ αποτελεσματικότητας και κλινικών αποτελεσμάτων. Υπάρχει διαφορά εδώ. Είναι ένα δύσκολο θέμα, αλλά το συζητήσαμε με όλους τους σκιοδησηγητές και ευχαριστώ πολύ την συγκέντρια που έλαβε υπόψη και τις θέσεις μας. Ευχαριστώ και την Επιτροπή. Βλέπαμε χαρά ότι καταλήγουμε σε συμβαστική λύση ως προς τις αρχές οι οποίες θα αναλαμβάνουν τέτοιου είδου μελέτες, θα είναι σε θέση μάλλον να θέσουν τέτοιες μελέτες ε, για φάρμακα όπου υπάρχει η δυνατότητα της παρακολούθησης εξέλιξης μιας νόσου ή πρόσθετα στοιχεία ενδεχομένως. Η έλλειψη αποτελεσματικότητα η έλλειψη κλινικών αποτελεσμάτων θα μπορούσε να θέσει κίνδυνο τη ζωή του ασθενού, γι' αυτό πρέπει να τη χειριστούμε μεγάλη προσοχή και πρέπει να έχουμε και καλύτερη αξιολόγηση των κλινικών αποτελεσμάτων. Εδώ, από τη Γενική Διεύθυνση υγεία και Προστασία του Καταναλωτού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής, βλέπω μια καινοτόμο προσέγγιση. Βλέπω δυναμικού ανθρώπου προσωπικού αποφασισμένο να λάβει καινοτόμε αποφάσει για τις ευθύνες, για τη φαρμακοεπαγρύπνηση, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο προτείνεται η συνεργασία. Θα πρέπει βέβαια η, αρμόδια, η αρχή CHMP, η Ευρωπαϊκή Αρχή, να παραμένει το αρμόδιο όργανο για την αδειοδότηση Επίσης η προσέγγιση των ΗΠΑ με το FTA αναφέρεται μέσα στο κείμενο και αυτό νομίζω αποτελεί μια καλή εξέλιξη έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη και ασφάλεια για τον καταναλωτή και διαφάνεια. Για την φαρμακοεπαγρύπνηση μπορούμε να έχουμε νομίζω μια προσέγγιση αδειοδότησης για τους ερευνητές διαφορετική, για τα ερευνητικά κέντρα διαφορετική, ώστε να μην κινδυνεύει ο ασθενής, το ευρύ κοινό δηλαδή, ε, να ε, παραπληροφορηθεί και να ε, έχει σφαρμένες πληροφορίες στη θέση του. Ε, Μαρίνα... Ευχαριστώ κύριε Γιανακουδάκη, έχει το λόγο. Uh, yes, I haven't really got more. Έχω δεν έχω και πολλά να πω. Καταρχάς, ε, συγχαρητήρια στη Λίντα. Έκανε πολύ καλή δουλειά και για την πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των ε, όσων συμμετείχαν στο συμβιβασμό. Νομίζω ότι ε, φαίνεται ότι αυτό είναι υπερκομματικό προς όφελος των πολιτών. Υπάρχουν δύο τομείς οι οποίοι μας ανησύχησαν, αλλά ασχοληθήκαμε με αυτούς ε, και το αντιμετωπίσαμε. Κυρίω μας ενδιαφέρει ε, η προστασία των ασθενών. Μας ανησυχούσε η φράση intensive monitoring, αλλά ευτυχώ τη διαγράψαμε αυτό, διότι θεωρούσα ότι θα μπορούσε να αποτρέπει τους ανθρώπους από το να χρησιμοποιούν ε, τα φάρμακα και υπάρχει διαφορά μεταξύ το να προειδοποιούμε τους ασθενείς και να τους τρομοκρατούμε. η αναφορά στο περιβάλλον. Με ανησύχησε λίγο αυτό. Το περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό θέμα, αλλά δεν θα πρέπει να επιβαρύνουμε την οδηγία και τον κανονισμό ε, προσθέτοντας στοιχεία ε, τα οποία δεν, υπάρχουν, δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Ε, βάζοντας το σαν εκτιμώντας, θεωρώ ότι επισημαίνουμε ότι είναι σημαντικό, αλλά δεν θα πρέπει να χάνουμε το στόχο μας. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι είναι ένα καλό κείμενο και θα πρέπει να υποστηρίξουμε το κείμενο αυτό και την οδηγία και τον κανονισμό. Ευχαριστώ, Πέτερ Λίζε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερως και την συγγήτρια και τους και τους συγγητές. Την κυρία Ιούσου ιδιαίτερως από εμά από το ΕΛΚΑ. Θα πρέπει να πω ότι δεν είμαι τόσο ενθουσιασμένος από τις συμβαστικές τροπολογίες όπως την έκθεση Ματίας. Έχω κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Πάντως αποτελεί μια καλή βάση η έκθεση. Με δυστεριστεί κάπως το γεγονός ότι σε αυτή την νομοθετική διαδικασία δεν μπορέσαμε να βελτιώσουμε τις προτάσεις ουσιαστικά. Και ύστερα από 1,5 χρόνο συστήσεις μέσα στην Επιτροπή μας, περίμενα ότι θα μπορούσαμε, αν όχι να κάνουμε την ραγδαία αλλαγή, πάντως κάποιες βελτιώσεις να επιφέρουμε. Αλλά φαίνεται ότι ήταν δύσκολος ο αγώνας, ε, καθώς και κάποιες από τις προτάσεις της Επιτροπής οδήγησαν σε ε, παρερμηνίε και προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, και εγώ έκανα τι δικέ μου προτάσει ε, τροπολογιών. Δεν είχα το χρόνο να τις συζητήσω όμω με του συναδέλφου, όπω θα ήθελα. Εν πάση περιπτώσει για την ενημέρωση όμω των ε, ασθενών παρακαλώ να επανέλθουμε και να έχουμε την ευκαιρία να προσφέρουμε τι ιδέε μα για να βελτιώσουμε αυτή τη δέσμη μέτρων. Γιατί πιστεύω ότι χωρί μια συνοπτική αναφορά δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε το «Είναι ανάγκη για ενημέρωση του ασθενούς. Γιατί βεβαίως πρέπει να είναι πολύ αναλυτικό το φυλάδιο ενημέρωσης για λόγους νομικούς και άλλους κτλ. Αλλά δεν ε, οδηγεί σε ουσιαστική ενημέρωση του ε, απλού πολίτη που δεν είναι ενήμερος για τα ιατρικά. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε κάποιο είδους σύντομη ενημέρωση με επαρκή ε, στοιχεία και με παραπομπές ενδεχομένω αν θέλει να μελετήσει περισσότερο. Βέβαια, σε αυτό θα επανέλθω αργότερα. Ω προ το περιβάλλον και τι επιπτώσει στο περιβάλλον, τόσο μέσα στην Επιτροπή όσο και στην ομάδα μα, εκφράζονται διαφορετικέ θέσει αντιφέμενε. Έχω καταθέσει και εγώ τι προτάσει μου, οι οποίε χωρί να έχουν συμπεριληφθεί κατά λέξη στι συμβαστικέ τροπολογίε, έχουν κάπως γίνει αποδεκτές. αποδεκτές. Δεν θέλω να πω το εξή ότι ναι, έχουμε προχωρήσει ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο περιβάλλον, όχι όσο θα θέλαμε, αλλά πάντως αναγνωρίστε το πρόβλημα και παραδείγματι αν, αν ασχοληθούμε με τις αλλαγές στα αλλιευτικά αποθέματα, μπορούμε να υποθέσουμε τι ίδιους αλλαγές γενετικές μπορεί να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος σε μερικά χρόνια, ο άνθρωπος ο οποίος καταναλώνει τα πόσιμα ύδατα μέσα στα οποία ε, κολυμπούν τα ψάρια. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το μας απασχολήσει ουσιαστικά. Και αυτόχρονα θα πρέπει να δούμε τους όρους υπό τους οποίους ενδεχομένως θα αποσύρεται από την αγορά ένα φάρμακο. Ένα φάρμακο δηλαδή θα πρέπει να αποσύρεται από την αγορά με μόνο γνώμονα τον κίνδυνο για το περιβάλλον. Θα πρέπει να δούμε και αν χρειάζεται ως φάρμακο για συγκεκριμένε ασθένειες. Χρειάζεται λοιπόν η έρευνα πάνω απ' όλα. Και όλοι να κοιτάξουμε προσεκτικά τα επόμενα βήματα. και στην αιτιολογική σκέψη και ενδεχομένω στο διατακτικό θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιε αλλαγέ. Θα δούμε αύριο που θα καταλήξει όλο με την ψηφοφορία. Ω προ την ε, απευθεία αναφορά προ τι αρχέ ενό ασθενού για τι παρενέργειε κτλ. Πάλι έχω πολλέ δυσκολίε. Νομίζω ότι ε, μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα, σε μπέρδεμα μεγαλύτερο από ότι λύσει. Περισσότερα προβλήματα λοιπόν παρά όφελο. Και ίσω ήταν καλό οι συνάδελφοι να επανεξετάσουν τροπολογία 231. Αν είναι δυνατόν να την κάνουν δεκτή, διότι έτσι επιτρέπει περισσότερη ευελιξία στην υπόθεση αυτή. Και παρακαλώ να ρίξουν άλλη μία ματιά στην 246 και 247, αν μπορούν να τις υποστηρίξουν. Πρόκειται για φάρμακα, για δραστικές ουσίες γνωστές, διαδεδομένες, που θα μπορούσε να διευκολυνθεί η αδειοδότησή τους. Για δε τις 276 και 279 ως προς την αδειοδότηση βλέπω ότι οι διεθνώς αναγνωρισμένες οι διεθνώς αναγνωρισμένοι ορισμοί ε, των ε, παρενεργειών ε, πρέπει να γίνονται δεκτοί. Δεν πρέπει δηλαδή να αποκλίνουμε από αυτούς. δε δεύτερη τροπολογία 280 η επιχείρηση, αυτό ισχύει πάνω πολλά, για, έχει μάλλον σημασία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μαγευτικές επιχειρήσεις, πρέπει να είναι σε θέση να ασκήσει ε, προσφυγή κατά μιας απόφασης Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φαρμάκων. Τώρα η δυνατότητα αυτή δεν είναι τόσο δεδομένη, αρκετά περίπλοκη για μια μικρομεσαία επιχειρήση, θα πρέπει να την απλουστεύσουμε. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Ναι, χωρίς να είμαι απόλυτο ικανοποιημένο, βλέπω ότι οι τροπολογίες τίνουν προς την ορθή κατεύθυνση και μπορώ να τι υποστηρίξω. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λεπάζ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Η κυρία Μακέουαν έκανε πολύ καλή δουλειά. Μακάβαν έκανε πολύ καλή δουλειά. Προσπάθησε για τις συμβαστικές τροπολογίες που θα μας έβρισκαν όλους σύμφωνους εγώ προσωπικώς είχα καταθέσει αρκετές δικές μου τροπολογίες. Οφείλω να πω όμως ότι είμαι απόλυτο ικανοποιημένη από τις συμβαστικές τροπολογίες της κυρίας Μακεών. Και για τη διαφάνεια και για τα τέλη. Δύο λόγια μόνο θα ήθελα να πω ότι το περιβάλλον και οι επιπτώσεις ε, στο περιβάλλον των φαρμακευτικών ε, προϊόντων μόνο μέσα από αιτιολογική σκέψη εξετάζονται, αλλά είναι σαφές ότι πρέπει το θέμα αυτό να τεθεί στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων, πρέπει να τεθεί επιτάπητος και ιδιαίτερα σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη ρήπανση των υδάτων, με τα συστήματα καθαρισμού υδάτων, βλέπουμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα βρούμε μπροστά μας. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις, ε, ε, με την αντίσταση πλέον στα αντιβιωτικά που είναι δεδομένη ή με το γεγονός ότι οι αντικαρκυνικές ουσίες ε, ρέουν απρόσκοπτα μέσα στα νερά των ποταμών μας. Είναι ένα θέμα λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να ε, εξετάσουμε. Όχι τώρα, αλλά κάποια στιγμή. Κύριε Στρεμόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα πω δύο λόγια, αν και σαν το report ήταν ε, η κυρία Ριβασί. Δεν μπόρεσε να είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Να πω πολύ σύντομα ότι στηρίζουμε τους συμβιβασμούς 2α και 2β και ζητάμε περισσότερη παρακολούθηση της ασφάλειας. Επίσης ζητούμε ε, περισσότερη πληροφορία. Επίσης στηρίζουμε τους συμβιβασμούς 4α και 4β γιατί θέλουμε να συμπεριληφθεί η περιβαλλοντική διάσταση στο ισοζύγιο ρίσκου ε, ωφέλειας. Γι' αυτό και μας ε, ξαφνιάζει που άλλες πολιτικές ομάδες και κυρίως το EPP θέλουν ε, το 4α ως προήμιο αλλά όχι το 4β που είναι άρθρο. Αυτά και επιφυλασσόμαστε. Je ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολλά υπόθηκαν. Και από την κυρία Ιούσο ιδιαίτερος, τη σκιώδης ηγήτρια. Σε δύο-τρία σημεία μόνο θα αναφερθώ. Δεν ε, επανεφευρίσκουμε το σύστημα της φαρμακοεπαγρύπνησης. Προσπαθούμε μόνο να απλουστεύσουμε το σύστημα αυτό και να έχουμε κάποια στοιχεία που θα μας επιτρέπουν, ε, κάποιο μηχανισμό που θα μας επιτρέπει να καταγράφουμε τις παρενέργειες ε, και ενδεχομένω να συνιστούμε και τις σχετικές στατιστικές. Αυτά. Εγώ είμαι ικανοποιημένη. Πολλές από τις προτάσεις μου και σε συνεργασία με μερικούς συναδέλφους επίσης έχουν κατευθεί, έγιναν δεκτές από τις συμβαστικές τροπολογίες, το εντατική επιτήρηση της surveillance intensive που είχαμε στα γαλλικά τουλάχιστον ε, αφαιρείται για ορισμένα φάρμακα, ε, εντατική παρακολούθηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε πανικό τον ασθενή. Γιατί βέβαια η φαρμακοεπαγρύπνηση δεν έχει λόγο να προκαλέσει πανικό στους ασθενείς, πρέπει μόνο να τους ευαισθητοποιεί, να τους ε, σπρώχνει σε επαγρύπνηση συγκεκριμένα έτσι ώστε να έχουμε τις πληροφορίες για τον ενδεχόμενο κίνδυνο. Το φάρμακο στόχο έχει να θεραπεύει, όχι να προξενεί επιπλέον προβλήματα στην υγεία του ασθενούς. Για την προστασία του περιβάλλοντος και τη σχετική αναφορά. Βεβαίως, όλοι σωστά επισημαίνουν ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό ωστόσο δεν αποτελεί αντικείμενο της φαρμακοεπαγρύπνησης. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να ενταχθεί σε αυτό εδώ το κείμενο. Γι' αυτό θεωρώ ότι αρκεί η αιτιολογική σκέψη. Από την άλλη βεβαίως θα πρέπει να στραφούμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τη ζητήσουμε να αναλάβει, να μελετήσει το θέμα αυτό συγκεκριμένα και να μας κάνει προτάσεις. Τίποτε άλλο δεν έχω να προσθέσω. Με έχουν καλύψει οι συνάδελφοι. Σημειώνω μόνο ότι χαίρομαι που λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των λεγόμενων οφαρμών, ορφανών φαρμάκων, αυτών δηλαδή που ε, στόχο έχουν να θεραπεύσουν τις σπάνιες ασθένειες. Ευχαριστώ κύριε Ροτ Ευχαριστώ πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις και μετά θα μιλήσω για τις τροπολογίες. Η πρώτη παρατήρηση έχει να κάνει με το περιβάλλον. Στην νομοθεσία τη σχετική με τα φάρμακα, ανέξαρτος ε, τύπου, πάντοτε προσπαθούσαμε να εισαγάγουμε τη διάσταση του περιβάλλοντος. Χωρίς ίσως να είναι απαραίτητα ο ιδεοδέστερος των χώρων αυτός εδώ της Επιτροπής μας, θεωρώ ότι θα πρέπει να συζητήσουμε και τη διάσταση του περιβάλλοντος και νομίζω ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και την ε, υπηρεσία φαρμάκων στο στόχο αυτόν. Η κυρία Παπάραβα είπε τι να το κάνουμε αυτό και πώς θα γίνει, θα απαγορεύσουμε τα φάρμακα για το ε, Alzheimer, γιατί είναι επικίνδυνα. Όχι, όμως η ίδια η συνάδελφος ανέφερε τις ορμόνες ή κάποιοι άλλοι μίλησαν για αντιβιωτικά. Ξέρουμε ότι υπάρχουν τέτοια ειζήματα, τέτοια αποθέματα ε, ορμονών και αντιβιωτικών μέσα στα ύδατά μας που δεν είναι παρά τις σημαντικές επενδύσεις δυνατόν να καθαριστούν. Και αν ε, πούμε ότι παρετούμαστε από αυτό στόχο του, ε, της απαλλαγής του περιβάλλοντος από αυτές τις ουσίες, ας ξεχάσουμε οποιαδήποτε έννοια προστασίας του περιβάλλοντος. Ναι, δεν μπορεί να μην υπάρχει πανάκια, αλλά ας αναγνωρίσουμε τουλάχιστον το πρόβλημα. Καθήκον μας είναι ως πολιτικών. Και γι' αυτό πιστεύω ότι 4α και 4β συμβαστικές τροπολογίες θα πρέπει να εγκριθούν με την ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία. Για το ε, φυλάδιο, το ενημερωτικό που ανέφερε και ο κύριος Λίσλ νωρίτερα. Διάβασα τις συμβαστικές τροπολογίες που αναφέρονται σε αυτό ναι, ευχαριστημένοι δεν είμαστε. Ούτε με να με ικανοποιεί μια διατύπωση που λέει ότι θα πρέπει σε 18 μήνε να έχει αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί ξέρουμε ότι η Επιτροπή στέλνει τα πόδια τη στην υπόθεση αυτή και η νομική υπηρεσία, ο κύριο Χέρμπεργκερ και οι συνάδελφοί του που κάθονται εκεί μα λένε ναι, ναι, ναι, βεβαίω θα το κάνουμε κτλ. Η νομική υπηρεσία του, του Κοινοβουλίου. Αλλά η, Ευρω... νομική υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σέρει τα πόδια της, μας λέει, κοιτάξτε τη δική μας, το δικαίωμα της το έχουμε εμείς λοιπά αλλά ένα μήνυμα σας αποστείλουμε, εν πάση περιπτώσει. Και φαντάζομαι ότι η συγκίτρια θα με ρημνήσει και με άλλους τρόπους, με άλλα μέτρα να ε, προωθεί στο θέμα αυτό, εφόσον δεν το αναλάβει εθελοντικά η Επιτροπή. Και επίσης θα ήθελα να επισημάνω τώρα ακόμα δύο σημεία, ναι και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δικές μου τροπολογίες συγκεκριμένα, οι οποίε ενδεχομένω να μην ήταν σαφεί ε, εκ πρώτη όψου για του συναδέλφου, θα ήθελα να σα εξηγήσω. Οι 72 και 77 καταρχάς για τη σύσταση της ε, Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης, Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Φαρμακοεπαγρύπνηση. Προτείνουμε λοιπόν, προτείνεται τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα για αποστολή ενός εκπροσώπου τους στην λόγω επιτροπή. Έτσι προτείνεται αρχικά. Εδώ για μένα είναι όπως θα λέγαμε στο χωριό μου να βάλουμε τον λύκο να φυλάει τα, τα πρόβατα. Ε, δεν ξέρω πώς θα το μεταφράσετε σε άλλες γλώσσες, αλλά πιστεύω ότι οι θα τα καταφέρουν είναι δηλαδή εκείνοι οι οποίοι επί χρόνια συνεχόμενα απέτρεψαν την ανάπτυξη της έννοιας της φάρμακοεπαγρύπησης γιατί δεν έφταγε η Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και με την αμέλειά τους και με, την, ε, με τις αδυναμίες τους, τις ε, πρακτικές, δεν μπορούσαν να διαμορφώσουν τις κατάλληλες δομές δηλαδή, καλούνται τώρα να ε, εξασφαλίσουν με την αποστολή εκπροσώπων του την απρόσκοπτη λειτουργία μιας τη συμβουλευτική Επιτροπής. Όχι κυρίε και κύριοι. Όχι. Ούτω ή άλλως παντού υπάρχει εκπροσώπηση ε, αντιπροσωπευτική και αναλογική όλων των κρατών μελών. Ούτε φτάνισμα δεν επιτρέπεται χωρί να υπάρχει ε, ικανοποιητική εκπροσώπηση των κρατών μελών. Εν πάση περιπτώσει, προχωρήσουμε και χωρί να έχουμε αυτή την εκπροσώπηση. Και γιατί να πληρώνουμε στη τελευταία ανάλυση και τα ταξίδια του ενό και του άλλου. Γι' αυτό παρακαλώ, για να έχουμε και τη δυνατότητα, και προσπάθησα και με τη συμβαστική τροπολογία στην 77 τη δική μου να προσφέρω μια λύση, δηλαδή να μπορούν να συμμετέχουν χωρίς όμως το δικαίωμα της ψήφου, παρακαλώ να με βοηθήσετε κι εσείς να γίνουν δεκτές αυτές οι τροπολογίες και να δούμε τι μπορεί να γίνει στο Συμβούλιο. Γιατί ξέρουμε τι θα γίνει στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο θα πει, Α, όχι εμείς θέλουμε όχι έναν, ε, αλλά τρεις εκπροσώπους για το κάθε κράτο μέλο. Και να περάσω τώρα στην 77. Έχω αλλάξει λίγο τη διατύπωση από το Executive Director σε Executive Director General. Ξέρω ότι είναι αμφιλεγόμενο το ζήτημα. είναι ένα θέμα στο οποίο και κάποιοι συνάδελφοι δεν ξέρουν πώς να τοποθετηθούν επακριβώς. Και ξέρω ότι δεν ε, με ακολουθεί σε αυτό και δεν είναι σύμφωνη μαζί μου 100% ούτε η Επιτροπή, ούτε η Επίτροπη, ούτε το λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε συζητήσει το θέμα και των ε, προκήρυξεων για τι υπηρεσίε ε, τη Ευρωπαϊκής Ένωση στο παρελθόν. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, είχαμε τελείω διαφορετικέ λύσει και σύνθεση προσωπικού. 60 φερρυπίν ε, μέλη προσωπικού και θέση γενικού διευθυντού ως προϊσταμένου τους σε κάποια περίπτωση. Αλλού έχουμε μόνο head of unit, δηλαδή τμήματάρχη, που έχει ε, υπό τις εντολές του περισσότερους ε, υπαλλήλους από ότι ολοκληρή επιτροπή, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Ενώ τώρα μιλούμε για ένα executive director εκεί που θα είχαμε μόνο έναν απλό διευθυντή. Γιατί λοιπόν να, φτάσουμε σε αυτά τα άκρα. Ναι, ξέρω ότι υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με, το, με τα διοικητικά και ποιο θα είναι ο γενικό διευθυντή. Μάλλον το ότι θα πρέπει να υπάρχει γενικό διευθυντή ο οποίο θα διοικεί, θα έχει υπό τι εντολέ του ένα διοικητικό συμβούλιο, ένα management board. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, άλλο είναι να έχει κανεί 600 υφισταμένου και άλλο να έχει 60. Και πρέπει να έχουμε μια κάποια λογική σε αυτή την κατανομή και των υψηλών θέσεων. Και σοβαρότητα, γιατί βεβαίω θα δούμε ποιος έχει ήδη υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση του Γενικού ε, Διευθυντού. Θα εκπλαγείτε γιατί θα δείτε ότι δεν είναι ο καλύτερος υποψήφιος ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι οι καλύτεροι υποψήφοι αυτοί που έχουν καταθέσει υποψηφιότητες τους για τις υψηλές αυτές θέσεις. βλέπουμε να υπάρχουν γενικοί διευθυντέ οι, οποίες, οι οποίοι έχουν το 1 τρίτο του, του προσωπικού από αυτό που έχει ένα απλό διευθυντή σε μια απλή διεύθυνση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α τα δούμε λοιπόν τα πράγματα προ τη σοβαρότητα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα επιμείνω, στο οποίο θα επιμείνω εγώ, όχι γιατί δεν έχω, δεν θέλω κάποιο να έχει υψηλότερο βαθμό και, να, ε, και υψηλότερο μισθό φυσικά, αλλά θέλω οι ευθύνε που θα αναλαμβάνει να έχουν και την κατάλληλη αμοιβή, τον κατάλληλο μισθό δηλαδή, αλλά ταυτόχρονα και να έχουν και την καλύτερη δομή για το προσωπικό που θα δουλεύει σε αυτήν την υπηρεσία. Και αν θέλετε να έχουμε τη σχετική υποπτία, ε, κυρίε και κύριοι, θέλω να σα δείξω, μπορώ να σα προσφέρω μια ε, επισκόπηση των επιχειρήσεων και της, ε, των υπηρεσιών και τη υπηρεσία για τα χημικά, που ξέρετε, το ξέρω, ναι, αλλά υπήρξε ειδική ρύθμιση και με κανονισμό και το υπεστήριξαν έκαθεν. Υπήρξαν όμω και άλλες υπηρεσίε που διαρωτώ με τι κάνουν, πώς περνάνε τη μέρα του αυτοί οι άνθρωποι. Τι κάνουν όλη μέρα. Και ο Executive Director τι κάνει. Με α15, α16 βαθμό. α αλλάξουμε πια αυτή την τακτική. Και γι' αυτό παρακαλώ την 70, λέει η κυρία Ρότσπεραντ, τροπολογία μου να την ε, εγκρίνετε. Euh, euh, Ευχαριστώ κυρία Ροτ Μπέρεντ, ο κύριο Παγνιού. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, και πάλι συγχαρητήρια, Λίντα, πολύ καλή δουλειά. Και πέραν της δουλειάς αυτής ε, συγχαρητήρια και για όλους τους σκιώδους συγητές που κύριο μέλημα είχαν να βελτιώσουν το κείμενο της προτινόμενης οδηγίας γιατί όλοι ξέρουμε την ώρα που κατατέθηκε και η οδηγία και ο κανονισμός, πολλοί έλεγαν ότι θα υποβαθμιστεί η φαρμακοεπαγρύπνηση στην Ευρώπη με τις νέες αυτές προτάσεις. Όμως οι τροπολογίες, οι συμβαστικές τροπολογίες βλέπουμε ότι εξισορροπούν και πάλι το νομικό πλέγμα. Πλην όμως σημειώνω ότι το κείμενο αυτό, το νομοθέτημα αυτό δεν είναι παρά ένα βήμα, ένα ακόμα στάδιο στον αγώνα που, ε, στον οποίο έχουμε αποδηθεί για περισσότερη φαρμακοεπαγρύπνηση και για περισσότερη προστασία του Ευρωπαίου πολίτη. Και θα ήθελα να επισημάνω ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να εγγύψουμε πιστεύω στα επόμενα χρόνια, δηλαδή την αντιπαράθεση, τη διελκυστίνδα περισσότερο μεταξύ της πολιτικής εξουσίας και της φαρμακοβιομηχανίας. Δεν έχει φτάσει στο βαθμό που θα έπρεπε στην ανάλυση της κατάστασης αυτή η οδηγία. Καταλαβαίνω βεβαίως ότι χρειαζόντουσαν και οι συμβασμοί, αλλά πρέπει να καταγράψουμε ότι είναι αδύναμη πολλές φορές η πολιτική εξουσία. Και πολλές φορές ε, στο ζήτημα της φαρμακοεπαγρύπνησης προσφέρουμε υπηρεσία ουσιαστικά στις, ε, ε, στα εργαστήρια των, της φαρμακοβιομηχανίας με, την, ε, με τις διατάξεις για την φαρμακοεπαγρύπνηση. Και όταν βλέπουμε ότι και τη συλλογή και την ανάλυση και την ερμηνεία των δεδομένων την έχουν σε απόλυτο ουσιαστικό έλεγχο οι φαρμακοβιομηχανίες, δηλαδή τους προσφέρουμε με το σύστημα αυτό οι υπηρεσίες, θα πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε με την εξουσία που έχει η πολιτική ε, εξουσία να τους ελέγξουμε και να περιορίσουμε αυτήν την χειραγώγηση των δεδομένων. Θα ε, έφερνα ως ένα μικρό παράδειγμα και υπενθύμηση τα όσα έλαβαν χώρα με την γρήπη H1N1, την γρήπη των χείρων δηλαδή το τελευταίο καιρό. Η κυρία Μακάβαν έχει το λόγο, με όλα αυτά τα εγκόμια ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους σκιώδεις οπωσδήποτε, το προσωπικό, τους βοηθούς που εργάστηκαν πάρα πολύ σκληρά και τη γραμματεία της ομάδας μας. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, νομίζω πως συμφωνούμε για το θέμα του περιβάλλοντος. Τώρα βεβαίως το πρόβλημα είναι πως ε, και από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοι εδώ που είναι 15 χρόνια όλο μιλάμε και τίποτα δεν κάνουμε. Ο, έφυγε και ο κύριος Λίζε. Κάποιες ε, τροπολογίες του ζητούσαν να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα η Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης. Ε, δεν είναι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ειδικοί στην ανθρώπινη υγεία. Τώρα ζητάμε πράγματι να το κάνει η Υπηρεσία Περιβάλλοντος και αυτό είναι το σωστό για αυτά τα οποία λέει ο Πίτερ Λίζα άμεση αναφορά των ασθενών. Ξέρω πως κάποιοι ε, είναι επιφυλακτικοί, αλλά λειτουργεί όπου γίνεται και δεν έχει καταρρεύσει το σύστημα και σύμφωνα με ανεξάρτητες αξιολογήσεις υπάρχουν άμεσα αποτελέσματα καθώς οι ασθενείς αναφέρουν άμεσα τις παρενέργειες για τις παρεκκλήσεις. Ε, για τις αναφορές ε, ομοιοπαθητικών φαρμάκων 2.46 και 2.47 εάν έχουν τα ομοιοπαθητικά φάρμακα δραστική ουσία πρέπει να ε, υπόκειται σε φαρμακοεπαγρύπνηση. Νομίζω πως αυτό καλύπτει τα περισσότερα ζητήματα και ελπίζω να ψηφίσουμε αύριο το πρωί αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. πολύ. Αύριο θα ψηφίσουμε το πρωί. Ψηφοφορία τον Ιούνιο στην Ολομέλεια. Και τελευταίο σημείο για την σημερινή μας ημερησία διάταξη. Μια και δεν είναι εδώ η κυρία Βέστλουντ, θα παρακαλέσω τον κύριο Γιώργενσεν αν θέλει να κάνει την παρουσίαση της εκθέσεως. Ευχαριστώ πολύ. Μιλώ εκ μέρους της κυρίας Βέστλουντ που δεν μπορεί να είναι εδώ. Το ψήφισμα αυτό θέλει να αποφύγει τη συμπερίληψη της τρομβίνης στο παράρτημα 4 της οδηγίας 95.2. Ίσως όμως ε, εισαγωγικά θα μπορούσα να σας δώσω λίγο το ιστορικό του, τι ακριβώς ε, είναι η ουσία αυτή. Μιλάμε για ένα ένζυμο, το οποίο προκύπτει από το αίμα χείρων ή βοηδών και είναι ένα ένζυμο το οποίο είναι φυσικό συστατικό του αίματος ε, των θηλαστικών και θεωρείται ο τελικός ε, σύνδεσμος σε αυτό που θα μπορούσε να αποκαλέσει κάποιος τη διαδικασία πήξης του, αίμα, αίματος. Ε, με λίγα λόγια είναι το ένζυμο το οποίο επιτρέπει στο αίμα να πίζει και αυτό σας δημιουργεί και τις σουλές ε, στις πληγές. Πρόκειται λοιπόν για μια φυσική ουσία. Ε, τι ακριβώς ε, θέλει να κάνει με την ουσία αυτή η βιομηχανία τροφίμων. Θέλει να συγκολά τμήματα κρέατος ε, μεταξύ τους ώστε να έχουμε ένα ενιαίο τμήμα και γι' αυτό θεωρείται ότι είναι κόλλα κρεάτων. Αυτή καθε αυτή η ουσία δεν είναι επικίνδυνη. Από τις μελέτες που έχουν γίνει αυτό το αποτέλεσμα έχει προκύψει και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να επιτρέψει τη χρήση αυτής της ουσίας. Δεν είναι επικίνδυνη αν την εξετάσουμε μεμονωμένα. Το πρόβλημα είναι η χρήση της ουσίας αυτής, η οποία μπορεί να έχει κάποιες πολύ ε, επιζήμιες συνέπειες και γι' αυτό και εμείς θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Να σας δώσω τρία επιχειρήματα κατά της χρήση της ουσίας αυτής. Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι παρά το γεγονός ότι αυτή η ουσία δεν είναι επιζήμια για την υγεία, μπορεί να έχει κάποιες ε, επιπτώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να είναι επιζήμιες για την υγεία. Όπως ε, ίσως πολλοί από σας γνωρίζουν, ένας από τους κινδύνους ε, χρήστης ε, κρέατος είναι ότι μπορεί να υπάρξουν βακτήρια και πολλά βακτήρια βρίσκονται στην επιφάνεια του κρέατος. Όσο μεγαλύτερη λοιπόν η επιφάνεια του κρέατος, τόσο μεγαλύτερος κίνδυνος ελοχεύει να έχουμε βακτηρίδια ε, στο κρέας, όπως για παράδειγμα η σαλμονέλα, που όλοι γνωρίζουμε πόσο σοβαρός κίνδυνος ε, ε, είναι. Αν όμως αντί να έχουμε ένα ενιαίο κομμάτι κρέατος, έχουμε πολλά διαφορετικά τμήματα κρέατος τα οποία συγκολούνται μεταξύ τους, καταλαβαίνετε ότι ο κίνδυνος αυτός μεγαλώνει. Επίσης, μπορεί να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση όπου θα παραπληροφορούμε και θα παραπλωνούμε τους καταναλωτές. Το γεγονός ότι κάποιος πουλά ένα κομμάτι κρέατος το οποίο παρουσιάζεται ως ενιαίο ενώ στην πράξη αποτελείται από διαφορετικά τμήματα και αυτό δεν είναι σαφές προς τον καταναλωτή σημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη διαφάνειας. Και αυτό ίσως θα μπορούσαμε να το επιλύσουμε μέσω της κατάλληλης ετικέτας, αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον καταναλωτή να γνωρίζει ότι αυτό που του φαίνεται ως ένα νέο κομμάτι κρέας είναι ε, ένα αμάλγαμα πολλών τμήματων κρέατος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπεται, για παράδειγμα, να σερβίρεται στα εστιατόρια αυτό. Εδώ προκύπτει και το πρόβλημα. Αν δεν επιτρέπεται να σερβίρεται στα εστιατόρια, γιατί θα πρέπει να, σε, να επιτρέπεται η χρήση του οπουδήποτε αλλού. Και ένα τελευταίο επιχείρημα το οποίο θα ήθελα να σα παρουσιάσω είναι το εξή. Εξ όσων διαπιστώνω εγώ, δεν υπάρχει κάποιο εύλογο επιχείρημα για να επιτραπεί η χρήση αυτής της ουσίας. Δεν υπάρχει κάποιο προστιθέμενο όφελος. Ε, δεν μπορούμε να πούμε πουθενά ότι ορίστε υπάρχουν αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις αλλά κοιτάξτε και, κοίτα, και κάποιες καταπληκτικές ε, ευεργετικές δράσεις που έχει. Και εγώ ποτέ δεν άκουσα κάποιο καταναλωτή να λέει ότι ε, θέλω ένα κρέας κολλημένο σε κομματάκια. Μας προσεγγίζουν πολλοί καταναλωτές και κανένα δεν μα είπε ότι είναι φρικτό ότι δεν μπορούμε να αγοράσουμε τέτοιο κρέα στο σούπερ μάρκετ. Ε, θα ήταν καταπληκτικό να έχουμε την ευκαιρία να αγοράσουμε ένα κομμάτι κρέα που θα αποτελείται από πολλά κομμάτια κρέατος κολλημένα μεταξύ του. Δεν φαντάζομαι δηλαδή ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση για αυτό το προϊόν. Υπάρχει όμως μια ομάδα ανθρώπων που το θέλει και είναι η ομάδα των ανθρώπων που θέλει να εξοικονομήσει χρήματα πολλώντας αυτό το προϊόν και μάλιστα θεωρούν ότι ο καταναλωτής ε, θα ε, το δεχτεί αυτό. Πολλές οργανώσεις καταναλωτών ήταν επικριτικές σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Σουηδία και στη Γερμανία σίγουρα. Το θέμα συζητήθηκε ιδιαίτερα στα μέσα ενημέρωσης και αποτελεί και πολύ καλό παράδειγμα του πώς ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ε, μπορεί να προσπαθεί να ε, βοηθήσει τους παραγωγούς να βγάλουν χρήματα εις βάρος των καταναλωτών. Νομίζω ότι η κατάσταση θα πρέπει να σταματήσει εδώ και ελπίζω να υποστηρίξετε και εσείς το ψήφισμα. Συνοψίζοντας, μιλάμε για μια ουσία η οποία θα μπορούσε να είναι παραπλανητική για τους καταναλωτές, έχει δυνητικά πολύ σοβαρές επιπτώσεις λόγω της ανάπτυξης βακτηριδίων, δεν υπάρχει κανένα όφελος το οποίο είναι γνωστό ε, και θεωρώ ότι στο μέτρο του δυνατού θα πρέπει να την αποφύγουμε. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει και αυτή η δυνατότητα να απορρίψουμε την έγκριση αυτής της ουσία. Euh, Εγώ προσωπικώς και έχουμε να ομάδας μου συμμερίζουμε απόλυτος απόψεις. Κυρία Αγίουσο, έχετε εσείς το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ήμουν σκιώδης εισηγήτρια για τα πρόσθετα Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να παρέμβω. Πράγματι, η οδηγία 95.2 επέτρεπε την τροποποίηση των παραρτημάτων και εδώ βρισκόμαστε ενώπιον μιας τέτοιας κατάστασης. Για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί κάποιο πρό, ε, πρόσθετο θα πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις και καταρχάς θα πρέπει να είναι ασφαλές. Η ΕΦΣΑ είπε ότι μελέτησε αυτό το δείγμα και σε γνωμοδότηση της 26 Απριλίου του 2009 είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάλλιστα η ουσία. Επίσης είπε ότι ε, από τεχνικής απόψεως ε, είναι καινοτόμο το προϊόν. όντω πρόκειται για καινοτόμο προϊόν που βοηθά στην αύξηση της σταθερότητα του τελικού προϊόν και από αυτή την πλευρά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει κάποιο όφελος όπως λέει ο κανονισμός για τα πρόσθετα. Επιπλέον ο κανονισμός λέει ότι δεν θα πρέπει να παραπλανά τον καταναλωτή και αυτό είναι το επιχείρημα που χρησιμοποιεί η συντάκτρια του ψηφίσματος. Ναι, ε, είναι λογικό το επιχείρημα, αλλά απαιτείται η ετικετοθεσία. Εάν λοιπόν ένα καταναλωτή θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό το προϊόν, το οποίο δεν είναι επιζήμιο σε καμία περίπτωση, θα πρέπει να είναι ασφαλέ, θα γνωρίζει ότι το χρησιμοποιεί, δεν επιτρέπεται η χρήση του σε εστιατόρια και επομένω δεν υπάρχει παραπλάνηση προ τον καταναλωτή. Το οποίο θεωρώ ότι είναι το μόνο το οποίο θα μπορούσαμε ίσω να χρησιμοποιήσουμε ως αιτιολογία για να ζητήσουμε την μη έγκριση του προϊόντος. Πρόκειται για ε, προϊόντα μεταποιημένα για τα οποία υπάρχει σαφής απέτηση ετικέτας. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι μπορεί να επαναπληρωθεί ο καταναλωτή. Το θέμα αυτό έχει ξανασυζητηθεί στο παρελθόν όταν συζητούσαμε τον κανονισμό για τα πρόσθετα και δεν υπήρχε κάποιο ε, επιχείρημα κατά της χρήσης. Για τους λόγους λοιπόν ε, στους οποίους σας εξέθεσα, κατά την άποψή μου δεν υπάρχει ε, βάση για να υποστηρίξουμε την άποψη της συντάκτριας βάση των όσων υπάρχουν και στην οδηγία. Να μην ξεχνάμε ότι το προϊόν ε, υπόκειται και στη χρήση περίπου άλλων 20 προσθέτων. Υπάρχουν ε, δηλαδή κάποια επιχειρήματα τα οποία ίσως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ε, μία έγκριση του προϊόντος, αλλά κατά την άποψή μου δεν είναι στοιχεία τα οποία στέκονται. Ε, δεν υπάρχει δυνατότητα παραπλάνησης του καταναλωτή διότι υπάρχει σήμανση η οποία θα γράφει ότι ο καταναλωτής αγοράζει ένα προϊόν το οποίο έχει προκύψει με τη χρήση αυτού του πρόσθετου και δεν επιτρέπεται και η χρήση του σε εστιατόριο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχουμε επαρκή βάση για να μπορέσουμε να αρνηθούμε την έγκριση της ουσίας αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ πλήρω με τον εισηγητή. Το μόνο νόημα που έχει αυτό το προϊόν είναι να πουλήσουν πράγματα στον καταναλωτή. Κάτι το οποίο δεν είναι κρέα το κάνουν να μοιάζει με ένα κομμάτι κρέας. Δηλαδή μπορεί να το λέει πουθενά στα ψηλά γράμματα, αλλά όταν το κοιτάει ο καταναλωτής νομίζει ότι είναι ένα κομμάτι κρέας. Εντάξει, η χημική ουσία δεν είναι επικίνδυνη, δηλητηριώδης, αλλά υπάρχει κίνδυνος στην διαδικασία επιμόλυνσης. Και βεβαίως ε, δεν αντέχει και τόσο πολύ. Είναι πιο ευπαθές, οπότε υπάρχει πιθανός βακτηριολογικός ε, κίνδυνος. Οπότε πιο σύντομη η ημερομηνία λήξη. Τόσο νομίζω πως είναι πιλωτική η περίπτωση αυτή. Δεν είναι ε, πραγματικά επικίνδυνο, αλλά πρέπει να σκεφτούμε για μία φορά και το νόημα της νομοθεσίας. Το νόημα της νομοθεσίας περί τροφίμων είναι να μην παραπλανείται ο καταναλωτής και τα πράγματα που εγκρίνουμε υποτίθεται ότι είναι καλά. Και εδώ πέρα δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Οπότε δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να περάσει. Πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Να πούμε δηλαδή ότι ε, μόνο και μόνο επειδή δεν βλάφτει και δεν πεθαίνει κανείς, ε, πρέπει να το εγκρίνουμε. Όχι. Υπάρχουν και ηθικές πτυχές. Κάποια στιγμή πρέπει να υψώσουμε το ανάστημά μας να τηρήσουμε αυτά τα οποία γράφει η συνθήκη και η νομοθεσία. Και εδώ πέρα πρέπει να πούμε πως δεν το θέλει αυτό το πράγμα ο καταναλωτής, υπάρχει κίνδυνο παραπλάνησης και ποιο θα πληρώσει όλου αυτούς τους ελέγχου, Ο καταναλωτή τους ελέγχου για, στα εστιατόρια για το ότι δεν κάνουν κόλπα. Είναι μόνο αρνητική λοιπόν η ολυμπόση και πρέπει να πούμε όχι. κυρία Ροτ Μπέρεντ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Βεβαίω χρησιμοποιείται στα εστιατόρια, στους κοιμάδες και αλλού. κοιτάω τώρα εγώ τους φίλους που παρακολουθούν τη σχετική νομοθεσία εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ νομίζω ότι χρειαζόμαστε άλλο ένα σκάνδαλο. Επί τρελών αγελάδων ούτε στα όνειρά της δεν θα ερχόταν με τέτοιο χαρτί η Κομισιόν. Αντιθέτως, τότε σκεφτόμασταν να απαγορεύσουμε το να γδίνουν το κόκαλο από το κρέας και να, να χρησιμοποιούν αυτό το κρέας. Οπότε, τουλάχιστον ο προκάτοχος του κυρίου, του κυρίου Μπουτιλέ ε, το είχε πει, είναι αειδιαστικό. Και αυτό το οποίο κάνουμε εδώ πέρα επίσης είναι αειδιαστικό. Είναι δύο οι πτυχές. Πρώτα απ' όλα η υγεία. τι γίνεται με την επιφάνεια των κομματιών που τα έχουμε κολλήσει μαζί, που δεν θα ζεσταθούν, που δεν θα μπουν σε κονσέρβα, που δεν μπορούν να καθαριστούν. Γιατί μιλάμε για ελάχιστα κομματάκια. Ε, ας είμαστε ειλικρινεί, πρόκειται περί αποβλήτων. Πρόκειται για κομμάτια που τρώγονται του κρέατος, αλλά τα οποία κανονικά κανείς δεν θα έτρωγε. Αυτό το πράγμα δεν επιτρέπεται να γίνει ζωοτροφή για τον χύψη λόγο. Δεν υπάρχει επιστημονικός λόγος κατά αυτού του πράγματος και εδώ πέρα θέλουμε να επιτρέψουμε αυτά τα ελάχιστα κομματάκια απόβλητα ή μάλλον παραπροϊόντα της παραγωγής να γίνουν ξανά προϊόν. Βεβαίως είναι παραπλανητικό, συγγνώμη δηλαδή και με κάθε σεβασμό στους συναδέλφους της Κομισιόν, και στον κύριο Πουντιλέτορα που είχαν παλέψει μαζί για την ε, ασθένεια των ε, τρελών αγελάδων. Δηλαδή, να πούμε ότι φτάνει να γράψουμε θρομπίνη. Εγώ είμαι και ενημερωμένη καταναλωτή και δεν μου φτάνει αυτό το πράγμα. Όχι. Ή να μπει δίπλα στο, στον τόπο προέλευσης συνδυασμένα μέρη κρέατος. Ε, δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει και αν τα έχετε πάρει χαμπάρι στην Κομισιόν τι γίνεται στα κρατη με το συνθετικό τυρί στην, ε, στις πίτσες. Όταν ξεκινάει ένα σκάνδαλο στην ε, Ισπανία και μετά καταραίει η αγορά με τα, με τα μούρα εκεί πέρα γιατί βρέστηκαν κάποια εντομοκτώνα θα, θα καταρρεύσει η αγορά και δεν υπάρχει εδώ πέρα καμία δικαιολογία ούτε χρειάζεται Ούτε μπορούμε να το εξηγήσουμε δηλαδή στον, στον καταναλωτή. Τι πάνε να πει συνδυασμένα α, προϊόντα. Όποιο θέλει να το κάνει, δηλαδή να κάνει ένα ζαμπ, όχι. Αυτό το, το προϊόν κατ' ουσίαν το κάνει, τα ανακατεύει με ζελατίνη και το κάνει. Αλλά πέρα από την ουσία, το πρόβλημά μου είναι πως σιγά σιγά επισέρχεται πάλι μία τάση να είμαστε έτσι λίγο πιο χαλαροί. Και ανησυχώ, ανησυχώ πραγματικά. Και ελπίζω να μην είναι τακτική της ε, Κομισιόν, γιατί έχουμε τώρα νέους βουλευτές που δεν ήταν εδώ πριν από 12 χρόνια όταν είχαμε τη μεγαλύτερη κρίση τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω πραγματικά ναι, να έχετε καταλαβεί ότι δεν είναι ο θέμα ο κίνδυνος ο υγειονομικός, είναι και η αντίληψη του καταναλωτή, τι βλέπει, τι, τι νιώθει ο καταναλωτής. Πρέπει εγώ να πάω να πω στους εκλογείς μου και θα μου πούν αυτοί οι άνθρωποι είχαμε το τεχνητό τυρί στην πίτσα και τώρα το κρέας δεν είναι κρέας και το χειρομέρι δεν είναι χειρομέρι. Όχι δεν, μπορώ εγώ να τα πω αυτά τα πράγματα. Το ψήφισμα είναι καλό, πρέπει να το δεχτούμε. Το προϊόν αυτό δεν επιτρέπεται να μπει στο παράρτημα και δεν επιτρέπεται και η ουσία αυτή να κυκλοφορήσει. Ευχαριστώ. Συμφωνώ πολύ με το όσο είπε η Ντάγμαρ. Κάλυψατε περισσότερα πράγματα και τις θα είμαι σύντομη. Το πρόβλημα είναι ότι δεν αγοράζει κανένα κομμάτι κρέας. Πια. Εάν πούμε βέβαια στον καταναλωτή ότι αυτό που πάει και αγοράζει το πακέτο είναι ε, πολλά μικρά κομματάκια τυριού, τα οποία έχουν, ε, κρέατος τα οποία έχουν κολλήσει μαζί με μια ουσία, μάλλον δεν θα ψώνιζε. Άρα είναι θέμα ενημέρωσης περισσότερο. Και υπάρχει, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, κίνδυνος μόλυνσης και επιμόλυνσης, πράγμα το οποίο βρίσκω πολύ πιο επικίνδυνο από το να παρα... Ε, να δίνονται να παραπληροφορείται ο καταναλωτής, που είναι ούτως ή άλλως πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε μια υπεύθυνη στάση στην υπόθεση αυτή και γι' αυτό δεν πρόκειται να υποστηρίξω την ε, ε, διάθεση στην αγορά τέτοιου είδου ε, προϊόντων. Θα υποστηρίξω λοιπόν το ψήφισμα. Πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτή τι τρώει, τι περιέχουν τα τρόφιμα που αγοράζει. Σα ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Και εγώ προσωπικώ συμμερίζομαι πλήρω τα όσα είπε η Ντάκμαρ, Ροτ Δεν βλέπω Πώς είναι δυνατόν να ισχυρίζεται κανείς ότι προσπέσετε τα δικαιώματα του καταναλωτή, ότι θέλει καθαρά τρόφιμα στην ευρωπαϊκή αγορά και επιτρέπει κάτι τέτοιο. Ο κύριος ε, που το κύριος Διευθυντής, έχετε την καλοσύνη να υπερασπιστείτε αυτές τις θέσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βαρύ έργο, αλλά σημαντικό. Ως προς την υγεία, καταρχάς, και τον κίνδυνο για την δημοσιογεία το ότι Το ανέφερε και ο κύριος Γιώργινσεν, είναι ένα, πολύ, ένα φυσικό προϊόν. Το βρίσκεται και στο αίμα των ζώων και στο αίμα του ανθρώπου. Διαγράμμισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος προς τον, ε, για τον καταναλωτή ω προ τη χρήση αυτού του προϊόντος. Ο κίνδυνο όμω από την ε, ανάμειξη διαφόρων τμήματων κρέατος μέσα στο ίδιο προϊόν και την ενίσχυση τη επιμόλυνσης λόγω τη αλμονέλας φυσικά είναι υπαρκτό. Ωστόσο είναι καθήκον τη βιομηχανία να μετριάσει τον ε, κίνδυνο αυτόν. Πρόκειται για ένα προϊόν με περισσότερους κινδύνους από το καθαρό κρέας, το φυσικό, αν θέλετε, μη ανασυσταθέν κρέας. Το ίδιο όμω, τον ίδιο κίνδυνο ενέχει και ο κοιμά ή τον αυξημένο κίνδυνο, να το πω διαφορετικά. Και πάλι πρέπει η βιομηχανία να ε, περιορίσει τον κίνδυνο, να τον ελέγξει και αν αποδειχθεί ότι δεν τα κατάφερε, έχει και τις σχετικές ευθύνες. Καθήκον όμως του κλάδου είναι να ε, προσέξει όταν ε, γίνεται επανασύσταση διαφόρων ε, τμήματων κρέατος να ελέγχει ιδιαίτερος ώστε στα φιλόκοκοι σαλμονέλες ή ληστερία να μην, πέφτουν, να μην μπαίνουν στην αγορά μέσω αυτών των ανασταθέντων τμήματων. Ξέρετε ότι στην οδηγία προβλέπεται μέσα στα κριτήρια για την έγκριση ενός πρόσθετου τροφίμων, να υπάρχει μια λογική ανάγκη, να ικανοποιείται μια λογική ανάγκη. Ό,τι σημαίνει αυτό έτσι. Αυτή η θρομβίνη λοιπόν που έχει σαν ε, λειτουργία την επανασύσταση του κρέατος έχει και σταθεροποιητική λειτουργία γιατί επιτρέπει να, ε, να συνδεθούν μεταξύ τους οι πρωτεΐνες έτσι αυτό το κρέας, το επανασυσταθέν, κρατάει περισσότερο και μάλιστα κρατάει και περισσότερο από ότι το, το γνωστό παραδοσιακό, λέει ο μιλητής, κρέας. και ως εκ τούτου προσφέρουν το εξή πλεονέκτημα, άσχετα αν υποστηρίζει κανείς ή όχι τη λύση αυτή, ότι μπορεί, επιτρέπει δηλαδή να προσφερθεί ένα κρέας, ναι, λιγότερο καλής ποιότητας, αλλά ε, διατροφικής, αλλά πάντως υγειονομικής ποιότητας ικανοποιητικής, σε τιμή πολύ χαμηλότερη από αυτήν του απλού κρέατος, λέει ο μιλήτης. Το επανασυσταθέν κρέας, ε, υψητό, είναι δεδομένο, είναι γεγονός. Υπάρχουν διάφορες ουσίες πρόσθετες, αλγινάτες, πολυφωσφορικές κτλ. που έχουν λάβει τη σχετική άδεια και κυκλοφορούν, χρησιμοποιούνται. Ή φεριπίν εμείς χρησιμοποιούμε στην ε, κουζίνα, κάθε ένα ε, στην μαγειρική του το ασπράδι, τον κρόκο του αυγού ή και πλάσμα ακόμη. Ναι κυρία Κρουστέτ, σας διαβεβαιώνω. Δεν ξέρω εσείς τι είδου ε, μαγειρική κάνετε, εν πάση περιπτώσει πατέ δεν κάνετε, το πατέ που αναμειγνύεται διάφορα κρέατα ή και λαχανικά και χρησιμοποιείτε το, το ασπράδι του αφού για να δέσουν όλα αυτά μαζί τους. Όχι με θρομβίνη, αλλά στην καθημερινή μας μαγειρική, ο καθένας στην κουζίνα του, είμαι σίγουρος ότι χρησιμοποιούμε αντίστοιχες μεθόδους. Επίσης, η τιμή και η σημασία για τον καταναλωτή. Είναι η πρώτη φορά που η νομοθεσία μας ενσωματώνει μια σειρά ε, δεδομένων για να αποφευχθεί η εξαπάτηση του καταναλωτή. Δηλαδή ούτε στο catering, ούτε στα εστιατόρια, ούτε στα ευρεία κατανάλωση τρόφιμα ε, μπορεί να υπάρξει αυτή η θρομβίνη. Μόνο στα προσυσκευαστικά τα προϊόντα, αυτά που αγοράζει κανεί στο σούπερ μάρκετ και μπορεί να είναι πιο φτηνά για τον καταναλωτή. Δεύτερον, και θα υπάρχει σχετική σήμανση, επισήμανση, το είπατε κι εσείς. Ανασυσταθέν κρέας. Μικρά γράμματα, μεγάλα γράμματα, μπορούμε να το διευκρινίσουμε στο μέλλον. Πάντως, δίπλα στον ε, τίτλο του προϊόντος ε, θα πρέπει να υπάρχει η σχετική επισήμανση έτσι ώστε να μην νομίζει κανείς ότι αγοράζει ένα μπούτι ψητό ή ένα, ένα κομμάτι νουά ας πούμε για ψητό καθαρό αλλά ότι είναι ένα νουά ανασυσταθέν. Και η ζωική προέλευση της τρομβίνης. Είτε πρόκειται για το βόδι, είτε πρόκειται για τον χείρο, γιατί βέβαια για λόγους θρησκευτικού ξέρετε ότι υπάρχουν ζητήματα και για λόγου, για, συστατικά δηλαδή υπάρχουν κάποιες πρωτεΐνες που χρησιμοποιούνται χωρίς να είναι πρόσθετα, των οποίων όμως δεν γνωρίζουμε την ζωική προέλευση. Και αυτό είτε ένα μουσουλμάνος, είτε ένα Ινδουιστής, είτε δηλαδή εκείνοι οι οποίοι θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι ιερό ζώο και δεν θέλουν να καταναλώνουν βόλιο κρέα, ε, δεν θέλει να ε, καταναλώσει αυτέ τι ουσίε μέσα στο φαγητό του. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που έχουμε τόσο ξεκάθαρη αναφορά και επιπλέον περισσότερη διαφάνεια, καλύτερη ενημέρωση για τον καταναλωτή, ο οποίο θα μπορεί γνωρίζοντα ε, επακριβώς περί τίνο πρόκειται να διαλέξει το προϊόν που θέλει. Βεβαίω έχουμε πρόβλημα απατών, δυνατότητα απατών από τα εστιατόρια. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Αλλά καθήκον των κρατών μελών θα είναι να επαγρυπνούν για την ομαλή και απρόσκοπτη τήρηση αυτή τη νομοθεσία, Η αγορανομία του, όταν θα, πάνε να όταν θα να ελέγχει τα εστιατόρια αυτά, εάν βλέπει τέτοιου είδου κρέα, θα πρέπει να επιβάλλει σχετικέ κυρώσει. Απλούστατα αυτό είναι το καθήκον των κρατών μελών με την ε, ε, παρακολούθηση τη ορθής εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Είτε λοιπόν πρόκειται για κτηνιατρικές, αγορανομικές, υγειονομικές υπηρεσίες, όταν επιθεωρούν αυτά τα εστιατόρια και κυρίως τα, τις αλυσίδες μαζικής παραγωγής, θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να μην χρησιμοποιούνται εκεί αυτά τα φέντα κρέατα. Και το κείμενο, εάν επιτρέψετε βέβαια την ε, έγκρισή του, ακριβώς σε αυτό θα δώσει έμφαση και η Επιτροπή θα επιμείνει, τα κράτη-μέλη, εφόσον υπάρχουν μέτρα τα οποία ε, τελικά σημαίνουν πως μόνο ο ιδιώτης καταναλωτής θα μπορεί να αγοράζει το και μάλιστα σε, προσ... σε προσυσκευασία το κρέας αυτό, θα έχει πρόσβαση σε αυτό και θα υπάρχει αντίστοιχο έλεγχος ότι θα μπορούν τα εστιατόρια και οι μεγάλες αλυσίδες εστίασης να τα διαθέτουν. Ίσως να μην σας ικανοποιούν οι διατάξεις. Ίσως. Πάντως αντιστοιχούν στα τρία κριτήρια της οδηγίας δεν υπάρχει πρόβλημα υγειονομικό, υγείας, δημόσιας υγείας για τον καταναλωτή. Ικανοποιείται μια τεχνολογική ε, ανάγκη, αν θέλετε, και δεν υπάρχουν άλλες περιπλοκές οικονομικές. Άλλες. Είναι αυτό που μας καλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε φορά να επαληθεύουμε όταν στα κράτη-μέλη και μετά βεβαίως στο Κοινοβούλιο υποβάλλουμε προς ε, τέτοιου είδους κειμένων η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Μας κατατρομάξατε. Αλλά ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Δύο λόγια για τον εισηγητή, αν έχει την καλοσύνη. Είναι περασμένη ώρα όμως. Δεν θα επαναλάβω όλα όσα είπα αρχικά. Να σχολιάσω λίγο αυτό το οποία είπαν οι συνάδελφοι και η Κομισιόν. Να ξεκινήσω από την Κομισιόν. Είπατε πως δεν υπάρχει κίνδυνος ή πως ο κίνδυνος δεν σχετίζεται με την ουσία, το ένζυμο κάθε αυτόν αφορά την χρήση του ενζύμου. Και εσείς το αναγνωρίσατε. Είπατε πως είναι ένας κίνδυνος που πρέπει να ελαχιστοποιήσει ο κλάδος. Ε, δεν επαφίεται μόνο στον κλάδο. Και οι πολιτικοί μπορούν να το κάνουν και οι κομισιόν. Αυτό κάνουμε συνέχεια. Οπότε νομίζω πως αυτό είναι το βασικό επιχείρημα για να κάνουμε αυτό το οποίο προτείνουμε να μην εγκρίνουμε αυτή την ουσία δηλαδή. Επίσης λέει μάλιστα σχετική νομοθεσία περί προσθέτων τροφίμων πως πρέπει η χρήση να έχει πλεονεκτήματα για τον καταναλωτή. Εσείς λέγατε, αντιμετωπίσατε στην ομιλία σας τα προβλήματα που επισημάναμε εμείς. Και δεν αναφέρατε κάποιο πλεονέκτημα. Ίσως να είναι φτηνότερα τα προϊόντα. Πού το ξέρουμε αυτό. Μπορεί. Γιατί θα είναι πολύ κακή ποιότητα κρέατος, αλλά το ξέρουμε αυτό. Μήπως διακινδυνεύουμε το ότι θα προσπαθήσουν απλά να βγάλουν μεγαλύτερο κέρδος. Πώς ξέρετε, έχει γίνει καμία μελέτη που μας λέει πως οι καταναλωτές θα ωφεληθούν. Ίσως, αλλά δεν το ξέρουμε. Είναι τόσο αβεβαίο που ακόμα και αν γίνει